Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, πρέπει να ξεκινήσουμε. Χαίρομαι που οι περισσότεροι συνάδελφοι είναι εδώ. Και κυρίως ο κύριος Χάρμπορ και η Εύλιν Γκέρπχαρτ και ο κύριος Κούρτοβιτς. Και επίσης η Επιτροπή έχει λάβει τις θέσεις της και επομένως μπορούμε να ξεκινήσουμε παρότι πολλοί από τους άλλους συναδέλφους λείπουν. Έχουμε την δημοκρατία της Τσεχίας και έτσι θα περάσω τώρα στα τσέχικα. Σας παρουσιάζω τον Υπουργό Μάρτιν Φρίμαν, Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας. Ήταν επίσης, διατέλεσε επίσης και Υπουργός Μεταφορών. Θα ήθελα επίσης να σας παρουσιάσω τον κύριο Ζάιτσεκ, που εκπροσωπεί την μόνιμη αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας της Τσεχίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι το πρόσωπο επαφής για τα θέματα που έχουν να κάνουν με την Επιτροπή μας. Και την κυρία Κοντομπόλαφ από την μόνιμη αντιπροσωπεία επίσης. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να ξεκινήσουμε με τα εισαγωγικά σχόλια του Υπουργού. Μια όμως και έχουμε μόλις 3,5 μήνες στη διάθεσή μας για να συζητήσουμε όλες τις εκθέσεις μας, πρέπει να θέσουμε ορισμένες προτεραιότητες. Πρέπει να συγκεντρωθούμε στα θέματα εκείνα για τα οποία μπορούν να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Εγώ συζήτησα νωρίτερα σήμερα με τον Υπουργό ε, τι δυνα, και είδαμε τι δυνατότητες έχουμε και πώς μπορούμε να συντονίσουμε τις ε, εργασίες μας για να μπορέσουμε να κλείσουμε κάποια θέματα. Ας δώσω λοιπόν το λόγο τώρα στον Υπουργό. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, βουλευτές, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να αρχίσω λέγοντας ότι θα χαρώ να σας παρουσιάσω σήμερα τις προτεραιότητες της ε, Δημοκρατίας της Τσεχίας πάνω στην εσωτερική αγορά τι. Θα θέλαμε να δώσουμε συνέχεια στο, στο έργο που επιτέλεσαν οι προηγούμενες προεδρίες η συνεργασία μεταξύ Γαλλίας, Σουηδίας και Δημοκρατίας της Τσεχίας υπήρξε πολύ επωφελής μέχρι στιγμής. Καταφέραμε να θέσουμε κάποιες κοινέ προτεραιότητες στο, σε ένα 18μηνο χρονικό πλαίσιο και ακολούθως ορίσαμε τις προτεραιότητες της, τσεχικής, της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Μας ενδιαφέρει η καλή συνεργασία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. έτσι ώστε οι διαπραγματεύσεις ε, στην διαδικασία της συναπόφασης να είναι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικές. Ξέρουμε ότι η θητεία του Κοινοβουλίου φτάνει στο τέλος της και γι' αυτό ο χρόνος που διαθέτουμε για να συζητήσουμε τις διάφορες προτάσεις είναι πολύ περιορισμένος. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί και να κάνουμε σωστή χρήση του χρόνου που μας απομένει. Αυτό είναι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθεί οποιαδήποτε πρόοδος. Η γενική προτεραιότητα της Προεδρίας μας συνοψίζονται στην οικονομία, την ενέργεια, και την Ευρώπη στον κόσμο. Πρόκειται για την πολιτική των τριών «Η» του γράμματος E της αγγλικής αλφαβήτου. Εγώ πιστεύω ότι σε συνεργασία με την Επιτροπή σας και μπορούμε να, να άρουμε πολλά εμπόδια στην συνεργασία μας. Η Δημοκρατία της Τσεχίας ανέλαβε την Προεδρία σε μια δύσκολη περίοδο. Ε, έχουμε το δύσκολο καθήκον εμείς μαζί σας να αντιμετωπίσουμε τα χρηματοπιστωτικά και οικονομικά προβλήματα όχι μόνο των κρατών μελών αλλά ολόκληρου του κόσμου. Τον περασμένο Δεκέμβρη τα κράτη-μέλη συμφώνησαν πάνω σε ένα σχέδιο, ευρωπαϊκό σχέδιο ανάνυψης. Αυτό περιλαμβάνει διάφορα μέτρα. Την ε, επιτάχυνση απελευθέρωσης κονδολίων για τα διαρθρωτικά ταμεία, επίσης η επιτάχυνση και η διευκόλυνση δανεισμού των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω των Ευρωπαϊκών Τραπεζών. Ε, επίσης έχουμε την εφαρμογή της πράξης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ε, οι βραχυπρόθεσμες πολιτικές μας πρέπει να εναρμονίζονται με τις μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες στρατηγικές μας. Και εδώ έχουμε τη δική σας επιτροπή της αρμοδιότητας σα ε, για την προστασία του καταναλωτή και την εσωτερική αγορά πρέπει να άρουμε τα σχετικά εμπόδια και για να το καταφέρουμε αυτό πρέπει να δράσουμε από κοινού. Είμαι πεπισμένο ότι μία από τι απαραίτητε προποθέσει για την ευόδοση ε, της υπέρβαση τη οικονομική κρίση είναι μια σωστά λειτουργούσα εσωτερική αγορά. Αυτό είναι ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα της Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση μέχρι στιγμή. Γι' αυτό και η, δημοκρατία, η Προεδρία η Τσεχική ενδιαφέρεται για την τήρηση των κανόνων που δέχτηκαν τα μέλη όταν συνυπέγραψαν τις συνθήκες προσχώρησης. Συνθήκες που δεν πρέπει να εφαρμόζονται μόνο στις καλές αλλά και στις κακές στιγμές των κοινωνιών μας. Η Ευρώπη χωρίς ε, φράγματα, χωρίς εμπόδια. Ε, δεν πρέπει να είναι μια Ευρώπη χωρίς κανόνες. Και γι' αυτό στηρίζουμε ένα υγιές ανταγωνιστικό περιβάλλον και την εξασφάλιση ενός δίκαιου πεδίου δράσης για όλους. Η Ευρώπη χωρίς φράγματα, περισσότερο από ποτέ, είναι προαπαιτούμενο μιας ανταγωνιστικής οικονομίας στο παγκόσμιο ιδίως επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην ιδέα των κοινών αξιών. Και η πιο σημαντική αξία είναι ασφαλώς η ιδέα της ελευθερίας. Η ελευθερία όμως έχει και μια οικονομική διάσταση. Μιλάμε για την ελευθερία της αγοράς, την ελευθερία να εκμεταλλεύεται κανείς το ταλέντο του, ανταγωνιζόμενος με άλλους παίκτες. Είναι η ελευθερία να επιλέγει κανείς ε, το γήπεδο στο οποίο θέλει να παίζει. Η Τσεχική Προεδρία θέλει να αποκαταστήσει την ε, πρωτοκαθεδρία της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Θέλουμε να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών. Γι' αυτό και θέλουμε να έχουμε έγκαιρη, γρήγορη και σωστή μεταφορά της ε, οδηγίας για την ενέργεια στο εσωτερικό δίκαιο των κρατών μελών. Η σχετική νομοθεσία ε, υιοθετήθηκε πριν από δύο εβδομάδες από τις κυβερνήσεις και έχει υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είμαστε η πρώτη χώρα που μετέφερε αυτό το δίκαιο, στη, αυτή τη νομοθεσία στο εσωτερικό της δίκαιο και σας βεβαιώνω ότι δεν ήταν εύκολο. Η μεταφορά αυτή, το, ο νόμος περί μεταφοράς της οδηγίας στο εσωτερικό μας δίκαιο καλύπτει δεκάδες νομοθετικά κείμενα σε διάφορους τομείς και αν θέλουμε να είμαστε εντάξει με, την, με τις προθεσμίες της οδηγίας για την ενέργεια, πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα σε όλη την Ευρώπη. Όσο αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών, αυτό είναι ένα θέμα πολύ αγαπητό σε εμά. Μέσα σε δύο, σε εβδομάδες από τώρα διοργανώνουμε μία, ένα συνέδριο για τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Και είναι χαρά μας να υποδεχθούμε πολλά μέλη της Επιτροπής σας σε αυτό το συνέδριο η φραγμή, τα εμπόδια στην ε, εσωτερική αγορά είναι ένα θέμα που θα συζητηθεί σε μια συνδιάσκεψη ε, το, Μάρτι... το Μάρτιο υπό την αιγίδα του κυρίου Πολάνεκ και του Επιτρόπου για την Ενέργεια καθώς και του Επιτρόπου Αλμούνια. Θα θέλαμε να σας θυμίσουμε ότι όλη η Ευρώπη έχει αποφεληθεί από την διεύρυνση. Το επόμενο θέμα είναι η ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών. Εκ μέρου ε, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή σας και τους εισηγητές, όλες τις ομάδες, για την πολύ καλή δουλειά που έκαναν κατά την εξέταση του πακέτου για την άμυνα. Η, συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση μπορεί να θεωρηθεί ως πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ σημαντική πρόοδος. πρόοδος. Η Τσεχική Προεδρία θα εξακολουθήσει να προσπαθεί να ρυθμίσει τις προϋποθέσεις της πρόσβασης στην αγορά για τους προμηθευτές και την απλοποίηση των σχετικών και την απλοποίηση αυτής της διαδικασίας. Συζητούμε κάποια νομοθετικά κείμενα για διάφορα προϊόντα, για καλλιντικά και επίσης για φυτοφάρμακα. Η οδηγία για τις κατασκευές θα μειώσει το διοικητικό φόρτο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και θα υπάρχει ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων κατασκευής, των κατασκευαστικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά. Αυτό θα συμβάλλει και στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς αυτοκινήτου μέσω της απλούστευσης ε, των διαδικασιών. Η Προεδρία μας επιθυμεί επίσης να απλουστεύσει τους κανόνες για τις επιχειρήσεις. Στον τομέα της καλύτερης ρύθμισης λοιπόν, θέλουμε να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και όχι μόνο. στο, υπάρχει επίσης και η μακροπρόθεσμη υποχρέωση να μειωθεί ο διοικητικός φόρτος των επιχειρήσεων κατά 25% μέχρι το 2012. Αυτός είναι ένας κοινό ευρωπαϊκός στόχος. Έχουμε συγκεντρώσει πολλή εμπειρία στην Τσεχία, όπου κόψαμε, όπου μειώσαμε από 20% στο 10% το σχετικό τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες και μπορώ να σας πω προσωπικά από τη δική μου εμπειρία ότι ήταν ένα από τα δυσκολότερα πράγματα που έκανα ποτέ. Ε, ξέρουμε ε, πολλές, μάλλον πολλές από τις λεπτομέρειες εξαρτώνται από την προσωπική αφοσίωση και δέσμευση και επιπλέον η δουλειά αυτή δεν σου αποφέρει άμεσα πολιτικά ωφέλη γιατί είναι αόρατη εν πωλής. Είναι, ε, είναι ένα καθήκον το οποίο δεν μπορείς να φέρει σε πέρα με επιτυχία διαρκώς και μακροπρόθεσμα. Το πετυχαίνεις μόνο που και που. Γι' αυτό και η προτεραιότητα της ε, Προεδρίας της Τσεχίας ε, στη για τη μείωση του διοικητικού φόρτου δεν πρέπει να αποτελεί δέσμευση μόνο της δικής μας Προεδρίας, αλλά όλων των Προεδριών. Γιατί διαφορετικά ποτέ δεν θα καταφέρουμε να μειώσουμε τις διοικητικές διαδικασίες επαρκώς. Ιδίως τώρα, σε εποχές ε, οικονομικών δυσκολιών, η μείωση του διοικητικού φόρτου είναι πιο σημαντική από ποτέ. Ιδίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τις οποίες το διοικητικό κόστος αποτελεί ένα πολύ σημαντικό, ένα πολύ μέρος του συνολικού κόστους. Είναι ανάγκη να συγκεντρωθούμε την προσοχή μας όχι μόνο στην κείμενη νομοθεσία όσο αφορά τη μείωση του διοικητικού βάρους, αλλά επιπλέον αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη και κατά την υιοθέτηση νέας νομοθεσίας. Πρέπει να επιμένουμε να αξιολογείται συνεπώς το διοικητικό κόστος στο πλαίσιο κάθε νέας πρότασης που υποβάλλει η Επιτροπή. τώρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τελευταίους έξι μήνες, μάλλον μέσα στους έξι μήνες της Προεδρίας μας, θέλουμε να υλοποιήσουμε συγκεκριμένα μέτρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σύμφωνα με το σχετικό σχέδιο και σύμφωνα με την νομοθεσία μας και ελπίζουμε να τα προχωρήσουμε πολύ τα θέματα αυτά. Θα θέλαμε να επιτευχθεί πρόοδος και με την οδηγία για, για τις πληρωμές η οποία θα δημοσιευθεί, θα εκδοθεί το Φεβρουάριο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από όσο ξέρουμε. Είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί πρόσβαση στους πόρους για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να δοθούν προνομιούχα δάνεια με τις σωστές εγγυήσεις. Και αυτό είναι απαραίτητο για να γίνονται και επενδύσεις, κυρίως επενδύσεις σε καινοτομία. Μιας και μιλάμε για επιχειρήσει, καλό είναι να μιλάμε και για επιχειρηματίε. Γιατί ο κύριος Μοχλός ε, ανάπτυξης ε, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι οι ίδιοι επιχειρηματίες. Σύμφωνα και με το Σύλλογο, ε, ο επιχειρηματίας γίνεται αντιληπτός στο πλαίσιο αυτών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ω ήρωα και πράγματι έτσι είναι. Ε, βεβαίως ο επιχειρηματίας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς πελάτες και χωρίς καταναλωτές. Και για να έχουμε πελάτες και καταναλωτές πρέπει να έχουμε μια εύρυθμη εσωτερική αγορά. Υπάρχει η οδηγία για την προστασία των οι οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών. Προτείνεται και ένα νέο κείμενο. Ε, η πρόταση αφορά την άρση εμποδίων, απλούστευση της κείμενης νομοθεσίας, ενημέρωση της κείμενης νομοθεσίας, επικαιροποίηση της έτσι ώστε να είναι πιο συμβατή με τις τρέχουσες συνθήκες. Φυσικά θα προσπαθήσουμε να διεξάγουμε τις ε, διαπραγματεύσεις και να τις ε, επεκτείνουμε όσο το δυνατόν περισσότερο ε, και να τις συζητήσουμε εξονυχιστικά. Πρέπει να είμαστε όμως ρεαλιστές. Για να επιτευχθεί πρόοδος πρέπει να ξέρουμε ότι η Προεδρία μας δεν έχει και πολύ χρόνο στη διάθεσή της. Έχει λίγο χρόνο στη διάθεσή της. Επομένως δεν μπορούμε να έχουμε και πολύ ωραία αποτελέσματα. Αυτή η πρόταση περιλαμβάνει πολλές αντιφάσεις ε, που συμπυκνώνουν τις διαφορετικές θέσεις των κρατών μελών και τη θέση των καταναλωτών σε αυτές. Ιδίως όπως όσον αφορά την αρχή της εναρμόνισης. Τα κράτη δεν θα μπορούν να διατηρήσουν διατάξεις ε, οι οποίες παρέχουν μεγαλύτερη προστασία. Δεν μπορούμε όμως να φανταστούμε να βασιστεί η οδηγία στο ανώτατο επίπεδο προστασίας που, την οποία εφαρμόζουν κάποια κράτη-μέλη. Ε, γιατί υπάρχουν ισχυρές διαφωνίες μεταξύ κρατών μελών. Αυτό είναι προφανές. Όταν συζητήθηκε η πρόταση αυτή σε εθνικό επίπεδο εμφανίστηκαν πολλά προβλήματα και γέρθηκαν πολλές αντιρρήσεις. Από την άλλη πρέπει να μην ξεχνάμε και τις θετικές εκφάνσεις αυτής της πρότασης, η οποία προσπαθεί να άρει τα εμπόδια της εσωτερικής αγοράς, να απλουστεύσει τις διαδικασίες και τις συνθήκες τόσο για τους επιχειρηματίες όσο και για τους καταναλωτές. Γι' αυτό ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί πρόοδος και θα βρεθεί ένα ισορροπημένο κείμενο που θα λαμβάνει υπόψη του όλες τις πλευρές. Έχω, υπάρχουν, ε, υπάρχει υλικό για τους υπουργούς που θα, ε, για την Σύνοδο Ανταγωνιστικότητας ε, που θα λάβει η χώρα τον Μάιο. Και εκεί θα επιτευχθεί κάποια πρόοδος. Έπειτα έχουμε το θέμα της εφαρμογής των δικαιωμάτων στην πράξη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την προστασία των καταναλωτών. Γι' αυτό παρακολουθούμε με μεγάλη προσοχή τις δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον τομέα αυτό. Η προσοχή μας αφορά την, ε, το θέμα της σωστής αποζημίωσης των καταναλωτών. Ε, δημοσιεύθηκε, όπως ξέρετε, μια πράσινη βίβλος για τις αποζημιώσεις των καταναλωτών, έχουμε κάποιες επιφυλάξεις. Δεν ξέρω αν είναι ανάγκη να εισαχθεί ένα, ένα σύστημα συλλογικής αποζημίωσης κοινή. Έχουμε κάποια αντίρρηση. Νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε τους ίδιους στόχους της Πράσινης Βίβλου χρησιμοποιώντας τα υφιστάμενα εργαλεία και μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Θα συνεχίσουμε την ε, διαδικασία αυτή διαβούλευσης και θα τα συζητήσουμε αυτά και στη Σύνοδο Ανταγωνιστικότητας που θα γίνει όπως είπα το Μάιο. Υποστηρίζουμε την παρακολούθηση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς τόσο στους καταναλωτές όσο και στους επιχειρηματίες. Τέλος, εν κατακλείδη, θα ήθελα να αναφέρω δύο προτάσεις που έχουν σχέση με, την, ε, με τις δραστηριότητε τις αρμοδιότητες επιτροπής σας. Πρώτον, τηλεπικοινωνίες. Είναι προτεραιότητά μας το πεδίο αυτό. Τα έχουμε, το συζητήσαμε και σήμερα το πρωί. Έχουμε το λεγόμενο πακέτο των τηλεπικοινωνιών. Θα συνεχίσουμε και εδώ το έργο που διεκπαιρέωσε η Γαλλική Προεδρία. Ήταν ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα. Ωστόσο το Συμβούλιο Υπουργών τον περασμένο φθινόπωρο ενέκρινε και υιοθέτησε ομόφωνα την δική του εκδοχή. Ξέρουμε ότι η εκδοχή του Συμβουλίου δεν βρίσκει σύμφωνο το Κοινοβούλιο και υπάρχουν πολλές διαφωνίες μεταξύ Επιτροπής Κοινοβουλίου και Συμβουλίου. Βρισκόμαστε μπροστά σε μια δύσκολη κατάσταση λοιπόν εδώ. Ελπίζουμε όμως ότι το πακέτο των τηλεπικοινωνιών θα εγκριθεί τελικά από την κοινή υπουργική συνάντηση για τις τηλεπικοινωνίες. Έχουμε τρεις μήνες μπροστά μας για να προσπαθήσουμε να καταλήξουμε σε ένα σχέδιο συμβιβασμού. Ε, είναι προς όφελος όλων των ε, πλευρών να επιτευχθεί η συμφωνία και αυτό μπορεί να γίνει μόνο αν όλες οι πλευρές επιδείξουν προθυμία ε, να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις, να υποχωρήσουν λίγο από τη διαπραγματευτική τους θέση. Το μεγαλύτερο μέρος του πακέτου είναι η οδηγία για τα δικαιώματα του πολίτη. Ομολογώ ότι η πρόταση αυτή ως μέρος του πακέτου τηλεπικοινωνίας δημιουργεί μια περίπλοκη και δύσκολη κατάσταση. Πρόκειται για δικαιώματα πολιτών και κυρίως δικαιώματα προστασίας των ιδιωτικών τους δεδομένων και της ιδιωτική του ζωής. Υπάρχει το θέμα της περιαγωγής στις τηλεπικοινωνίες. Οι υπηρεσίες Υπάρχει το θέμα ρύθμισης των υπηρεσιών περιαγωγής, το οποίο μας απασχολεί. Εμείς, η Δημοκρατία της Τσεχίας, είμαστε μεταξύ των λίγων χωρών που έχουν εκφράσει αμφιβολίες και επιφυλάξεις για το κατά πόσο η ρύθμιση των υπηρεσιών περιαγωγής γίνεται με το σωστό τρόπο. Νιώθουμε λίγο μόνοι βέβαια εδώ, έχουμε μείνει μόνοι, ίσως μαζί και με την Ιταλία. Βεβαίως, σε σχέση με την σημερινή κατάσταση, ελπίζουμε πως θα γίνουν συζητήσεις και οι συζητήσεις αυτές θα καταλήξουν σε κάποια πρόταση από την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Οι προτάσει των δύο οργάνων μέχρι στιγμή είναι αρκετά όμοιε και νομίζω ότι μπορούμε να τις πλησιάσουμε και στις θέσεις του Κοινοβουλίου και ελπίζουμε ότι θα επιτευχθεί συμφωνία κατά την πρώτη ανάγνωση ε, πράγμα που θα επιτρέψει την υιοθέτηση του πακέτου τηλεπικοινωνιών τον Ιούνιο. Κυρίες και κύριοι, αυτό με φέρνει στο τέλος της παρουσίασής μου Eh, eh, Νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικότερα σημεία που αφορούν την πολιτική μας για την εσωτερική αγορά και την προστασία του καταναλωτή. Ασφαλώς η Προεδρία μας, όπως είπα, δεν ε, ανελήφθη σε μια εύκολη συγκυρία. Ε, έχουμε μια σειρά οικονομικών προβλημάτων έχουμε τη λήξη της θητείας του Κοινοβουλίου, κάτι που συντομεύει ακόμα περισσότερο το χρόνο που έχει στη διάθεσή της η Προεδρία μας. Ελπίζουμε όμως ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία και στο τέλος της Προεδρίας μας θα μπορέσουμε να βγούμε και να πούμε ότι έχουμε κάνει πραγματικά Πρόεδρο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που αναφερθήκατε και στις δύο πτυχές τη εσωτερικής αγοράς. Αυτό αφορά δηλαδή και τις επιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Κάποιες κυβερνήσεις υποτιμούν το ρόλο των ε, καταναλωτών και το πόσο σημαντική είναι η προστασία τους. Θα πρέπει εδώ να τονίσω ότι η δημοκρατία της Τσεχίας έχει επιτύχει να να θεωρήσει 40 νομοσχέδια δικά τη και να θέσει σε ισχύ την ε, οδηγία για τις υπηρεσίες. Θα πρέπει όμως τώρα να ασχοληθεί με το συντονισμό των παρόμοιων ε, προσπαθειών και σε άλλες χώρες. Όσοι βρίσκονται λοιπόν εδώ, το τέλος της επόμενης χρονιάς, εφόσον βρίσκονται και πάλι εδώ, θα δουν κατά πόσον ε, μπορούμε να κάνουμε μια θετική αποτίμηση της υλοποίησης της οδηγίας και της υπηρεσίας. Επίσης, να θυμίσω και την ημέρα των καταναλωτών στις 16 Μαρτίου. Υπουργέ οργανώνεται στις Βρυξέλλες υπό την Προεδρία της κυρίας Χωνέβα και του κ. Μακάφη. Και θα ήθελα να απευθύνω την επίσημη πρόσκληση και σε εσά, σε κάποιον εκπρόσωπο του Υπουργείου σας, διότι αυτή η μερίδα είναι σημαντική. Θα ασχοληθούμε με θέματα που αφορούν άμεσα τους Ευρωπαίους καταναλωτές δώσατε έμφαση στο γεγονός ότι είναι αναγκαίο τα κράτη-μέλη να φτάσουν στο ύψος των ε, υποσχέσεων, που, μάλλον να ανταποκριθούν στις υποσχέσεις που έχουν αναλάβει. Ιδίω ό,τι αφορά την περίπτωση των αγαθών και την ε, εμπορία των αγαθών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λόγου χάρη, έχει ανεβάσει τον πύχη των προδιαγραφών για συγκεκριμένα αγαθά και προϊόντα. Και αυτά τα έχουμε εξετάσει και εδώ. Και τώρα να ζητήσω από τους συντονιστές να μιλήσουν εκ μέρους των πολιτικών ομάδων και να σχολιάσουν την παρουσίαση της Τσεχικής Προεδρίας. Πρώτος, ο κύριος Χάρμπορ. Σε ευχαριστώ, Σουζανά. Καταρχάς να καλωσορίσω και εγώ θερμά τον ε, Τσέχο Υπουργό. Να πω ότι είναι μεγάλη μας χαρά που η κυρία Ρόιτοβα προεδρεύει της συνεδρίασης, ο κύριος Μακόφη δεν είναι εδώ βέβαια σήμερα, όμως εσείς είσαστε μια πολύτιμη συνάδελφος και είναι πολύ καλή αυτή η σύμπτωση. Ε, να πω ότι είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι με τι φιλοδοξίε σα. Θέλετε να δώσετε και πάλι μια πρωταρχική θέση στην εσωτερική αγορά. Εμεί, ω μέλη τη Επιτροπή τη Προστασία των Καταναλωτών, νομίζουμε ότι σε κάποιο βαθμό έχουμε συνεισφέρει σε μια τέτοια προσπάθεια. Όμω, οπωσδήποτε πρέπει να εντείνουμε την ε, τάση αυτή. Όπω είπε και η Σουζάνα, σημαντικό για την Επιτροπή μα είναι να προχωρήσει η εσωτερική αγορά παράλληλα με την βελτίωση τη προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών διότι θέλουμε να έχουν ισχυρά δικαιώματα οι καταναλωτέ, να μπορούν να τα ασκούν ώστε να υποφελούνται πλήρω τη εσωτερική αγορά. Βρίσκω λοιπόν ότι αυτό ω στόχο είναι ήδη πολύ ενδιαφέρον. Επίση, θα ήθελα να μα πείτε λίγο περισσότερα, αν θέλετε, για τις φιλοδοξίες σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών και σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε και το πρωί ε, στην Επιτροπή μα. Νομίζω ότι δεν θα έχουμε χρόνο να περατώσουμε επί τη Προεδρία σα την πρώτη ανάγνωση τη σχετική πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμω νομίζω ότι θα επιτελέσουμε σημαντική πρόοδο, ιδίω κατά τη διερεύνηση των στατικικών, των ζωτικότερων θεμάτων, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και να ανοίξουμε το δρόμο για να περατωθεί η εξέταση του στην επόμενη Προεδρία. Ήθελα Επίση, να κάνω και κάποιε ακόμη παρατηρήσει. Ε, λόγω χάρη για το πακέτο των τηλεπικοινωνιών, το οποίο σχολιάσατε σε κάποιο βαθμό. Ε, ε, έχω αναλάβει συντονισμό, αλλά είμαι και εισηγητή για το θέμα αυτό και πρέπει να πω καταρχά ότι δεν ήμουν πολύ σαφής, δεν ήσασταν πολύ σαφείς για τη θέση που θα λάβετε εδώ. Εμείς στο Κοινοβούλιο είπαμε ότι θέλουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία δυνατόν το εξα... κατά τη διάρκεια του εξαμήνου της Προεδρίας σας. Όμως την ε, περασμένη Παρασκευή ήδη κυκλοφόρησε ένας κατάλογος με τις πολιτικές προτεραιότητες που θα να θέσουμε και κάποιες πρώτες ενδείξεις για ενδεχόμενες συμβαστικές λύσεις και ένα χρονοδιάγραμμα για το πώς θα πρέπει να γίνουν τα πράγματα. Έχω να σχολιάσω ότι πέραν της Ευρωπαϊκής Ένωσης θε, ε, μάλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση θέλουμε να φτάσουμε σε μια συμφωνία δυνατόν ε, τον Απρίλιο και ε, θα θέλαμε η δεύτερη ανάγνωση αν γίνεται να έχει ολοκληρωθεί γέρος. Όχι να μείνει το θέμα αυτό για τον Ιούνιο, άρα θα πρέπει να εντεθεί η συνεργασία μεταξύ μας. Επίσης υπάρχει και στις 17 Μαρτίου το Συμβούλιο για τις Τηλεπικοινωνίες, είναι νομίζω ιδιαίτερης σημασία. Και να πω και κάτι που έχω ήδη εντοπίσει στους συναδέλφους σας. Θα πρέπει οι σκιώδεις εισηγητές και οι εισηγητές, καθώς και οι πρόσωποι του Συμβουλίου, να συναντηθούν εγκαίρως, ώστε σε υπουργικό επίπεδο να επιληθούν ζωτικά ζητήματα, τα οποία μπορεί να παραμένουν εκκρεμοί. Αυτό είναι λοιπόν το μήνυμά μου προς εσάς. Εάν συμμερίζεστε την άποψή μας, εάν θέλετε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση τον Απρίλιο ήδη, θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να το πετύχουμε αυτό. Θα χρειαστούμε λοιπόν τη δική σα υποστήριξη για να το πετύχουμε. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έπειτα, κάτι που θα συζητήσουμε και σήμερα το απόγευμα. Πολλοί από εμά έχουμε ενδιασμού ε, για το να έχουμε υπέρμετρα αυστηρά και υπέρμετρα παρεμβατικά ε, υπερβατικού κανονισμού για την ε, εσωτερική αγορά. Το να θέσουμε όρια για την άνοδο των τιμών μπορεί να προκαλεί και επιζήμιες συνέπειες για τους καταναλωτές. Εδώ λοιπόν στηρίζουμε τις φιλοδοξίες της Επιτροπής να τονώσει τον ανταγωνισμό. Όμως δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα προηγούμενο για μακροχρόνιους ελέγχους και για ε, την υποβηγέτηση ε, της εσωτερικής αγοράς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν θέλουμε να γίνει κοινή αγροτική πολιτική αγορά της τηλεπικοινωνίας και να καθορίζει τιμέ ε, η Επιτροπή για μια σειρά από υπηρεσίε που παρέχονται μαζί με τι τηλεφωνικέ. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ούτω ή υπάρχει και η διεθνή περιαγωγή και τριών λογιών προϊόντα τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν στη διεθνή αγορά και μάλιστα ικανοποιητικά. Άρα θα πρέπει να το δούμε πολύ προσεκτικά αυτά και όχι απλώ να προσυπογράψουμε στην πρόταση τη Επιτροπή. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσουμε σε κάποια ζωτικά μέτρα σχετικά με τη διαφάνεια στον τομέα αυτό, τα οποία, χρειαζό, τα οποία θεωρούμε απολύτω απαραίτητα. Όμω μπορεί να κάνουμε και προτάσει για μια πολύ γενική απλώ ε, ε, συγκράτηση των τιμών. Όμως θα πρέπει να είμαστε πολύ συνετοί και προσεκτικοί σε σχέση με αυτό το δυσχερέ θέμα. Θα περιοριστώ σε αυτά νομίζω γιατί θα έχουν ε, και οι συνάδελφοι πολλά ερωτήματα να σα θέσουν για την οδηγία περί των ε, υπηρεσιών. Πάντως ε, χαιρετίζουμε τι φιλοδοξίε σα και ανυπομονούμε για τη συνεργασία μαζί σα, που μπορεί να μην κρατήσει πάρα πολύ σε χρονικό διάστημα μεν αλλά ελπίζουμε να έχει μακροχρόνιε συνέπειε. Η Εύελιν Κέπχα τώρα εκ μέρου των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα ε, να σας ευχαριστήσω κύριε Προεδρεύοντα που βρήκατε το χρόνο να μιλήσετε εδώ σήμερα για τις ε, προτεραιότητες στον τομέα της ενιαίας αγοράς και στο, από το παρελθόν έχει φανεί ότι είναι σωστό και σημαντικό να συναντιόμαστε η ε, οδηγία για τις υπηρεσίες έδειξε ότι μέσω της συνεργασίας όχι μόνο εντός ε, του Κοινοβουλίου αλλά και με το Συμβούλιο Υπουργών ε, είναι δυνατό να βρίσκεται μια ε, σωστή λύση η οποία όχι μόνο να λαμβάνει υπόψη τους εργοδότες αλλά και τους εργαζόμενους και θα ήθελα να έρθω έτσι σε ένα θεμελιώδης για μένα ερώτημα που με απασχολεί από τότε που διάβασα ένα άρθρο του Βάκλαφ Κλάους ε, για, ε, σε μια μεγάλη γερμανική εφημερίδα ε, σχετικά με την αξιοπρέπεια του εργαζομένου ως, τα δικαιώματα του εργαζομένου ως εμπόδιο στην έννοια αγορά. Αυτό με συγκλονίστηκε. Ήθελα λοιπόν να, ήθελα να σας ρωτήσω ε, πώς το βλέπετε εσείς αυτό. Θέλετε μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια και εγώ το ίδιο, χωρίς φραγμούς. Θέλετε ελεύθερη κυκλοφορία των ε, υπηρεσιών και εγώ το θέλω αυτό. Θέλετε ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και εγώ το ίδιο. Θέλετε μια πολύ ωραία ε, κοινοτική αγορά στην Ευρώπη και εγώ το ίδιο. Ε, δεν έχουμε καμία διαφορά στους στόχους μας. Αυτό είναι καλό. Όμως έχω την εντύπωση ότι με τον ορισμό, ε, ότι στους ορισμούς ε, αυτών που κρύβονται πίσω από αυτούς τους στόχους ε, υπάρχουν μεγάλα χάσματα. Θέλουμε να ε, διαμορφώσουμε μια κοινή ε, αγορά στην οποία να ε, παίζουν σημαντικό ρόλο τα δικαιώματα των εργαζομένων, θέματα περιβαλλοντικά κλπ. Εσείς όμως ενιαία αγορά λέτε την ελεύθερη αγορά. Εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω με κάτι τέτοιο. Εμείς οι σοσιαλδημοκράτες δεν μπορούμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο και Είδαμε ε, κατά την οικονομική κρίση που οδηγούν ε, αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει λοιπόν να συζητήσουμε τι ακριβώς ε, συμβαίνει και προς τα πού θέλουμε να κινηθούμε. Νομίζω ότι δεν θέλουμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεύτερον, η προστασία του καταναλωτή. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε εδώ στην Επιτροπή και συζητιέται και στο Συμβούλιο Υπουργών θέλουμε πλήρη εναρμόνιση ή όχι. Εγώ είπα σαφώς ότι θέλω να ε, σεβαστούμε αυτά που υπάρχουν στις συνθήκες. Ε, βρήκα και το σχετικό κείμενο, λέει στις ε, συνθήκες για την Ευρωπαϊκή Ένωση στο άρθρο 153, δεν θα σας διαβάσω το σύνολο διότι είναι μεγάλο άρθρο, αλλά η πέμπτη παράγραφος ε, είναι αυτή που μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, όπου λέει ότι ε, τα μέτρα ε, σύμφωνα με την παράγραφο 4 δεν εμποδίζουν τα κράτη-μέλη να διατηρήσουν ή να, εφαρμο... ή να υιοθετήσουν πιο αυστηρά μέτρα. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να συνάδουν με τη συνθήκη και να ενημερώνεται αναλόγως η Κομισιόν. Δεν θα πρέπει λοιπόν με, κάποιο, με κάποια λάθους τύπους, τύπου εναρμόνιση ε, να εμποδίσουμε κάποιο κράτος μέλος ε, να έχει πιο αυστηρούς κανόνες στην προστασία του καταναλωτή. Η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να ε, έχει προστιθέμενη αξία για τους καταναλωτές. Εάν πούμε εάν στην πλήρη εναρμόνιση ε ε, ε, ε, πάρουμε το, την, το υψηλότερο επίπεδο προστασίας που υπάρχει ε, σε κάποιο κράτος μέλος, τότε συμφωνώ. Εάν όμως με το μέσο όρο, τότε δεν συμφωνώ, διότι αυτό σημαίνει ότι ναι μεν θα ανέβει το επίπεδο σε κάποια κράτη-μέλη, θα κατέβει όμως σε κάποια άλλη, θα πέσει. και δεν μπορώ να δεχτώ κάτι τέτοιο. Θα πρέπει κάτι τέτοιο να το ξανασυζητήσουμε λοιπόν. Ε, τρίτο θέμα που θέλω να αναφέρω, γιατί δεν θέλω να μακρηγορήσω, ε, διαφωνώ με τον ε, συνάδελφο Μάρκορν Χάρμπορ. Μιλήσαμε για την τηλεφωνία, μιλήσαμε για την περιαγωγή και είπαμε αυτό θέλει η Κομισιόν. Αυτά θέλει και το Κοινοβούλιο. Εμείς ακούσαμε ε, τις ε, υπηρεσίες ε, κινητής τηλεφωνίας, της επιχειρήσης κινητής τηλεφωνίας. Εάν με τα μέτρα που λαμβάνονται διαπιστώσουμε ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός ειδικά στις διασυνοριακές υπηρεσίες, τότε θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε και νομίζω ότι το Ευρωπαϊκό ε, ε, Κοινοβούλιο και η ε, Κομισιόν θα πρέπει να τηρήσουν αυτά που υποσχέθηκαν στους καταναλωτές και ελπίζω το Συμβούλιο Υπουργών να μας ακολουθήσει και να κάνει ακριβώς αυτό. Δεν μπορούμε να δεχτούμε αυτοί που έχουν λιγότερα χρήματα να αποκλείονται από υπηρεσίες που σήμερα ουσιαστικά είναι γενικές. Επειδή οι υπηρεσίες αυτές θα είναι πιο ακριβές θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι και χρειαζόμαστε κανόνες είναι σαφές ότι η αγορά από μόνη της δεν ρυθμίζει τα θέματα αυτά. Υπάρχουν μονοπόλια τα οποία δεν μπορούμε να δεχτούμε. Θα πρέπει λοιπόν να αναλάβουμε δράση για να το ε, παρεμποδίσουμε αυτό. Και πρέπει, θα με συγχωρήσετε, δυστυχώς πρέπει να προλάβω ένα τρένο. Ε, πριν πολλούς μήνες είχα κλείσει ένα ραντεβού στο Παρίσι. Δεν γνώριζα το ότι θα είσαστε εδώ πέρα σήμερα, διότι στην περίπτωση αυτή δεν θα είχα ε, ε, ε, δεν, θα είχα κλείσει το ραντεβού αν ήξερα ότι θα είσαστε εδώ πέρα σήμερα. Ε, Δυστυχώ πρέπει να καταλήψω όμω ε, την αίθουσα. Δεν είναι επειδή δεν θέλω να ακούσω την απάντησή σα, αλλά θα με ενημερώσουν εκ των υστέρων οι, οι συνεργάτε μου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ενημερώσω τον Υπουργό ότι ακούσαμε σήμερα ότι η Κομισιόν θα στείλει λεπτομερή μελέτη στην Επιτροπή των Δικαιωμάτων των Καταναλωτών. Θα παρακαλούσα την κυρία Φουρτού να μιλήσει εκ μέρου ε, των φιλελευθέρων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ήρθατε σήμερα να μας μιλήσετε, διότι αναλαμβάνετε την Προεδρία σε μια στιγμή ιδιαίτερα δύσκολη και δυσχερή, θα έλεγα. Οπότε καλωσορίζουμε τις δεσμεύσεις σας ως φιλελεύθεροι Επίσης, ε, καλωσορίζουμε όσο είπατε για το διοικητικό άχθος και την ε, ενέργεια που πρέπει να καταβάλουμε για να το περιορίσουμε. Δεν θέλουμε να υπάρξει υπερβολική αυστηρότητα στα μέτρα που θα προβλέψουμε, οπότε ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουμε κατευθύνσεις πιο φιλελεύθερες και πιο ανοιχτόμυαλες προφανώς. Ήθελα να ρωτήσω σε ποια επίπεδο φτάνουν οι φιλοδοξίες σας για ένα θέμα που συζητούμε αυτή τη στιγμή, για τα οικοδομικά προϊόντα. Διότι εδώ βεβαίως, η συγγήτρια φαντάζομαι θα σας θέσει και ίδια κάποια ερωτήματα. Όμως, ποια είναι η άποψή σας για το συγκεκριμένο θέμα. Και θα σας ευχαριστήσω τον προτέρων για τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ. να προσθέσω ο πρόεδρος και εγώ ένα ερώτημα προς τον Υπουργό. Θα, θα ασχοληθείτε και με το θέμα του κοινοτικού σήματος, το σήμα CE, διότι ήδη έχουν γίνει σχετικά συζητήσεις, έχουν ακουστεί πολλά Και έχει γίνει συζήτηση και για το σήμα CE+, ένα ακόμα πιο ενισχυμένο σήμα. Όμως, ε, ακόμα όμως μας απασχολεί το θέμα του σήματος CE της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Πολλέ είναι επιχειρήσει που δεν ξέρουν ακριβώ πώ να αξιοποιήσουν την ύπαρξη του σήματο αυτού. Σε ποια κατάσταση λοιπόν βρισκόμαστε, θα μπορούσε να μα πει κάτι και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γι' αυτό. Πώ θα προστατεύσουμε τα σήματά μα, τι δικέτε μα. Ε, μιλάμε για μια προσπάθεια προστασία εδώ του κοινοτικού μα σήματο. Και επίση θα παρακαλούσα τον Υπουργό αν ήθελε να απαντήσει στα ερωτήματα των ε, συντονιστών. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε, ε, απαντώντας σε αυτά που υπόθηκαν εδώ πέρα, να πω καταρχάς ότι είναι κρίμα που έφυγε, η κυρία Γκέπχαρτ, διότι θα είχαμε πολλά να πούμε νομίζω αν είχε μείνει. Αλλά σε ό,τι αφορά τις παρατηρήσεις του κυρίου Χάμπορ, Χρειάζονται περισσότερα βήματα στον τομέα της προστασίας των καταναλωτών. Σαφώς και όσο για την πρόταση που έχουμε προς εξέταση, θα προσπαθήσουμε να καταβάλουμε όσο δυνατόν μεγαλύτερη πρόοδο στο επίπεδο των ομάδων εργασία του Συμβουλίου που ασχολούνται με το συγκεκριμένο ζήτημα και ελπίζουμε ότι όλη αυτή η επεξεργασία θα οδηγήσει σε τη δημιουργία ενό καλού προηγουμένου, στο οποίο να βασιστεί η Σουηδική Προεδρία για να ολοκληρώσει την εξέταση του θέματο. Αν και πιστεύω ότι το θέμα αυτό περιέχει πολλέ παγίδε, διότι οι παρεμβάσει σα σήμερα εδώ προ αυτό το στοιχείο καταδεικνύουν. Η Γαλλική Προεδρία έκανε ό,τι καλύτερο μπορούσε για το συγκεκριμένο θέμα. Και πέτυχε να συζητήσει τελικά 12 από τα 50 άρθρα της ε, εν λόγω πρότασης. Φανταστείτε. Δεν είναι πολύ ρεαλιστικό να περιμένουμε ότι τα υπόλοιπα 38 άρθρα θα προλάβουμε να τα εξετάσουμε πλήρως επί Τσεχικής Προεδρίας. Οι ομάδες εργασίας συναντώνται δύο φορές το μήνα. Αρκετά συστηματικά θα έλεγα και η πρώτη συνεδρίαση έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα. Άλλη μια συνεδρίαση πρόκειται να διεξαχθεί την επόμενη εβδομάδα. Άρα, σαφώ θέλουμε να προωθήσουμε το όλο θέμα, όμως θα πρέπει να είμαστε και λίγο πραγματιστές. Θέλουμε να είμαστε προσγειωμένοι σε ό,τι αφορά τι ε, προσδοκίε μα. Και η κυρία Γκέμπχαρτ είπε ακόμη ότι η πλήρης εναρμόνιση σημαίνει ότι τίποτε δεν θα πρέπει να εμποδίζει τα κρατημέλη να μπορούν να υιοθετήσουν μέτρα που να εξασφαλίζουν υψηλότερο επίπεδο προστασίας από εθνικής σκοπιάς. Φαντάζομαι λοιπόν ότι η σχετική συζήτηση θα είναι αρκετά ταραχώδη. Δεν νομίζω να έχουμε τελικά πλήρη εναρμόνιση, αλλά τουλάχιστον μια ελάχιστη εναρμόνιση. Αυτό ελπίζουμε. Σε ό,τι αφορά το πακέτο τηλεπικοινωνιών και τη δική μου την απεσιοδοξία. Όπω είπατε κύριε Χάμπορ, δεν θα έλεγα ότι είμαι ακριβώ απεσιόδοξο σε ό,τι αφορά το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει εδώ η δική σα επιτροπή. Όμω θέλω να είμαι ταυτόχρονα και πραγματιστής. Δηλαδή, υπάρχουν ε, πτυχέ του ντοσχέ αυτού του όλου θέματο, ε, οι οποίε ε, υπόκειται στην αρμοδιότητα τη Επιτροπή Ήτρε. Επίση, το Συμβούλιο των Υπουργών, στην τελευταία του συνάντηση Γαλλικής Προεδρίας ενεργοποιήθηκε Ιδιαίτερο και όλε οι συνεδριάσει που οργανώθηκαν σε αυτό το εξάμεινο, το προηγούμενο δηλαδή, ε, κατέβαλαν μεγάλε προσπάθειε για να πετύχουν ομοφωνία. Και για έναν πολύ απλό λόγο. Υπάρχει σαφώ η ένδειξη ότι εάν το Συμβούλιο καταφέρει να φτάσει σε ομόφωνη απόφαση, τότε μπορεί να δημιουργήσει, να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρία που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπλοκάρει την πρόταση. Αυτό λοιπόν ε, είναι γνωστό σε όλους αυτή τη στιγμή και κατά τη διάρκεια της διαδικασίας των διαπραγματεύσεων ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι υπάρχει σαφής ε, πρόθεση των κρατών μελών όπως φάνηκε από την ομόφωνη ψηφοφορία και συμφωνία στο Συμβούλιο των Υπουργών την τελευταία φορά. Τώρα, για την επερχόμενη συνάντησή του τον Ιούνιο, για το επερχόμενο Συμβούλιο του Ιουνίου. Είχαμε σκεφτεί ότι το σημείο αυτό θα περιληφθεί ως σημείο προς έγκριση στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου. Για την περιαγωγή, συμφωνώ ότι δεν θέλουμε πάλι να δημιουργήσουμε μια πολιτική ανάλογη της κοινή αγροτικής, όμως, να είστε βέβαιοι ότι θα βασιστεί και στην κοινή της λογική εδώ η ε, τσεχική προεδρία. Θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο είναι αρκετά εύστοχο στάση. Ε, παρόλα αυτά, πιστεύουμε κιόλα ότι καλό είναι να έχουμε ξεκάθαρες ιδέες εδώ. Γι' αυτό και τις ανέφερα προηγουμένως. Άλλωστε, η χώρα που προεδρεύει στο Συμβούλιο δεν έχει σκοπό να κάνει κατάχρηση της θέσεις της ως προεδρεύουσας ε, για να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα και θέσεις. Ο ρόλος μας μάλλον τον αντίθετο σκοπό έχει. Θέλουμε να οδηγήσουμε σε συμφωνία, να δημιουργήσουμε το πεδίο για μια συνένεση μεταξύ των ε, κρατών μελών. Άρα, σε ό,τι αφορά την περιαγωγή, θα αφήσουμε τη συζήτηση να εξελιχθεί ανάλογα με τις επιθυμίες όσων θέλουν να ρυθμιστεί κατά κάποιο τρόπο η υπηρεσία της περιαγωγής, οι υπηρεσίες της περιαγωγής. Δηλαδή θα την αφήσουμε τη συζήτηση αρκετά και στα χέρια του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εάν Μα ρωτάτε τι προτιμούμε, την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου ή τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα έλεγα ότι βρισκόμαστε πιο κοντά στην τοποθέτηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, που συνάδει περισσότερο και με του δικού μα σκοπού. Όμω, ε, σε κάθε περίπτωση να είστε βέβαιοι ότι θα ασκήσουμε το ρόλο διαμεσολαβητού που μπορεί να διαδραματίσει σε, αυτέ τι διαπραγματεύσει η προεδρεύουσα χώρα. Ε, ε επίσης για τι παρατηρήσει του κυρίου Χάρμπορ. Νομίζω ότι απάντησα τόσο σε εκείνον όσο και στην κυρία Γκέπχαρτ. Τώρα για το άρθρο του κυρίου Κλάου στην γερμανική εφημερίδα και την προστασία των εργαζομένων που αναφέρατε. Δεν το γνωρίζω επακριβώς, όμως σε γενικές γραμμές φαίνεται να υπάρχει σαφής διάθεση για να συζητηθεί εδώ το θέμα και από τη σκοπιά δύο διαφορετικών κοσμοθεριών. κοσμοθεριών κοσμοθεωριών, συγγνώμη. Το θέμα είναι τι μέτρα θα λάβουμε. Τον φθινόπωρο ήμουν στο Βερολίνο και έμαθα ότι μια Ινδική εταιρεία με περισσότερους από χίλιους εργαζομένους δεν έχει δικαίωμα να απολύσει τους εργαζομένους αυτούς σε καμία περίπτωση χωρίς έγκριση της κυβέρνησης. Είμαι βέβαιος ότι τέτοιου είδους φραγμοί μπορούν να παρακαμφθούν από κάποιους ε, με την διαίρεση κάποιων ε, ομίλων, την διάσπασή τους σε διαφορετικές εταιρείες. Οπότε η πολιτική μας τοποθέτηση δεν είναι το να αποφασίσουμε αν θα πρέπει να υπάρξουν κανόνες ή όχι. Είναι σαφές ότι χρειάζονται κανόνες. Η συζήτηση θα πρέπει να επικεντρωθεί στο τι οι ευρωπαϊκοί οι κυβερνητικοί κανόνε θα πρέπει να διέπουν και τι είναι απολύτω απαραίτητο. Νομίζω λοιπόν ότι η συζήτησή μα για την περιαγωγή ακριβώ αποδεικνύει αυτό που σας εξηγώ. Ε, νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα ζητήματα συμπεριλαμβανομένη τη περιαγωγής. Κυρία Ρόιτοβα, νομίζω ότι στη διάρκεια των εντατικών μας συζητήσεων το καλύψαμε αυτό που αναφέρατε και να πω ότι γενικά θεωρώ ότι αυτή είναι μια καλή πρωτοβουλία. Ωστόσο, υπάρχει εδώ ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα. Δηλαδή, το σύνολο των κανόνων μα θα πρέπει να καταρτιστεί κατά τον τρόπο τέτοιον ώστε να μην μπορούν να παρακαμφθούν κάτι που σήμερα σαφώς συμβαίνει. Θα είναι δύσκολο λοιπόν οι νέε μας διευθετήσεις να μας οδηγήσουν στο να αποφύγουμε πλήρως κάθε είδους παράκαμψη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας, αν και το πρόβλημα αυτό πρέπει να πω ότι είναι ουσιαστική σημασία ε, για την κοινωνία μας και τον τρόπο που λειτουργούν οι κανόνες. Η κυρία Σεζίνσκα, ευχαριστώ. Υπουργέ, επιτρέψτε μου να σας καλωσορίσω. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα με τον ήχο. Χαιρόμαστε που σας καλωσορίζουμε στην Επιτροπή μας. Ε, και το τέλος της θητείας μας συμπίπτει με τη Τσεχική Προεδρία. Η κυρία Φορτού ε, σας ρώτησε σχετικά με την ε, οδηγία για ε, τα συγκεκριμένα προϊόντα σε μια Ευρώπη χωρίς φραγμούς. Θα ήθελα εγώ να αναφερθώ στον τομέα οικοδομικών κατασκευών μα ενδιαφέρει να εναρμονίσουμε ε, τους βασικούς κανόνες ε, ε, του σήματος e και να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα παραγωγών και καταναλωτών. Θέλουμε να απλοποιήσουμε την νομοθεσία, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και γι' αυτό ετοιμάζουμε πολλά συγκεκριμένα μέτρα στον τομέα αυτών. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Η Τσεχική Προεδρία θα επιδιώξει να κλείσει τις συζητήσεις ε, για την ρύθμιση των ε, προϊόντων ε, οικονομικής κατασκευής με την πρώτη ανάγνωση μέχρι τον Μάιο του 2009. Ποια είναι η θέση της ε, Προεδρίας σχετικά με, την, ε, ε, σχετικά με το σήμα CE. Αυτό είναι ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει από τότε που υιοθετήσαμε το πακέτο για την διάθεση στην αγορά των προϊόντων. Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με την προστασία των καταναλωτών. όταν η Τσεχική Προεδρία θα... Η Τσεχική Προεδρία θα πρέπει να γνωρίζει ότι τα νέα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν πολλά πράγματα για να φτάσουν τις, τα κράτη-μέλη της Ευρώπης των 15 και γι' αυτό η παρατήρησή μου είναι ότι ε, μόνο ε, καλά χρηματοδοτημένοι και ε, καλά χρηματοδοτημένε μη κυβερνητικέ οργανώσει ε, ε, θα μπορέσουν να ασχοληθούν με τέτοιες διαμάχες. Τι προβλέπει η Προεδρία για να αυξήσει την οικονομική υποστήριξη των μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με την προστασία του καταναλωτή. Πρόεδρος, θα ήθελα να σημειώσω ότι έχει αναβάλει την ψηφοφορία τη η Επιτροπή ώστε η Προεδρία να μπορέσει ε, να ασχοληθεί με την πολύ σημαντική ε, αυτή οδηγία. Η κυρία Χάνσλικ ε, από το ΕΛΚ. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ που ε, ήρθατε εδώ στην ε, συνεδρίασή μας. Ε, θα ήθελα να αναφέρω δύο πράγματα. Αναφερθήκατε εσείς στην οδηγία για τις υπηρεσίες και τη μεταφορά της στα κράτη-μέλη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα, δεδομένου ότι πλησιάζει το 2010. Φτάνουμε δηλαδή στο τέλος της προθεσμίας για τη μεταφορά της οδηγίας αυτής στις διάφορες χώρες. Ε, αναφέρθηκε ότι η Τσεχία ήδη έχει εφαρμόσει 40 νομοθετήματα, αλλά τι ισχύει στις άλλες χώρες ε, και πώς βλέπετε εσείς την κατάσταση. Τι ισχύει για τις ε, ηλεκτρονικές διαδικασίες στα διάφορα κρατημέλη. Ξέρουμε ότι η Κομισιόν θα προτείνει ένα πρόγραμμα, ένα σύστημα. Πώς όμως αξιολογείτε εσείς τα συστήματα στα διάφορα κρατημέλη. Πιστεύετε ότι η μεταφορά αυτή στο εθνικό δίκαιο πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση και θα έχουμε αρκετό χρόνο μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2010. Ε, αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. Η δεύτερη είναι η εξή. Θα ήθελα να ξέρω εάν κατά τη διάρκεια της Προεδρίας σας προβλέπετε την καταπολέμηση της απάτης και της πειρατείας. μπορείτε να αναφερθείτε στο Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την καταπολέμηση της απάτης. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, κύριε Ρούτοβιτς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σας καλωσορίζω στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την παρούσα πολιτική της Τσεχικής Προεδρίας. Βλέπουμε αυξήσεις των τιμών σε πολλούς τομείς, σε υπηρεσίες κοινής ωφελίας κλπ. Και ενώ ταυτόχρονα βλέπουμε ε, σημαντικές απολύσεις. Ε, βλέπουμε πολιτικές απειλές, βλέπουμε εξωσικομούς και θα ήθελα γι' αυτό να σας ρωτήσω τι κάνετε στα πλαίσια της πολιτικής υπέρ των καταναλωτών για να μειώσετε, να περιορίσετε αυτά τα δυσάρεστα φαινόμενα τα οποία ε, επηρεάζουν ε, κυρίως ε, τις πιο στερημένες ομάδες. Δεύτερον, όσον αφορά την περιαγωγή, είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία. ε, ιδιαίτερα καθότι η μία πλευρά θεωρεί ότι είναι πιο ισχυρή από την άλλη. Θα θυμάστε τις καθυστερήσεις που είδαμε στη μείωση των τιμών ε, περιαγωγής. Και θα ήθελα γι' αυτό να αναφερθώ σε ισχυρά διοικητικά μέτρα, διότι οι υπάροχοι υπηρεσιών αυξάνουν τις υπηρεσίες, μεγιστοποιούν το κόστος, ενώ η κοινωνία γενικά επηρεάζεται από την αύξηση των τιμών. Είναι σημαντικό και γι' αυτό ήθελα, κυρία Υπουργέ, να σας ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι πρέπει να επιταχύνουμε τα μέτρα για την προστασία των Ευρωπαίων καταναλωτών στον συγκεκριμένο τομέα. Τελευταία παρατήρηση της κυρίας Νέρης. Μπορείτε παρακαλώ να είστε σύντομοι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και κύριε Υπουργέ. Χαίρομαι που είσαστε εδώ ε, μαζί μας ε, σήμερα. Ε, θα ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις διότι μου φαίνεται πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή που, παίρνετε, που αναλαμβάνετε την Προεδρία να γνωρίζω ποια είναι η προτεραιότητα των προτεραιοτήτων. Ε, για μένα ε, είναι και ελπίζω να συμφωνείτε και εσείς μαζί μου αν ε, εξετάσουμε τον κατάλογο των θεμάτων ε, που συζητήθηκαν σήμερα μιλάμε για εναρμόνιση και μέχρι να έχουμε οριζόντια εναρμόνιση θα είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσουμε πόσο έχουν προχωρήσει οι ευρωπαϊκές πολιτικές στους διάφορους τομείς ε, ιδιαίτερα στην ενιαία αγορά και στην προστασία των ε, δικαιωμάτων του καταναλωτή. Υπάρχει το θέμα της δικαιοσύνης για τους ε, καταναλωτές. Έχουμε την κινητή τηλεφωνία, έχουμε την περιαγωγή, όπου, που είναι σαφής σε τομείς όπου μιλάμε για τέτοια πράγματα. Υπάρχουν όμως πολλοί τομείς όπου δεν ε, προστατεύονται επαρκώ οι καταναλωτές, ε, όχι μόνο στις δικές μας χώρες, αλλά ε, και στις προσπάθειες εξάλληψης φραγμών ώστε οι καταναλωτές να χαίρουν τις ίδιες προστασίες με τις επιχειρήσεις στις αγορές. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να έχουμε όλο και περισσότερη Ευρώπη στις πολιτικές της ε, Κομισιόν που έχουν ανακοινωθεί για την ενιαία αγορά. Αυτό το θεωρώ ζωτική σημασία, θεωρώ ότι αποτελεί προτεραιότητα ε, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της θητείας μας. Ε, πιστεύω ότι αυτό είναι ένα θέμα προτεραιότητας το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, έχετε 10 λεπτά το πολύ, διότι ε, θα πρέπει να ε, αποχωρήσει ο κύριος Υπουργός ε, για μια συνέντευξη τύπου. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Είμαστε υπέρ του, της μέγιστης εναρμόνισης με κανονισμούς και με το νέο νομοθετικό πλαίσιο με το σήμα CE ε, ε, θα έχουμε μία και μοναδική υποχρεωτική επισήμανση. Θα θέλαμε να πετύχουμε συμφωνία κατά την ε, πρώτη ανάγνωση στις 9 Μαρτίου και είμαστε διατεθειμένοι να καταλήξουμε σε συμβιβασμό για τις απλοποιημένες διαδικασίες για το σήμα ε, πιστεύω ότι υπάρχει καλή βούληση και από τις δύο πλευρές ε, και σίγουρα συμφωνώ με αυτά που είπατε. Όσον αφορά τις οργανώσεις καταναλωτών, ε, είναι θέμα των μεμονωμένων κρατών μελών να ασχοληθούν με το ζήτημα και πιστεύω ότι θα πρέπει να παραμείνει αυτό έτσι, διότι σε κάθε κράτος μέλος υπάρχουν διαφορετικές συνθήκες, υπάρχουν διαφορετικές διαφορετικές ε, δομές ε, οργανώσεων προστασίας του καταναλωτή. Ε, η αρχή της επικουρικότητας εδώ πέρα λοιπόν η αρχή της επικουρικότητας νομίζω ότι είναι η καλύτερη αρχή που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Όσον αφορά την οδηγία για τις υπηρεσίες, η κυρία Χάνσλικ ρώτησε ποια είναι η κατάσταση στα άλλα κράτη-μέλη. Θα πρέπει να μάθουμε πώς έχει η κατάσταση στα άλλα κράτη-μέλη για να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες ως προς ε, την ε, προθεσμία. Ε, θα έχουμε άτυπη υπουργική διάσκεψη στην Πράγα, όπου το θέμα αυτό θα είναι το κύριο θέμα στην ημερησία διάταξη. Η οδηγία για τις υπηρεσίες, κατά τη γνώμη μας, είναι πολύ σημαντική, είναι ζωτικής σημασίας, ωστόσο πρέπει να αναφέρω ότι θα πρέπει να εφαρμόζεται ε, στα πλαίσια των εθνικών νομοθεσιών ε, με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Δεν ε, μπορούμε να παρέμβουμε στα διάφορα κράτη-μέλη. Η μόνη δυνατότητα παρέμβασης ανήκει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο όσον αφορά την απάτη και την πειρατεία. Αυτό είναι πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε κυρίως σε σχέση με τρίτες χώρες. Όπως ε, σας είπα χθε, ε, θα πρέπει να κάνουμε χρήση όλων των ε, διαθέσιμων μέσων που έχουμε για την εμπορική πολιτική και θα πρέπει να προωθήσουμε την δημιουργία αρμόδιων αρχών στα διάφορα κράτη-μέλη. Στο Υπουργείο μας έχουμε πολλά προβλήματα λόγω παραποιημένων προϊόντων, ιδιαίτερα στα σύνορα με τη Γερμανία και την Πολωνία. Για να απαντήσω στο ερώτημα του κύριου Ρούτοβιτς, ε, νομίζω ότι είναι σαφές και το είπα και πριν, οι προσωπικές μου θέσεις, ε, αλλά βέβαια πρέπει να κάνω διάκριση ανάμεσα στις προσωπικές μου θέσεις και τις επίσημες ε, θέσεις της Προεδρίας. Η προσωπική μου θέση πάντως ως προς την διαμόρφωση των τιμών είναι ότι με ακόμα μεγαλύτερη ρύθμιση των τιμών από ό,τι έχουμε αυτή τη στιγμή ε, θα έχουμε οπισθοχώρηση. Δεν συμφωνώ ότι οι τιμές θα πρέπει να ρυθμίζονται επειδή ο κόσμος φτωχαίνει. Μιλάμε για περιαγωγή, μιλάμε για διασυνοριακή επικοινωνία. Αυτό που μόνο του δείχνει ότι ο κόσμος δεν φτωχαίνει, διότι εάν συνέβαινε αυτό δεν θα είχε χρήματα να κάνει τηλεφωνήματα διασυνοριακά. Μπορείτε να διτάξετε ότι στο παρελθόν ε, δεν υπήρχαν ε, κινητά τηλέφωνα. Είχαμε όμως σταθερά τηλέφωνα. Τώρα ο κόσμος έχει περισσότερα ε, χρήματα από ό,τι είχε στο παρελθόν. Ε, η τελευταία, ως προς την τελευταία παρατήρηση και το ελάχιστο επίπεδο εναρμόνισης. Και εγώ το παρορίτερα στη συζήτηση και από άλλους ακούστηκε. Η συζήτηση θα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη και στο μέλλον. Θα είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουμε σε συμφωνία σχετικά με το επίπεδο εναρμόνισης. Θα πρέπει να έχουμε ελάχιστη ή μέγιστη εναρμόνιση ή να έχουμε απόλυτη ενερμόνιση που δεν θα επιτρέπει καμία απόκληση ούτε προς τα πάνω ούτε προς τα κάτω. Οχτώ άρθρα απομένουν να συζητηθούν. Ε, θα συντονίσουμε τη συζήτηση, δεν θέλω όμως να προδικάσω το αποτέλεσμα. Συμφωνούμε στην αρχή της πλήρους εναρμόνισης. Ο βαθμός εναρμόνισης όμως ε, θα πρέπει ε, να καθοριστεί πολύ προσεκτικά. για να μην καταργήσουμε βασικές αρχές. Δεν θέλουμε να κάψουμε τα ε, χλωρά μαζί με τα ξερά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Κάποιες ε, ε, παρατηρήσεις για την περιαγωγή να σας εξηγήσω τη θέση του Κοινοβουλίου. Χρειάστηκε να αλλάξουμε την κατάσταση, διότι ο κόσμος από το νέο, από το βορρά πληρώνανε στο νότο το δεκαπλάσιο από ό,τι πλήρωναν ε, οι πολίτες από το Νότο όταν πήγαιναν στο Βορρά. Και τώρα κοιτάμε τα θέματα του διαδικτύου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη. Γι' αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Είναι ένα θέμα πολιτικό και η Τσεχική Προεδρία φαίνεται να έχει πολλή ενέργεια η Τσεχική Δημοκρατία δεν αποτελεί μια από τις πλουσιότερες χώρες. Έχει αποφασίσει λοιπόν να ασχοληθεί με το θέμα. Επιτρέψτε μου να απαντήσω. Δεν ήθελα να επικεντρώσω τη συζήτηση στην περιαγωγή, αλλά είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Υπάρχουν ε, διαφορές ανάμεσα ε, στις τιμές των διαφόρων ε, επιχειρήσεων στις διάφορες χώρες, αλλά θα πρέπει να ρωτήθει κανείς σχετικά με τη λειτουργία των ε, εταιριών τηλεπικοινωνιών στον Νότο και στο Βορρά. Ποιο είναι το επίπεδο ανταγωνισμού σε κάθε δεδομένη χώρα. Πόσες επιχειρήσεις υπάρχουν στην αγορά σε κάθε χώρο, ποια είναι η πολιτική τιμών τους. Κάποιοι, κάποιες επιχειρήσεις επικεντρώνονται σε κάποιες πτυχές, σε άλλες σε κάποια άλλα πράγματα στη διαμόρφωση των τιμών τους. Προτού λοιπόν αναλάβουμε ε, δραστική, διοικητική, ε, δραστικά διοικητικά μέτρα θα πρέπει να κοιτάξουμε την δομή των αγορών, να δούμε αν το κανονιστικό πλαίσιο για τις αγορές αυτές ε, είναι στρεβλωμένο και μόνο κατόπιν θα πρέπει να αναλάβουμε διοικητική δράση. Χωρίς εις βάθος ανάλυση των αγορών δεν μπορούμε να αρχίσουμε να τις καταστρέφουμε. Αυτά λέει η Πρόεδρος. Όσον αφορά τις εθνικές αγορές. Ωστόσο, χαίρομαι που ήρθατε. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να συνομιλήσετε μαζί μας. Θα ήθελα να ενημερώσω τους υπόλοιπους ε, βουλευτές ότι ε, Έχω συζητήσει και άλλα θέματα με τον Υπουργό, όπως είναι τα τυχερά παιχνίδια, ε, η διασυνοριακή ε, ε, φροντίδα υγείας κλπ. Και είναι ενήμερος ο Υπουργός. Δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα στη θητεία μας. Ίσως όμως να προλάβετε να μας επισκεφτείτε τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Okay. Okay, we will continue straight away. Να συνεχίσουμε ευθύς αμέσως. Θα ξεκινήσουμε με τα τεχερά παιχνίδια. Κυρία Σάλντε Μόζε. Ευχαριστώ. Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρον το θέμα και θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους ε, συναδέλφους ε, που υπέβαλαν τόσες τροπολογίες. 149 τροπολογίες έλαβα για την ε, έκθεση των τυχερών παιχνιδιών σε απευθεία σύνδεση. Ε, ακούγεται χειρότερη η κατάσταση από την διότι νομίζω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε καλές, ε, κάποιους καλούς συμβιβασμούς, ώστε να ε, έχουμε τελικά μια καλή έκθεση. Διαβάζοντας τις ε, τροπολογίες, βλέπω σαφώς ότι Υπάρχουν δύο βασικές γραμμές στις τροπολογίες και ο βασικός πυρήνας στις δύο βασικές γραμμές αυτές είναι ότι από τη μία έχουμε μια σειρά τροπολογιών ε, σχετικά με ε, τις ε, συγκεκριμένες ε, προτάσεις ε, αλλά και τα εκτιμώντας. Η γραμμή αυτή είναι ότι τα τυχερά παιχνίδια σε απευθεία σε σύνδεση θα πρέπει να τα εξετάσουμε ως μια κανονική οικονομική δραστηριότητα και γι' αυτό η εσωτερική αγορά, το ευρωπαϊκό δίκαιο θα πρέπει να έχει το κύριο βάρος εδώ πέρα. Απ' την άλλη έχουμε μια σειρά τροπολογιών που ε, θεωρούν ότι ε, αποτελεί μια αρνητική δραστηριότητα, ε, αποτελούν τα τυχερά παιχνίδια αρνητική δραστηριότητα και θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για να ε, παρεμποδίσουμε την εξαπλωσή τους και έτσι τα κράτη-μέλη έχουν ένα θεμητό συμφέρον να διατηρήσουν την ομοθεσία τους στον τομέα αυτών. Έχουμε λοιπόν αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις. Ακόμα και αν ε, οι τροπολογίες δεν το λένε αυτό ρητά, αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στι δύο κατευθύνσεις. Και ε, σκέφτηκα πώς θα πρέπει να ε, παρουσιάσω το θέμα σήμερα για να είναι σαφέ για του συναδέρφους σε ποιες τροπολογίες ε, στηρίζω και ποιε όχι. Και νομίζω ότι τελικά κατέληξα ότι ο ευκολότερος τρόπος να γίνω κατανοητή είναι να πω τα εξής. Πιστεύω ότι είναι δυνατό να καταλήξουμε σε πολύ, καλούς, σε πολύ καλές συμβαστικές τροπολογίες μεταξύ ε, των τροπολογιών του κυρίου Μάντερς, ε, του κυρίου Τουρών, της κυρίας ε, και, Κορόλα και της της δικές μου. Νομίζω ότι μεταξύ των τροπολογιών αυτών θα είναι εύκολο να βρούμε κάποιες συμβαστικές, καλές συμβαστικές τροπολογίες. Του Ναντίον. Δεν επιθυμώ η ε, έκθεσή μου να πάει προς την κατεύθυνση ε, που επιθυμούν ε, η κυρία Κάριν Ρίση ο κύριος Ντάν, ο κύριος Φιέλνερ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να βρούμε καλές συμβαστικές τροπολογίες και μεταξύ αυτών, αλλά αυτή είναι η βασική μου κατεύθυνση. Να αναφερθώ στα επιμέρους θέματα γίνονται κάποιες συζητήσεις σχετικά με το σε τι βαθμό η έκθεση θα πρέπει να αναφέρεται στην ε, αρχή της ε, επικουρικότητας, την ομολογία του δικαστηρίου και τέτοια θέματα. Μιλάω για τις ε, τροπολογίες 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Αυτή είναι μία κατηγορία. Και ευχαρίστως να συμβιβαστώ, να αναφέρουμε την ομολογία του δικαστηρίου. Θέλω όμως επίσης να επιμείνω ότι είναι σημαντικό να αναφερόμαστε και στην αρχή της επικουρικότητας. Άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα και που αναφέρεται με μεγαλύτερη σαφήνεια στις ε, τροπολογίες είναι ε, το θέμα του fair return προς τις, οργανώσεις, ε, προς αθλητικές οργανώσεις. Δηλαδή, αν το θέμα είναι σε τι βαθμό ε, γίνονται αντικείμενο εμπορική εκμετάλλευση τα αποτελέσματά του. Ε, και πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να βρούμε ε, καλού συμβιβασμού. Έχουμε εδώ πέρα τι τροπολογίε 81, 84, 87 και κάποιε άλλε ενδεχομένω. Πιστεύω ότι θα πρέπει να βρούμε εδώ καλό συμβιβασμό. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι θα πρέπει να έχουν ένα δίκαιο αντίκρισμα οι αθλητικές οργανώσεις. Κατόπιν έχουμε το θέμα του κώδικα δεοντολογίας και πώς θα πρέπει ε, να ε, τον χειριστούμε. Θα πρότεινα να επιμείνουμε ο κώδικας δεοντολογίας να είναι αποκλειστικά συμπληρωματικό μέσο και όχι υποκατάστατο πιο ε, ε, αυστηρών σαφών νομοθετικών μέτρων. Ε, και εδώ θα ήθελα σχετική τροπολογία. Επίσης υπάρχει συζήτηση σχετικά με το σε τι βαθμό τα τυχερά παιχνίδια σε απευθείας σύνδεση οδηγούν σε μεγαλύτερα ρίσκα από ότι ε, τα, τα, τα μη επιγραμμικά. Υπάρχει μια τροπολογία που διαγράφει κάποιες από τις παρατηρήσεις μου ότι υπάρχει ε, αυξημένος κίνδυνος εθισμού ε, στα επιγραμμικά παιχνίδια λόγω της ε, πιο εύκολης πρόσβασης. Για μένα είναι σημαντικό να αναφέρουμε, διότι υπάρχουν αποδείξεις ότι η πιο εύκολη πρόσβαση στα επιγραμμικά παιχνίδια οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο εθισμού. Όχι όλων των παικτών. Υπάρχει όμως ε, αυξημένος εθισμός ε, και ε, αυτό έχει αποδειχθεί και σε διάφορες υποθέσεις μεταξύ άλλων στην πατρίδα μου. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35 είναι κάποιες από τις τροπολογίες που αναφέρονται στο θέμα αυτό. Δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο, απλά ήθελα να αναφέρω ότι υπάρχουν κάποια θέματα, κάποιες ε, κατηγορίες τροπολογιών, όπου νομίζω ότι είναι δυνατόν να πετύχουμε πολύ καλές συμβαστικές προτάσεις. Ε, θα σας υποβάλω σχετικές προτάσεις. Θα συγκαλέσουμε, δεν νομίζω ότι έχει ήδη συγκληθεί, αλλά την επόμενη εβδομάδα θα προσπαθήσουμε να ε, έχουμε μια συνάντηση των σκιωδών εισηγητών στις, την Πέμπτη Τετάρτη, συγγνώμη, 28 Ιανουαρίου στις 11 η ώρα, όπου θα μπορούμε ε, να εξετάσουμε τις τροπολογίες αυτές ε, ενδελεχέστερα. Κατόπιν προτείνεται να ψηφίσουμε εδώ στην Επιτροπή στις 11 Φεβρουαρίου και η έκθεση θα ψηφιστεί ε, τον Μάρτιο στην Ολομέλεια, σε κάποια από τις Ολομέλειες του Μαρτίου. Πάντως είναι καλές οι τροπολογίες. Σας ευχαριστώ για το μεγάλο ενδιαφέρον και είμαι απολύτως πεπισμένη ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλές συμβαστικές τροπολογίες. Ευχαριστώ προς το παρόν. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη σκιώδη εισηγήτρια, την κυρία Κορόλα καταρχήν. Ευχαριστώ, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, λέει η ίδια. Ευχαριστώ για το σχέδιο έκθεσης και τις τροπολογίες. Στην τελευταία συνάντηση με το ΕΛΚ είδα ότι η πλειοψηφία των συναδέλφων μου υποστηρίζουν τις τροπολογίες που κατέθεσα. Είμαι πολύ αισιόδοξη για μια πιθανή συμφωνία μεταξύ εισηγήτριας και σκιώδους εισηγήτριας για σε όλα τα θέματα. Θα μιλήσω καταρχήν για τα γενικότερα θέματα που η κυρία Γόιλε και η πλειοψηφία των συναδέλφων μου συμφωνούν για, την, ε, για τα επιγραμμικά στοιχήματα. Ε, είναι μια οικονομική δραστηριότητα πολύ ιδιαίτερης φύσης σε έναν πολύ ευαίσθητο τομέα όπως ήδη προαναφέρθηκε. Η πάγια νομολογία του ΕΛΚ έτσι έχει του 10 έτσι έχει κρίνει. Γι' αυτό και το Κοινοβούλιο έχει εξαιρέσει την τα επιγραμμικά στοιχήματα και παίγνια από μια σειρά άλλων οδηγιών για το ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Η... Η επόμενη υπόθεση που θα δικάσει το δικαστήριο αφορά τα αφορά το γεγονός ότι οι κανόνες για τα επιγραμμικά στοιχήματα και παίγνια δεν ε, εμπίπτουν στο πεδίο της γενικής νομοθεσίας. Βεβαίως έχουμε την εσωτερική αγορά, την απελευθέρωση των διαφόρων δραστηριοτήτων και αυτά τα δύο πρέπει να συμβιβαστούν. Δεύτερον, συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν τις τάσεις των παιγνίων γενικά και των επιγραμμικών παιγνίων ειδικότερα θέτουν κινδύνους ε, στα άτομα, στις οικογένειες και, και στην κοινωνία γενικότερα. Ε, εγώ στις τροπολογίες μου δεν, ε, μελετώντας για τις τροπολογίες μου δεν βρήκα καμία επιστημονική μελέτη που να έρχεται σε αντίθεση με τα επιχειρήματα του ειδικού μας, του κυρίου Άνταμς, ο οποίος μελέτησε τους κινδύνους που συνδέονται με τα επιγραμμικά παίγνια. Όπως εξηγώ στην έκθεση, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Μελέτη είναι μερολεπτική και περιλαμβάνει πάρα πολλά σφάλματα και ανεπαρκή τεκμηρίωση σε σχέση με την έρευνα και τη μεθοδολογία και δεν μπορεί να χρησιμεύσει λοιπόν ως βάση για τη διαμόρφωση πολιτικής. Τρίτον, τέλος, συμφωνώ με την εισηγήτρια ότι η απλή αυτορύθμιση σε μια τόσο ευαίσθητα τομέα όπως τα στοιχήματα δεν μπορεί να υποκαταστήσει την νομοθεσία έχει προταθεί σε παλαιότερες ε, συζητήσεις της Επιτροπής ε, ε, μάλλον έχει επισημανθεί ότι είναι μια άγνωστη ζώνη, μια ζώνη όπου επικρατεί λίγο ανομία και ότι το να ρυθμιστεί κάπως αυτή η ζώνη θα συνεπάγεται μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών. ορισμένες μορφές επιγραμμικών παιγνίων και στοιχημάτων υπόκειται σε αυστηρότερη νομοθεσία σε πολλά κράτη-μέλη από αυτό που βλέπουμε στους ε, γενικούς κώδικες δεοντολογίας, στους κώδικες αυτορύθμισης, τους οποίους εκδίδουν οι ίδιες οι εταιρείες ε, ε, στοιχημάτων και παιγνίων. Ah, Μια και λείπει ο επόμενο ομιλητή που είχε ζητήσει το λόγο, δίνω το λόγο στην κυρία Ρούλε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια καθώς και την κυρία Κορόλα για την εξαιρετική της ε, συνεργασία. Όπως ε, είπε ήδη η εισηγήτρια, πιστεύω ότι θα είναι δυνατόν να καταλήξουμε σε συμβιβαστικές τροπολογίες έτσι ώστε να υπάρξει μια σωστή απόφαση συμβιβασμού μεταξύ δύο διαφορετικών ε, κατευθύνσεων. Η συγγήτρια δούλεψε πάνω σε μια πολύ συγκεκριμένη βάση. Υπάρχουν τροπολογίες που κινούνται σε αντίθετη κατεύθυνση, αλλά πιστεύω ότι μπορούν να επιτευχθούν ε, σωστές συμβιβαστικές τροπολογίες. Ωραία, η Μπριγκίτε. Εγώ δεν ήθελα να πάρω το λόγο, αλλά αφού δεν είναι εδώ η σκιά μου σε εισαγωγικά, να πω ότι έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες κι εγώ και ελπίζω η Επιτροπή να τις εγκρίνει. Δεν είμαι και πολύ βέβαιη όμως. από τις τροπολογίες μου θα δείτε ότι εγώ δεν συμφωνώ ότι ο τομέας υπάγεται στο πλαίσιο της επικουρικότητας, αλλά αφού υπάρχει πλειοψηφία στην υπόλοιπη επιτροπή, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Ποιος ξέρει, ίσως εγώ να είμαι αυτή που θα κερδίσει την επόμενη μάχη. αυτό θα έλεγε και η σκιώδης ε, συνάδελφός μου, οπότε τα λέω κι εγώ. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Χάρμπορ. νομίζω ότι και οι δικές μου τροπολογίες και των άλλων έτυχαν ευνοϊκής αποδοχής. Ας, πούμε, ας απαντήσουμε σε μερικές από τις ανησυχίες που εκφράσατε. Κάποια από τα σημεία που αναφέρατε δεν είναι τεκμηριώνονται από την έρευνα, όπως το είπατε και εσείς εξάλλου. Και είχαμε και μια πολύ ένθερμη συζήτηση πάνω σε αυτό με τους συναδέλφους. Υπάρχει μια ουσιώδης μειονότητα η οποία υιοθετεί μια πιο ρεαλιστική προσέγγιση, την οποία υποστηρίζω κι εγώ. Η αγορά εξελίσσεται και είναι πολύ ευμετάβλητη και αλλάζει ταχύτατα. Νομίζω ότι πολλές φορές αγνοούμε τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα. Και δεν θέλω να στρουφτοκαμιλίζουμε έτσι και να, να μην βλέπουμε ότι η κατάσταση δεν είναι ικανοποιητική. Νομίζω ότι πιο βαθιά πρέπει να μπούμε και να δούμε ε, την ε, διαθεσιμότητα επιγραμμικών παιγνίων, ε, πόσο εύκολα μπορούν αυτά να αναπτυχθούν στο διαδίκτυο και να υπάρχουν εκεί διαθέσιμα προς όλους πολύ φοβάμαι ότι οι σχετικοί φορείς δεν ανταποκρίνονται με ευθύνη στα σχετικά προβλήματα και νομίζω ότι καταρχήν πρέπει να ενθαρρύνουμε τους παρόχους και τους υπεύθυνου διαχειριστές αυτών των παιχνίων να λειτουργούν πιο υπεύθυνα και οι ανεύθυνοι να τεθούν εκτός αγοράς. Υπάρχουν θέματα τα οποία <laughs> μοιάζουν να προσποιούνται ότι όχι δεν, υπάρχει τέτοιο, δεν υπάρχουν τα επιγραμμικά παίγνια και στοιχήματα. Ε, ιδίω τα κρατικά λαχεία, τα οποία σε μερικές περιπτώσεις κάνουν πολύ καλή δουλειά και χρηματοδοτούν ε, τα, την αθλητική δραστηριότητα κτλ. Εγώ μέχρι στιγμή ε, δεν βλέπω να απειλούνται αυτά τα λαχεία από τα επιγραμμικά παίγνια και στοιχήματα. Πολλά μάλιστα από αυτά τα κρατικά λαχεία μπαίνουν και αυτά στο διαδίκτυο και αναπτύσσουν και αυτά επιγραμμικές δραστηριότητες. Πολλά μάλιστα από τα επιγραμμικά παίγνια και στοιχήματα που αναπτύσσονται. Μπορεί να είναι και πιο υγιείς επιχειρήσεις από τα κρατικά λαχεία. Ε, βέβαια υπάρχει πρόβλημα. Ε, μάλλον πρέπει να γίνει διάκριση ανάλογα με το αν ε, συμμετέχεις στα ιδιωτικά παίγνια και στοιχήματα ή αν συμμετέχεις στα κρατικά και δημόσια επιδοτούμενα παίγνια και στοιχήματα. Είναι διαφορετικά αυτά τα δύο. Ε, αυτό δεν, ε, εγώ δεν είμαι μεροληπτό υπέρ του ενός ή του άλλου. Ε, απλά υπάρχει μια αίσθηση ότι το δικαστήριο στις σχετικές υποθέσεις προσπαθεί να καθοδηγήσει, να χειραγωγήσει τους μάρτυρες και να κρίνει κατά αντίθεση των απόψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπα και όπως είπαμε, δεν υπάρχει αρκετή και αξιόπιστη επιστημονική έρευνα και πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω λοιπόν δύο διαφορετικές ομάδες ε, ε, τροπολογιών. Καταρχήν, πρέπει να είμαστε πολύ πιο ρεαλιστές και να αρχίσουμε να επιλύουμε μερικά από τα προβλήματα. Η ανάπτυξη παιγνίων και στοιχημάτων επιγραμμικά και σε πραγματικό χρόνο αρχίζει να καθίσταται πολύ δημοφιλής σε ορισμένες ομάδες πολιτών οι οποίοι θέλουν να συμμετέχουν, θέλουν να παίζουν. Αλλά ανοίγει δυνάμει, ε, ανοίγει περιθώριο για πολλά θέματα χειραγώγησης και ακεραιότητας ο Χάρη σίγουρα θα μπορούσε να απαντήσει μερικά από αυτά τα θέματα που ανέκυψαν και κατά τη δημόσια ακρόαση για την ε, έλλειψη συνεισφοράς. Υπάρχουν πολλά επιγραμμικά παίγνια και στοιχήματα τα οποία ενώ υποτίθεται ότι εκτιλήσονται για να συνεισφέρουν οικονομικά στην ανάπτυξη του αθλητισμού, στην ουσία δεν το κάνουν. Θυμάμαι μάλιστα και μια περίπτωση μια ενός επιγραμμικού παιγνίου ε, σε αγώνες ε, δρόμου, ε, υποδρομίες, συγγνώμη. Και Υπάρχει ένα κοινό, ξέρετε, υπάρχει ένα κοινό που συμμετέχει πάρα πολύ ενεργητικά στις υποδρομίες και στις ηλεκτρονικές υποδρομίες και πρέπει να το δούμε. Και εκείνη και η, διαφορά και η δυσκολία σε σχέση με άλλες ομάδες παιγνίων και στοιχημάτων. Όπως είπα όμως υπάρχουν δύο ξεχωριστές απόψεις πάνω σε αυτό. Εν μέρη, ίσως αν θέλετε, ότι Υπάρχει γενικώ μια τάση αγιοποίησης των κρατικών λαχείων και κρατικών παιγνίων και αυτές οι επιχειρήσεις εισαγωγικά οι κρατικές πρέπει επίσης να υπάγονται σε έλεγχο και δεν μπορεί να τους επιτρέπεται ανεξέλεγκτα να κάνουν ό,τι θέλουν μόνο και μόνο επειδή έχουν μια καλή φήμη πίσω τους και ένα κύρος. Ε, όσοι από εμά ε, θέλουμε να υιοθετήσουμε μια πιο ρεαλιστική άποψη, μπορεί να υποβάλουμε μια έκθεση μειοψηφία. Όπω ξέρετε, μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και ξέρετε ότι κάθε φορά που υποβάλλεται μια έκθεση πλειοψηφία, μπορεί κανεί να υποβάλει και μια έκθεση μειοψηφία. Νομίζω ότι αυτό θα αντανακλά καλύτερα τι απόψει του Κοινοβουλίου και θα, τουλάχιστον για τα θέματα που άπτονται του δημόσιου τομέα και θα δείξει και στο κοινό ότι υπάρχουν και άλλε απόψεις. Ίσως λοιπόν θα μπορούσαμε να αναλάβουμε μία έκθεση ίδιας πρωτοβουλία. Δεν ξέρω τι λένε. Ε, δεν το εννοούμε αυτό ως μια εχθρική πράξη προς την πλειοψηφία. Απλώς θέλουμε το κοινό έξω να ξέρει τι κάνουμε και να ξέρει τι απόψεις υπάρχουν για τα θέματα αυτά. Ε, νομίζω ότι είναι μια πιο όρημη άποψη αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που και η Γαλλική Προεδρία εργάστηκε πάνω σε αυτό και εγγενίασε κάποιες διαδικασίες. Ε, ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε κάποια στιγμή στο μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Χάρμπο. κύριο Χάρι, παρακαλώ. Νιώθω λίγο σαν τον Πίτερ Παν. Νιώθω πολύ μακριά από τον σκιώδη εισηγητή μου. Αντίθετα με την προλαλή σας που νιώθει πολύ καλά με την σκιώδη εισηγήτριά σας. Τέλο πάντων δεν κατάφερα να, συμμετάχω, να συμμετάσχω στη συνάντηση την περασμένη φορά. Ε, έμαθα όμως και ενημερώθηκα για το ποιος υποστηρίζει τι. Αποφάσισα επειδή υπάρχει ένα πρόβλημα με τις ακαδημαϊκές μελέτες στον τόμο αυτό, να, μιλή, να σας διαβάσω δύο παραγράφους από την μελέτη που ανατέθηκε από τη δική μας Επιτροπή. Λέει λοιπόν, αυτό το απόσπασμα ίσως θα μας δείξει τη σωστή κατεύθυνση. Σημείο 7. Θα διαβάσω δύο από την περίληψη, δύο όρους από την περίληψη και ένα από το κύριο Σώμα. Σημείο 7. Σε σχέση με τα τυχήματα και τα παίγνια. Καταφέραμε να κάνουμε μια απλή σύγκριση μεταξύ τη Σουηδία που έχει ένα κρατικό μονοπωλίο παιχνίδων και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχει απελευθερωμένη αγορά. Ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι ε, το ίδιο πράγματα ισχύουν πάνω κάτω και στι δύο ένομε τάξει. Και έτσι μπορεί κανεί να καταλήξει ότι η οργανωτική δομή, η κρατική οργανωτική δομή παιχνίων και στοιχημάτων δεν παίζει αποφασιστικό ρόλο. Σημείο 8. Υπάρχουν λίγα επιστημονικά στοιχεία που δείχνουν ότι εξαπατούνται οι συμμετέχοντας σε επιγραμμικά παίγνια και στοιχήματα στους ιστότοπους εκτός και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πολύ φοβάμαι ότι υπάρχει μεγάλη παραπληροφόρηση και ατεκμηρίωτες απόψεις που κυκλοφορούν. Σημείο 2-3-5 στο κύριο σώμα της ε, έκθεσης και διαβάζω. Ο κύριο Μπέρμανς από το Σύλλογο Ευρωπαϊκών Καζίνο μας είπε ότι υπάρχουν 2.600 παράνομα δικτυακά κέντρα παιχνίων και στοιχημάτων στον κόσμο και τα χρήματα που διέρχονται μέσω αυτών των ιστότοπων ε, αφορούν βασικά πλήσιμο βρώμικου χρήματος. Η ακαδημιακή μελέτη που προαναφέρθηκε εκτιμά ότι υπάρχουν μόνο 2.069 επιγραμμικοί ιστότοποι παιχνίων και στοιχημάτων και δεν είναι όλοι απολύτως νόμιμοι. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά επιχειρήματα. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει κάποια ειλικρίνεια στη συζήτηση και να μιλούμε με στοιχεία και γεγονότα ε, πάνω στα οποία θα μπορούμε να συμφωνούμε γιατί στην Επιτροπή αυτή πάντοτε κοιτάμε τις μελέτες και τις χρησιμοποιούμε ως βάση της συζήτησής μας. Χρειάζεται κάποια μια εντιμότητα. Εγώ καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν πολύ διαφορετικές απόψεις για, το επιγραμμικά, για τα επιγραμμικά στοιχήματα και καταλαβαίνω τι προβλήματα μπορούν να προέλθουν. Προέρχομαι από το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουμε ένα πολύ φιλελεύθερο και ανοιχτό σύστημα επιγραμμικών παιχνίων και στοιχημάτων ε, με, προσ... με ιδιωτικούς κώδικες δεοντολογίας και τελικά από τις μελέτες φαίνεται ότι τα ίδια προβλήματα έχουμε εμείς με τη Σουηδία που υπάρχει κρατικό και μονοπόλιο στοιχημάτων. Νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα εδώ να υποβληθεί μια έκθεση μειοψηφία. Γιατί δεν νομίζω ότι δεν βλέπω να συγκλίνουν αυτέ οι απόψει στο εγγύ μέλλον. Επίση, για το θέμα τη ακαιρεότητα και του δίκαιου πεδίου. Βλέπω το επιχείρημα, το καταλαβαίνω και σίγουρα θα μπορούσε να υιοθετήσει θετηθεί κάτι που να καθησυχάζει ε, τον κόσμο ότι δεν υπάρχουν περίεργες σχέσεις μεταξύ των επιγραμμικών στοιχείων και παιχνίων και του επίσημου αθλητισμού των αθλημάτων. Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που, και ομάδες που έρχονται και μας ζητούν να υποβάλουμε συγκεκριμένες ε, τροπολογίες. Για παράδειγμα κυβερνητικοί φορείς οι οποίοι δεν θέλουν να ασχοληθούν ιδιαίτερα. Τους ενδιαφέρει απλά να ενισχύσουν ε, τη βάση του αθλητισμού και δεν τους ενδιαφέρουν τα θέματα της ακαιρεότητας. Εγώ νομίζω ότι οι πόροι αυτοί ε, πρέπει να, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι πόροι πραγματικά πηγαίνουν εκεί που θέλουμε σε αυτή την Επιτροπή να πηγαίνουν. Ναι, μας θυμίζετε το Πίτερ Παν, το αγοράκι που δεν ήθελε να μεγαλώσει. Ο κύριος Τουμπό. Και πολύ γρήγορα θα πρέπει να περάσουμε και στην επόμενη έκθεση, τα σχολεία που σχετί. Ναι, πολύ γρήγορα. Εδώ και πολλά χρόνια παρακολουθώ την υπόθεση αυτή. Και νομίζω ότι μπορεί κάποιος με ασφάλεια να καταλήξει στο εξή συμπέρασμα. Ότι δηλαδή τα επιγραμμικά παίγνια, η ύπαρξή τους η ίδια, αναμφισβήτητα προκαλεί και εγείρει νέα ζητήματα. Πρέπει να μην σκεφτόμαστε απλοϊκά. Σαν να ήταν τελείω ουδέτερη αυτή η τεχνολογία, η εξέλιξη τεχνολογική. Σαν να επρόκειτο για ένα τελείως διαφανές μέσο. Γι' αυτό ακριβώς οι ιδέες που απαριθμούνται στην έκθεση της κυρίας Αντεμόζε, οι κίνδυνοι οι προφυλάξεις καθώς και τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για σκοπούς προφύλαξης για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους, όλα αυτά μου φαίνεται ότι τα αποκρίνονται πραγματικά στις ε, επιδράσεις που μπορεί να έχει, στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει το διαδίκτυο και η χρήση του, στο πώς παίζονται τελικά τα παιχνίδια σε κάθε περίπτωση οι σωματικές ασκήσεις, τα παιχνίδια τα ίδια, είναι δραστηριότητες που ελέγχονται αυστηρότατα σε όλα τα κρατη και παρακολουθούνται μεταξύ άλλων και για σκοπούς φορολογικούς. Εάν λοιπόν τα νέα τεχνολογικά μέσα έχουν αυτό το στιγμιαίο, τον άμεσο χαρακτήρα και επιπλέον παρουσιάζουν και αυτούς τους πρόσθετους κινδύνους, αυτό μάλλον σημαίνει ότι χρειαζόμαστε αυστηρότερα προφυλακτικά μέτρα για τα επιγραμμικά παιχνίδια ακριβώς. Άλλωστε, είτε είναι δημόσιοι φορεί είτε ιδιωτικοί αυτοί που τα χειρίζονται, νομίζω ότι θα πρέπει να έχουμε την ίδια στάση. Αυτό ω προ το γενικό μα προσανατολισμό. Θα κατέληγα ότι δεν νομίζω, όπω ο Μάλκομ και ο Κρίς, ότι η οικονομία των τυχερών παιγνίων είναι μια οικονομία υγιής. Όταν μιλάμε για ιστότοπους νομίμους, νόμιμους μάλλον, αυτό μπορεί και να ισχύει, αλλά δεν μπορούμε να διεξάγουμε από το γεγονός ότι η οικονομία αυτή λειτουργεί εύρωστα, να καταλήξουμε από αυτό στο ότι στη σχέση με τον παίκτη δεν συμπεριλαμβάνονται και κάποιοι κίνδυνοι, κίνδυνοι οικονομικού χαρακτήρα, που εξορισμού είναι και ανθρώπινοι και κίνδυνοι υγείας και εξαπάτησης και ούτω καθεξής. Γι' αυτό ακριβώς νομίζω σωστό είναι να, προτείνουμε, να προτείνουμε να ληφθεί μια σειρά από μέτρα. Πρέπει να καταπολεμήσουμε κάθε είδους παρατυπία και ατασταλία εξορισμού, τα τυχερά παίγνια τα επιγραμμικά είναι πιο επικίνδυνα. Και για τα παίγνια που θα εγκριθούν και από νομική σκοπιά, εκεί θα πρέπει να λάβουμε πολύ συγκεκριμένα μέτρα. Το βρίσκω λοιπόν βάσιμο το να θέλουμε τέτοια μέτρα. Όσο και αν λειτουργεί το οικονομικό αυτό σύστημα που έχει δημιουργηθεί, όπως είπε και ο Μάλκομ. Και η τρίτη μου παρατήρηση Αποφεύγοντα να σχολιάσω τι τροπολογίε που υπέβαλα, η κυρία Κορχόλα είπε πολύ σωστά ότι προσπαθούμε να καταλήξουμε και σε κάποιες κοινέ συνανετικές τροπολογίες. Εδώ λοιπόν ήθελα να επιμείνω στην αθλητική διάσταση. Όταν ο κύριος Μάντερς είχε ετοιμάσει την έκθεση για τον αθλητισμό στην Ευρώπη είχαμε επισημάνει ότι είναι σημαντικό το στίχημα, το παίγνιο να έχει καθοριστική επίδραση στην ακαιρεότητα, τον ακαιρό χαρακτήρα των ε, διαφόρων ε, αθλητικών συναντήσεων. Άρα πρέπει να ληφθούν και κάποια μέτρα προφύλαξης. Τώρα, όταν ο Κρίς λέει ότι πρέπει να συμμετέχουν ε, τα νομικά συστήματα και οι νομικώ συγκεκριμένε επιχειρήσεις στο ΣΥΚ στο, που έχουν τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο στην χρηματοδότηση των αθλητικών διοργανώσεων, αυτό ίσω είναι μια ιδέα. Ο γαλλικό νόμο που ανέφερε και ο Μάλκομ, ο νέο γαλλικό νόμο που πρόκειται να αρχίσει να συζητάται στο Γαλλικό Κοινοβούλιο σύντομα, θα περιλαμβάνει ένα ολόκληρο κεφάλαιο όπου θα εξετάζει το πώ οι επιχειρήσει, οι ιδιωτικέ επιχειρήσει που έχουν έγκριση να παρέχουν την υπηρεσία των, ε, των τυχερών παιχνίων θα μπορούσαν να χρηματοδοτούν και τα άλογα στον υπόδρομο και άλλες αθλητικές δραστηριότητες. Νομίζω λοιπόν στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης <clears throat> και θα έπρεπε και στόχος ακριβώς της έκθεσης να είναι κάποιες, κάποια μέτρα προφύλαξης μέτρα προφύλαξη που πρέπει να προγραμματιστούν ώστε τα παίγνια να μην επηρεάζουν τη διοργάνωση, την διενέργεια και το αποτέλεσμα αθλητικών διοργανώσεων. Thank you. Ευχαριστώ. Κυρία Σαλντεμόζα, έχετε σχόλια. Uh, uh, ναι, έχω κάποιες παρατηρήσεις, δεν θα μακρηγορήσω. Να πω καταρχήν ότι δεν θα θεωρήσω καθόλου ε, εχθρική ενέργεια το να υποβάλλετε έκθεση της μειοψηφία. Έχετε κάθε δικαίωμα να το κάνετε αυτό. Θεωρώ όμως ότι θα μπορούσατε να περιμένετε μέχρι να δούμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας στην Επιτροπή μας. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό σαν έκφραση του ότι θεμελιωδώς διαφωνούμε πολιτικά για το τι πρέπει να γίνει στον τομέα αυτόν και γι' αυτό είμαστε άλλωστε εδώ πέρα. Είναι η δουλειά μας και έχουμε κάθε δικαίωμα να διαφωνούμε. Ένα πράγμα θέλω να πω όμως τώρα, διότι, διότι υπάρχει κάτι που με εκνευρίζει επανειλημμένα. Επειδή διαφωνούμε πολιτικά, θυμώνω όταν υπονοείτε ότι επειδή δεν συμφωνώ μαζί σας ε, ότι δεν έχω την παραμικρή ιδέα τι συμβαίνει στον τομέα αυτών. Υπάρχουν στοιχεία. Αλλά παραδεχόμαστε όλοι ότι υπάρχει και έλλειψη στοιχείων σε πολλούς τομείς. Ζητάμε στην έκθεση να έχουμε καλύτερα στοιχεία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Αλλά θυμώνω όταν υπονοείτε ότι δεν γνωρίζω αρκετά για το θέμα και ότι γι' αυτό το, έχουμε το αποτέλεσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή αλλά μια πολιτική και δίκαιη διαφωνία στο θέμα αυτό ε, δεν είναι κανένα πρόβλημα. Προτείνω να συναντηθούμε και να δούμε πώς μπορούμε να φτάσουμε σε συμβαστικές τροπολογίες τουλάχιστον σε κάποια θέματα. Νομίζω ότι θα είναι δυνατό αυτό για να μπορέσουμε έτσι να καταλήξουμε σε στήριξη της πλειοψηφίας στην έκθεση αυτή συμπέρασμα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένα έξω από το Κοινοβούλιο που θα αμφιβάλλει ότι υπάρχει μεγάλη πολιτική διαφωνία προ τα που θα πρέπει να κινηθεί το θέμα, άσχετα από το αν υπάρχει έκθεση ε, της μειοψηφίας ή όχι. Νομίζω ότι ο, ο κόσμος έξω γνωρίζει ότι, υπάρχει, ότι υπάρχουν σημαντικές πολιτικές διαφωνίες γιατί θα πρέπει να γίνει στον τομέα αυτών. Πρόεδρος, ευχαριστώ κυρία Σάντε Μόζε. Η ψηφοφορία στην ΙΜΚΟ θα γίνει, όπως είπα, στις 11 Φεβρουαρίου και στην Ολομέλεια θα ψηφιστεί τον Μάρτιο. Το επόμενο θέμα είναι η έκθεση του κυρίου Καμάλ για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Παρακαλώ κύριε Καμάλ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ λοιπόν. Εξετάζοντας τον τομέα αυτόν, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να υπάρξει συνέχεια του προηγούμενου κανονισμού στον τρόπο που θα εξετάσουμε το θέμα. Σε κάθε περίπτωση το χρονικό διάστημα για να συντάξουμε την γνωμοδότηση ήταν πολύ σύντομο. Θα συμφωνούν και οι σεώδεις συζητητές ότι είχαμε μεγάλη χρονική πίεση. Αυτό που θέλαμε όμως είναι να έχουμε σαφώς λεπτομερή συζήτηση και μετά την ψηφοφορία. Δεν θέλω να μονοπολίσω τη συζήτηση λοιπόν για την έκθεση αυτή, αλλά πριν περάσω στις λεπτομέρειε α προσπαθήσουμε να δούμε το γενικότερο πλαίσιο μέσα στο οποίο χρειάστηκε να συντάξουμε την έκθεση αυτή. Θεωρούμε ότι τα κινητά τηλέφωνα είναι μια ιστορία επιτυχία για την ε, ευρωπαϊκή οικονομία. Οι τιμέ έχουν μειωθεί και αν κάνουμε κάποιε συγκρίσει με άλλου βιομηχανικού τομεί, οι τιμέ των κινητών έχουν περικοπεί πολύ περισσότερο από τι άλλε σε άλλους βιομηχανικούς κλάδους. Οι τιμές παρά τις αξιώσεις δεν ξέρω κατά πόσον ε, απαιτούν παρέμβαση. Πάντως υπάρχουν βιομηχανίες, προϊόντα, όπου όταν υπάρχουν καινοτόμες εξελίξεις, η τιμή στην αρχή είναι πολύ υψηλή και σιγά σιγά μειώνεται. Νομίζω λοιπόν ότι είναι προ όφελο μια εταιρεία, των εταιρεών γενικών, να διατηρήσουν υψηλά τι τιμέ αλλά να υπάρχει και μεγάλος αριθμός χρηστών. Ο τομέας όμως αυτός δεν αποτελεί ακόμα πηγή για τις κυβερνήσεις, πηγή που να τους δίνει τρόπο να λάβουν ε, ένα μέρος των ε, φόρων των φορολογουμένων, των φόρων που καταβάλουν φορολογουμένων. Αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Και κάποια τεχνικά σημεία τεχνικές λεπτομέρειες, νομίζω κάποιες από τις ομάδες ζήτησαν ε, αναβολή της ψηφοφορίας. Νομίζω ήδη προαναγγέλθηκε αυτό στην αρχή της συνεδρίασης, ενώ δεν ήμουν εδώ. Θα συμφωνήσω όμως, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες συζητήσεις και με τους σκεώδεις εισηγητές. Τώρα, τι προσπάθησα εγώ να κάνω, να προκαλέσω διάλογο για το θέμα αυτό. Γι' αυτό ακριβώς απορρίψαμε τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον περιορισμό τα ανώτατα όρια των τιμών, καθώς και την διεύρυνση του κανονισμού για τις φωνητικές υπηρεσίες. Επίσης, συζητήσαμε με την Επιτροπή Ήτρε και είδαμε κατά πόσο μπορούμε να επικεντρωθούμε στα ζητήματα προστασία των καταναλωτών και την διαφανή χρήση. Εμείς, διότι εκείνοι θέλουν να επικεντρωθούν σε ό,τι αφορά τη δική τους αρμοδιότητα κατά κύριο λόγο. Σε κάθε επεξηγηματικό σημείωμα έχει κανείς περιορισμένο αριθμό χαρακτήρων που μπορεί να χρησιμοποιήσει. Γι' αυτό έχω επισυνάψει ένα επεξηγηματικό έγγραφο, ένα έγγραφο εργασία στην έκθεση αυτή. Το οποίο θα πρέπει να διαβάσετε για να δείτε λίγο το ιστορικό πλαίσιο της όλης πρότασης. Νομίζω ένα από τα επικριτικά σχόλια που άκουσα από όλε τι πολιτικέ πρατάξει είναι ότι δεν σκεφτήκαμε αρκετά τον αντίκτυπο που είχε ο προηγούμενο κανονισμό. Έχουμε αρκετά δεδομένα, είχαμε αρκετό χρόνο στη διάθεσή μα. Γιατί περνάμε στο roaming 2, ενώ ήδη δεν έχουμε καταμετρήσει τον αντίκτυπο τη περιαγωγή 1. Εάν δείτε τα δεδομένα και τα στοιχεία που έχουμε και προσπαθήσετε να τα αναλύσετε, θα καταλήξετε σε ένα ερώτημα. Γιατί προσπαθούμε να ρυθμίσουμε ένα τέτοιο τομέα. Θα μπορούσε να το σκεφτεί αυτό, καν... να το σκεφτεί αυτό κανείς και για άλλους τομείς. Αν δείτε τώρα τους αριθμούς ERG, για τις φωνητικές υπηρεσίες και τα στοιχεία που προκύπτουν από την περιαγωγή 1. Δεν υπάρχει αλλαγή στον... Μάλλον υπάρχει αλλαγή στις φωνητικές υπηρεσίες, στον όγκο φωνητικών υπηρεσιών, 15 25%. Όμως το πρώτο τρίμηνο του 2008 θα δει κανεί αύξηση και στα, στον όγκο των SMS και την περιαγωγή SMS, που έχει αυξηθεί περισσότερο από την περιαγωγή τη φωνητική. Άρα τι συμπέρασμα να διεξάγει κανείς από αυτό, ότι χρειαζόμαστε βεβαίως δεδομένα. Αλλά ότι τα δεδομένα μας αυτά είναι αρκετά περιορισμένα. Και θα πρέπει κανείς να σκεφτεί ότι ο όγκος τους τομεί που ρυθμίζουμε αυξάνεται, αλλά λιγότερο από του τομεί που δεν ρυθμίζονται ακόμη. Άρα γιατί να προσπαθούμε να ρυθμίσουμε του τομεί αυτού. Τι προτείνει λοιπόν η Επιτροπή, προτείνει ε, όρια, ανώτατα όρια στις τιμές, στις λιανικές τιμές των SMS, των γραπτών μηνυμάτων. Έχει γίνει όμως μελέτη αντικτύπου στον πρώτο χρόνο υλοποίησης του προηγούμενου κανονισμού. Και ποιες είναι οι εναλλακτικέ μας λύσεις. Φαντάζομαι κάποιοι καταλαβαίνουν ότι είναι προκλητικέ αυτέ οι θέσει, αλλά αυτό είναι θελημένο για να προκαλέσουμε και διάλογο. Και ενδεχομένω να αλλάξει αρκετά και η μορφή τη έκθεση, όπω θα καταλήξει να φύγει από την Επιτροπή μα. Δεν είμαι καθόλου αφέλη. Θέλω να προκαλέσω συγκεκριμένη ε, συζήτηση για συγκεκριμένα ζητήματα του κανονισμού. Τώρα, και στο έγγραφο εργασία περιλαμβάνονται κάποια ερωτήματα, Όπω, είναι η αγορά περιεγωγή μια ξεχωριστή αγορά, Α το σκεφτούμε αυτό σύντομα. Εάν δει κανεί οποιοδήποτε πρότυπο αγορά, ε, μοντέλο αγορά για οποιαδήποτε εταιρεία, θα σκεφτεί, θα δει ότι αυτό που απασχολεί την εταιρεία είναι το κέρδο, το πλεόνασμα. Αλλά επίση ότι πολύ συχνά οι εταιρείε έχουν και προβλήματα με απώλειε που αντιμετωπίζουν. Πολλέ φορέ λοιπόν παίρνουν το πλεόνασμα που έχουν σε κάποιου τομεί, το επιπλέον εισόδημα, για να χρηματοδοτήσουν του τομεί όπου υπάρχει απώλεια. Τώρα, το κομμάτι τη περιαγωγή είναι ένα τομέα όπου υπάρχει κέρδο, αλλά μπορεί διασταυρούμενα να χρηματοδοτηθούν και από το κέρδο αυτό το μέσο που οι, οι εταιρείε προσφέρουν υπηρεσίε στι οποίε έχουν απώλειε. Λίγα κερδίζουν ε, από άλλε υπηρεσίε οι εταιρείε. Και ένα τρόπο να ανακτούν κάποια ποσά είναι μέσω τη συνδρομή των πελατών ή κέρδο από άλλου τομεί, από άλλε υπηρεσίε που προσφέρει η εταιρεία. Εάν δούμε τώρα ξεχωριστά εταιρείε ή μοντέλα στην αγορά, επιχειρήσει και πώ λειτουργούν και απομονώσουμε το κέρδο στον καθένα από του τομεί, θα δούμε το καθαρό κέρδο μεν. Αλλά πρέπει να συνεξετάσουμε σε ποιου κλάδου επανεπενδύει μια εταιρεία τα ποσά αυτά για να καλύψει απώλειες. Φαίνεται τελικά ότι το κέρδος είναι κακιά λέξη. Όμω, εάν δείτε πόσο μέρο του κέρδου αυτού πηγαίνει στι τσέπε των μετόχων μια εταιρεία, θα δείτε ότι είναι πολύ περιορισμένο το ποσοστό αυτό. Αν ε, διαβάσετε τι λέγεται και στι εφημερίδε, αυτό το επιπλέον κέρδο ε, χρηματοδοτεί του φόρου, άλλε υποχρεώσει τη εταιρεία, καθώ και τι επενδύσει για τι νέε τεχνολογίε. Συνεχώ γίνονται επενδύσει για νέα τεχνολογικά μέσα. Και ε, αυτή τη στιγμή οι εταιρείε κοιτάνε ε, τι τεχνολογίε τι λεγόμενε 4D και πολλά άλλα. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία επίση έχει ηγετικό ρόλο στον τομέα αυτό που δεν θέλουμε να τον χάσει. Ποιε είναι οι εναλλακτικέ λύσει λοιπόν που προτείνω. Πρώτον, όχι διεύρυνση του πεδίου με ρήτρα λήξη, σταδιακή μείωση μάλλον, sunset close. Επίσης, εάν προσπαθήσουμε να ορίσουμε τώρα τιμές πριν τις ευρωπαϊκές εκλογές τελικά μήπως έχουμε περισσότερο πολιτικούς υπολογισμούς στο μυαλό μας παρά οικονομικούς ας το αφήσουμε αυτό στα χέρια των ειδικών που συνεργάζονται με τους ε, εμπορευόμενους και τους καταναλωτές απευθείας μήπως τις αποφάσεις αυτές δεν μπορούν να τις λαμβάνουν ρυθμιστές και νομοθέτες Ξέρω βέβαια ότι υπάρχει πρόταση, υπάρχει νομοθετικό πακέτο για να ενδυναμώσουμε το ρόλο των ρυθμιστών εδώ, αλλά απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε από το Συμβούλιο και τώρα ακόμη το συζητούμε. Παρόλα αυτά, ένα άλλο επικριτικό σχόλιο που έλαβα για την πρόταση αυτή είναι το ERD. Τα ERD μάλλον, τα αρμόδια συμβούλια δεν έχουν αποδειχτεί αρκετά ανεξάρτητα. Δεν έχουν ε, υψώσει το ανάστημά του ενώπιον τη επιτροπή. Όμω, εάν αφήσουμε το θέμα στα χέρια των ρυθμιστών για να αποφασίσουν, θα πρέπει να αποδείξουν και την ανεξαρτησία του, να μα πείσουν ότι οι αποφάσει του είναι σωστέ και βασίζονται σε σωστή ανάλυση τη αγορά. Και εξισορροπούν τα συμφέροντα των καταναλωτών και αυτά των επιχειρηματιών. Επίση, μα απασχόλησε και το θέμα μια ρήτρα μη διακριτική μεταχείριση και στο έγγραφο εργασία γίνονται κάποιε σχετικέ προτάσει. Και εάν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν ξεχωριστά μερίδια αγορά ε, όπου όλοι οι πελάτες της περιαγωγής ε, πληρώνουν πολύ ψηλές τιμές και υψηλά τέλη, θα πρέπει τότε να επικεντρωθούμε ακριβώς στα συγκεκριμένα αυτά μερίδια αγορά, συγκεκριμένε εταιρείε και συγκεκριμένε επιχειρήσει. Και αυτέ να αντιμετωπίσουμε. Και μετά πρέπει να δούμε και τι ε, ισοτιμίες. Δηλαδή, θα πρέπει να είμαστε καινοτόμοι, επινιωτικοί να μην περιοριστούμε σε ένα χονδροειδές εργαλείο ανώτατων των ορίων των λιανικών τιμών. Εγώ αυτό που προτείνω είναι ανταλλαγέ. Ανταλλαγέ να μπορεί κανεί λόγω χάρη να αγοράσει ένα σύλλογο δεδομένων. Α σκεφτούμε λοιπόν στη συζήτησή μα, τι εναλλακτικέ λύσεις υπάρχουν. Και αν θέλετε να τι απορρίψετε αυτές τι εναλλακτικέ λύσει, κάντε το τεκμηριωμένα. Ελάτε και υποβάλλετε μου προτάσει ιδέε αιτιολογημένες για το τι, για το λόγο για τον οποίο θεωρείτε ότι οι εναλλακτικέ λύσει δεν είναι εύστοχε. Νομίζω όμω ότι υπάρχουν δύο σημεία στα οποία θα συμφωνήσουμε όλοι, μεταξύ σκιωδών εισηγητών και μου, ότι χρειάζεται διαφάνεια στον τομέα αυτό. Δεν έχει υπάρξει αρκετή διαφάνεια για του πελάτε. Σε μια από τι ακροάσει για την περιαγωγή 2, ένα από του χρήστε είπε, εάν ο πελάτη θέλει ακριβώ την τιμή τη περιαγωγή, να πάει στο διαδίκτυο να δει. Αλλά δεν βρίσκω ότι αυτή είναι σωστή απάντηση. Διότι όταν ο πελάτη καταναλώνει την υπηρεσία, ο χρόνο και ο τόπο που γίνεται η κατανάλωση είναι ακριβώ η στιγμή και ο τόπο που χρειάζεται για το, την πληροφορία. Θα πρέπει λοιπόν να ενδυναμώσουμε τον, τη διάσταση τη διαφάνεια. Εδώ δεν έχω συμπεριλάβει καμία ιδέα, γιατί ξέρω ότι οι σκιώδει συζητητέ το έχουν αναλάβει αυτό και του έχει απασχολήσει. Άρα επαφίαμε στι θετικέ του τροπολογίε για να ενισχύσουν το, τη διάσταση τη διαφάνεια. Θα το συζητήσουμε λοιπόν μεταξύ των ομάδων. Και κάτι άλλο που μα απασχολεί είναι ότι γίνεται και με του μικρού τους εμπορευόμενους, δηλαδή μικρές εταιρείες που πρέπει να ανταγωνιστούν μεγάλες εταιρείες με πολύ ευνοϊκούς όρους στην αγορά. Επίσης αυτοί οι μικροί εμπορευόμενοι μπορεί να είναι μικροί στη συνολική ευρωπαϊκή πραγματικότητα, αλλά μπορεί να έχουν μεγάλη σημασία για την εσωτερική τους, την εγχώρια αγορά. Και μπορεί να είναι και σημαντικό το εισόδημα που φέρνουν στην εσωτερική αυτή αγορά. Θα παραμείνω σε αυτά και ελπίζω να έχω προκαλέσει αρκετά θέματα για συζήτηση. Περιμένω και την τοποθέτηση των σχεδόν εισηγητών. Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα τους σκιώδεις εισηγητές. Ο κύριος Μπουφών, δεν ξέρω αν το προφέρω σωστά. Κατάλαβα ότι υπάρχει ανάγκη να εφαρμόσουμε ρυθμιστικά μέτρα και υπάρχει μια σειρά οργανώσεων καταναλωτών αλλά και μια σειρά δικαιολογημένων ε, αξιώσεων ε, Ευρωπαίων χρηστών. Κάποιες στιγμές είχαμε δραματικά γεγονότα, με άλλα λόγια δραματικούς λογαριασμούς. Ε, βρέθηκαν προ σημαντικών εκπλήξεων οι καταναλωτές. Το πλήθος των παραπώνων των καταναλωτών οδηγεί στην ανάγκη να συζητήσουμε ανοιχτά το θέμα. Και όπως είπε ήδη ο κύριος Καμάλ, μου φαίνεται και εμένα πολύ σημαντικό να προωθήσουμε μέτρα διαφάνειας ώστε ο πελάτης κατά την περιαγωγή δεδομένων να έχει τις σχετικές πληροφορίες και να μπορεί να αποφασίσει εάν θέλει να συνεχίσει να υποφελείται από την υπηρεσία αυτή. Όταν μιλάμε για πλαφόν τιμών, Συχνά τα πλαφόν αυτά δεν δικαιολογούνται με, την, ε, με τις δαπάνες στον, ε, στον χοντρικό κρίκο της αλυσίδας. Ε, μας ενδιαφέρει το τι τελικά θα πληρώσει ο καταναλωτής. Προσπάθησα να βρω την αιτιολόγηση για τη διαμόρφωση των τιμών. δεν καταλαβαίνω γιατί εντός της Ευρώπης, εντός ενός κράτους μέλους ε, διαφέρουν τόσο πολύ μεταξύ τους οι τιμές ε, περιαγωγής, ε, καθότι συνήθω αιτιολογούνται οι τιμές αυτές με τις δαπάνε για τα πιστοποιητικά λειτουργία των επιχειρήσεων. Θα ήταν λογικό λοιπόν να εφαρμόσουμε σχετικό μέσο. σε πολλές ε, συνομιλίες μου με καταναλωτές, με πελάτες. Ε, επιβεβαιώθηκε ότι Επιβεβαιώθηκε ότι οι καταναλωτέ δεν γνωρίζουν τις τιμέ που πρόκειται να πληρώσουν και οι υποχρεωτικές πληροφορίες των επιχειρήσεων δεν φτάνουν ουσιαστικά στον καταναλωτή. Ε, υπάρχουν και άλλες τεχνικές εφαρμογές όπως το VOIP, τις οποίες πιστεύω ότι θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στο νομοθετικό αυτό μέτρο. Η τεχνική, η τεχνολογία θα εξελιχθεί πολύ ε, σύντομα και ε, ας μην βρεθούμε στη θέση να πρέπει να συμπληρώσουμε ε, την νομοθετική πράξη με τις τεχνολογίες αυτές. Τέλος, ως προς ε, την ρήτρα απόσυρση στο Sunset Clause για το 2013. Δεν μπορώ να συμφωνήσω με μια τέτοια ρήτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ναι, έχω περάσει χρόνια στην Αυστρία, γι' αυτό ε, μου είναι πολύ γνωστή η πολύ γνωστά τα γερμανικά που μιλάτε. Η κυρία Κάριν Ρίς Ευχαριστώ, εγώ θα μιλήσω δανέζικα. Και θα με αγαπήσετε. Μάτς μούτς. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα θυμούνται κάποιοι ότι κάποιο με κατηγόρησε, ότι ο συνάδελφο κύριο Καμάλ με κατηγόρησε σε προηγούμενη συνεδρίαση ότι είμαι κομμουνίστρια. Αν είμαι εγώ κομμουνίστρια δεν ξέρω καθόλου τι είναι ο κύριο Καμάλ, αλλά τέλο πάντων αυτό είναι άλλη συζήτηση. Θα ήθελα να τονίσω ότι οι ε, απόψεις μου στο θέμα αυτό δεν ε, προέρχονται από τη Μόσχα, προέρχονται από ε, τη φιλελεύθερη σκέψη και την κοινή λογική. Ως φιλελεύθερη δεν θέλω να ρυθμίσω την αγορά μόνο και μόνο για να, έχω, για να έχουμε ρύθμιση, αλλά επειδή έχουμε μια αγορά που δεν λειτουργεί. Καλά. Είχα μια συνάντηση με τον κύριο Καμάλ, πολύ επικοδομητική συζήτηση, μου υποσχέθηκε ότι θα γράψει προκλητική έκθεση και να πω ότι τήρησε το λόγο του και χαίρομαι γι' αυτό. Ε, βρίσκω πολύ λογική την πρόταση της Κομισιόν ως σημείο κίνησης. Θα ήθελα όμως το πλαφόν για τα SMS και στη χοντρική και στην ε, λιανική ε, να μειωθούν, διότι τα πρότυπα που προτείνει η Κομισιόν συνεχίζουν να είναι υπερβολικά ψηλά σε σχέση με το πραγματικό κόστος ε, για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Ταυτόχρονα θα ήθελα ο ε, καταναλωτής να προστατεύεται από ε, παραφουσκωμένους ε, λογαριασμούς. Θα πρέπει λοιπόν ο, κα, καταναλωτής να έχει τα κατάλληλα μέσα στη διάθεσή του ώστε να μπορεί να προβλέψει το κόστος θα πρέπει να θυμόμαστε ότι ε, η ρύθμιση του roaming ε, σκοπό έχει να προωθήσει την καινοτομία. Όταν ζούμε σε μια Ευρώπη χωρίς ε, σύνορα δεν θα πρέπει η επικοινωνία μας να εμποδίζεται από υπερβολικές τιμές. Θα πρέπει δηλαδή να μειωθούν οι τιμές ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να υποφεληθούν από αυτές τις υπηρεσίες. Η ισορροπημένη ρύθμιση θα βελτιώσει την ασφάλεια για τους καταναλωτές και θα δώσει αρκετή ευελιξία στους, ε, ε, ε, στις επιχειρήσεις. και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, τους συντρόφους θα έπρεπε να πω. Ευχαριστώ. Βλέπω να αλλάζουν τα μέτωπα στο θέμα αυτό. Αν σκεφτούμε ποιος επωφελείται από την περιαγωγή, Ποιο ε, επωφελείται από την εσωτερική αγορά. Μόνο οι υπάροχοι των υπηρεσιών εποφελούνται διότι οι καταναλωτές ε, ε, είναι αποκλεισμένοι από την κυρία αγορά. Αν είμαι στο, στο ΚΕΛ και θέλω να στείλω ένα SMS στην Γαλλία, πρέπει να πληρώσω περιαγωγή. Κάτι πάει στραβά εκεί και γι' αυτό θα ήθελα να συμφωνήσω απόλυτα με την προλαλήσασα. Δεν λειτουργεί η αγορά και θα θέλουμε, θέλουμε να, να κάνουμε την αγορά αυτή να λειτουργεί καλύτερα και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, παραταθεί η, ο κανονισμός ε, για την παριαγωγή και θα ήθελα να αναφέρω ένα θέμα που πρέπει να συζητήσουμε. Ε, το 2009 λίγη η θητεία του Κοινοβουλίου και θα ξεκινήσουμε πάλι τις εργασίες μας στο δεύτερο εξάμεινο του 2009 και θα είναι ήδη αργά να συζητήσουμε την παράταση του κανονισμού. θα πρέπει να το κάνουμε αυτό τώρα εδώ. Συμφωνώ με τον κύριο Καμάλο ότι δεν έχουμε επαρκή στοιχεία. Όμω όμως ο χρόνος και θα ήθελα να σας θυμίσω ότι ε, η Επιτροπή αυτή του Κοινοβουλίου μας ε, ζήτησε να συμπεριληφθούν τα SMS στο δεύτερο στάδιο και υπήρχαν λόγοι γι' αυτό. Οι λόγοι ήταν οι μη διαφανείς τιμές στα SMS αλλά και στα δεδομένα. Δεν υπάρχει διαφάνεια. Όταν ακούω να μιλάμε για ε, καινοτομία και μιλάμε για τις συσκευές, κύριε Καμάλ, πρέπει να διαφωνήσω μαζί σας. Προέρχομαι από χώρα όπου γίνονται συσκευέ με νέε συμβάσει, αλλά ο καταναλωτή δεν έχει ελευθερία απόφαση, ε. και αυτό δεν είναι διαφανές. Ε. Δεν θέλω αυτομάτως με νέα σύμβαση να μου δίνουν νέα συσκευή. Θέλω να μπορώ να αποφασίσω ε, αν θέλω μια ε, πιο, πιο καλή σύμβαση ή πιο σύντομη διάρκεια της ε, σύμβασης αυτής. Θα πρέπει ο καταναλωτής να έχει ελευθερία επιλογής. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Και τώρα ανοίγω, θα δώσω το λόγο στους ελεύθερους αγορητές. Πρώτο τον κύριο Μάιλομπ. Ευχαριστώ. Καταρχήν συμφωνώ με τον κύριο Καμάλ ότι όντως χρειαζόμαστε περισσότερες πληροφορίες για την υλοποίηση της πρώτης οδηγίας. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Του πρώτου κανονισμού, με συγχωρείτε, διορθώνει ο μιλητής. Ιδίως υπό το φως των συζητήσεων που γίνονται αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε βεβαίως να ξεφύγουμε από το φιλοσοφικό ερώτημα που εγείρεται. Η Ευρώπη κάποτε είχε την πρώτη θέση, γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι εξακολουθεί να την έχει στην ε, τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας. Ε, ποια είναι τα αποτελέσματα των ρυθμίσεών μας στις εξελίξεις της τεχνολογίας. Ήμασταν οι πρώτοι. Δεν πρέπει να το χάσουμε αυτό, ούτε να χάσουμε τη θέση που είχαμε. Συμφωνώ βέβαια ότι η διαφάνεια είναι ένα θέμα κλειδί και πρέπει να το εξετάσουμε. Ένα από τα κυριότερα σημεία της διαφάνειας είναι το πώς οι πελάτες ή οι καταναλωτές ενημερώνονται για τα όρια. Όλοι μας έχουμε εμπειρίες ε, ε, όταν ξεπεράσαμε τα όρια και ε, χρειάστηκε να ξανακάνουμε σύνδεση με το κινητό μας και χάσαμε και χρόνο και χρήμα. Ε, είναι πολύ σημαντικό αυτό, ιδίως όταν κανείς κατεβάζει διάφορα δεδομένα και στοιχεία και ξαφνικά φτάνει στο όριο και κόβεται η σύνδεση. Το μέλημα είναι πώς να το κάνουμε πιο φιλικό προς τον καταναλωτή το όλο ζήτημα. Κάποιες πολύ σύντομες προτάσεις. Καταρχήν πιστεύω ότι οι καταναλωτές καταναλωτές δεν πρέπει να, ότι η σύνδεση των καταναλωτών δεν πρέπει να αποκόπτεται απότομα. Ε, οι καταναλωτές θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να επιλέγουν αν θέλουν αυτόματα να κόβεται η σύνδεσή τους όταν φτάνουν στο όριο. Θα πρέπει να έχουν δηλαδή αυτή την επιλογή, τη δυνατότητα επιλογής. Γιατί κάποιοι δεν θέλουν να διακοπεί η σύνδεσή τους και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν τις συνέπειες. Δεύτερον, ο τρόπος που εκφράζουν οι εταιρείε τα όρια όπου κόβεται η σύνδεση είναι λίγο ασαφή Τι, το όριο που έγκυται στον όγκο των δεδομένων, στην οικονομική του αξία. Ε, το ζήτημα αυτό έχει μεγάλο αντίκτυπο σε εκείνε τι χώρε και σε εκείνε τι εταιρείε που είναι καθαρή εισαγωγή τη περιαγωγή και οχι εξαγωγή. εξαγωγής. Έχουμε μεγάλα κράτη-μέλη και μικρά κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά υπάρχουν και μικρέ και μεγάλε εταιρείε επίση και έχουμε και μικρές χώρες με μικρές εταιρείες. Και αυτό έχει σημασία. Γιατί ιδίως για τις νότιες, τις μικρές νότιες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες βασίζονται στον τουρισμό. Ε, είναι καθαρή εισαγωγή οι χώρες αυτές και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γενικά ως τελευταίο μου σχόλιο, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια πολύ πιο ισόρροπη προσέγγιση και ίσως να υποβάλω και κάποιες τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να προστατεύσουμε ε, αυτούς που είναι καθαροί εισαγωγής. Να μην ε, προστατεύσουμε μόνο τις εταιρείες που είναι εξαγωγής. Πρέπει να βρούμε μια ισορροπία Ίσως μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία στην Επιτροπή μας, γιατί το σημαντικό, όταν το δει κανεί από το παγκόσμιο πρίσμα της προστασίας του καταναλωτή, το ζήτημα είναι πώς θα προστατεύσουμε τα συμφέροντα του καταναλωτή και πώς να το κάνουμε αυτό με λογικό τρόπο και χωρίς να υπονομεύσουμε την αξιοπιστία του κλάδου γενικά, αλλά και για κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Πράγμα που είναι πολύ δύσκολο Ε, εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση της ε, διακοπής της ε, σύνδεσης, νομίζω ότι τα πράγματα όλο θα περιπλέκονται και όλο και σε πιο δύσκολη θέση θα περιελχόμαστε. Ο κύριος Χάρμπορ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνδέσω τη συζήτηση εδώ με την στήριξη που είχα από την Επιτροπή για το έργο που έκανα για τη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή. Τότε διαπραγματεύτηκα πολύ έντονα είχα μακρές διαπραγματεύσεις με την ε, Προεδρία, την Τσεχική και τη Δανική. Ε, υπάρχει μια σημαντική αύξηση των μέτρων διαφάνειας που έχουν υιοθετηθεί. Άλλο ένα σημαντικό μέτρο είναι να τους δώσουμε δικαιώματα ε, ως προς το μέγιστη διάρκεια των συμβάσεων και άλλα μέτρα διαφάνειας. Νομίζω ότι η Επιτροπή μας πραγματικά έχει πάρει το σωστό δρόμο. Και νομίζω ότι έχουν δίκιο όσοι συγκεντρώνουν την προσοχή τους σε αυτά τα πολύ κρίσιμα μέτρα για τους καταναλωτές. Να μπορούν δηλαδή οι καταναλωτές να κάνουν επιλογές ε, όταν τους γίνονται πολλές και πολύπλοκες προσφορές, να μπορούν να επιλέξουν σωστά. Βλέπουμε διαρκώς διάφορες προσφορές, δωρεάν πακέτα ή δέσμες προσφορών, ε, οι προτιμησιακές ταρίφες για ορισμένες χώρες, ε, για χώρες στις οποίες υπάρχει υψηλός όγκος δραστηριοτήτων και χάνεται ο καταναλωτής. Κάτι που δεν είδα στα έγγραφά μας είναι κάποια αλλαγή στη στάση της Επιτροπής. Ε, εσείς είσαστε ευχαριστημένος με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που περιλαμβάνονται στον κύριο Φάκελο ή πρέπει εμείς να κοιτάξουμε και να ερμηνεύσουμε τα πράγματα και να προσπαθήσουμε άλλα σημεία να τα ενισχύσουμε και να επιλύσουμε κάποια περίπλοκα ζητήματα, ιδίως με τα θέματα περιαγωγή. Ε, για του χρήστε του διαδικτύου, εγώ βρίσκω τι προσφορέ πραγματικά κατανόητε. Εγώ πρέπει να διαβάσω πολύ προσεκτικά το λογαριασμό μου για να καταλάβω γιατί πράγμα με, ε, σε τι αντιστοιχούν οι διάφορε χρεώσει. και καταλαβαίνω ότι τα πράγματα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Όλα αυτά προκαλούν πολύ μεγάλη απαγόρε, απογοήτευση. Ένα, μια από τι εταιρείε ε, μου κάνει μία σημείωση όταν υπερβαίνω ένα συγκεκριμένο ποσό μηνιαίως. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό ε, και γενικά θεωρώ ότι πρέπει να παράσχονται υπηρεσίες τέτοιες στους καταναλωτές, κάτι που πρέπει να δούμε και στο πακέτο μας για την περιαγωγή. Εδώ τι μας ζητούν να κάνουμε, να δούμε τι γενικέ αρχέ. Κάναμε μια πολύ παρατεταμένη συζήτηση στην Επιτροπή αυτή, η οποία άλλαξε ριζικά τι αρχικέ προτάσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το διεθνή περιαγωγή. Είπαμε ότι καλό είναι να πυροδοτήσουμε τον διεθνή ανταγωνισμό, αλλά εγώ και άλλοι προειδοποιήσαμε τότε ότι αν θέλουμε να μειώσουμε τον ανταγωνισμό, αν θέλουμε να κάνουμε τη ζωή εύκολη για τι εταιρείε, γιατί η τιμολόγηση είναι η πιο δύσκολη απόφαση σε οποιαδήποτε εταιρεία στον χώρο των τηλεπικοινωνιών όπου έχει υψηλό πάγιο κόστο και προσπαθεί να δει πώ να αυξήσει τα κέρδη σου μέσα από τι προσφορέ που κάνει κτλ. Αν θε λοιπόν να μειώσεις, να κάνεις τη ζωή εύκολη στους ανθρώπους πρέπει να, δια, να περάσεις διατίμηση και να θεσπίσεις ανώτατες τιμές. Αυτό όμως κανείς δεν το θέλει. Και αν δει κανεί την αρχική έκθεση για, το διεθνέ, για τη διεθνή περιαγωγή θα το δει και μην ξαφνιάζεται ότι οι τιμές ε, που προσφέρονται στους καταναλωτές είναι όλες εκεί κοντά, στην ανώτατη τιμή. Μας ξαφνιάζει αυτό. Υπάρχει και αυτή η πρόταση για τα SMS, τα μηνύματα. Και αυτό με ξάφνιασε. Η πρόταση σε μερικές χώρες μάλλον ε, χρεώνουν περισσότερο για τα SMS. Εντάξει, αυτό είναι θέμα αγοράς. Και μια πιστεύω ότι μια ευρωπαϊκή ανώτατη τιμή θα επηρέαζε τις τιμές σε κάθε εθνική αγορά. Εντάξει, μπορεί να προστατεύει τους καταναλωτές αυτό, αλλά θεωρούμε ότι είναι σωστό να δουλεύει έτσι η αγορά. Όσο αφορά τώρα η περιεγωγή δεδομένων και μηνυμάτων, για άλλη μια φορά θα ήθελα να, πω, να προσθέσω σε αυτά που είπε ο Νίκολάη Μάρτινοφ. Είμαστε σε μια θέση όπου όλες οι εταιρείε κινητής τηλεφωνίας ε, εξετάζουν αυτή τη στιγμή διάφορες επενδύσεις. Θέλουν να αυξήσουν τη χωρητικότητα του δικτύου γιατί η ζήτηση για την περιαγωγή δεδομένων αυξάνεται δραματικά και προσπαθούν τώρα να κάνουν τις τιμές τους και τις προσφορές τους κατά τρόπο που να μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις υπηρεσίες τους από τον υπολογιστή σου στο σπίτι σου. Και αυτό συμβαίνει σε πολλές ε, χώρες, ε, είναι κάτι που το ζητούν και οι τακτικοί πελάτες των εταιριών και και υπάρχει τώρα συνδυασμός διαφόρων προσφορών ε, για τον κόσμο αντί να στέλνει ηλεκτρονικά μηνύματα να στέλνει SMS. Και καλό θα είναι δεν είναι δυνατόν μάλλον να επιβάλλονται ανώτατα όρια, να επιβληθεί διατίμηση δηλαδή ε, στις υπηρεσίες αυτές όταν η κατάσταση μεταβάλλεται με τέτοια ταχύτητα όπως στις τηλεπικοινωνίες. Πολλοί από εμά χρησιμοποιούμε το Skype που είναι τηλεφωνία μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το χρησιμοποιεί πολλοί κόσμος, ιδίως άμα θέλει να κάνει ε, τηλεφωνήματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί το κόστος είναι πάρα πολύ μικρό. Επίσης, αν έχεις ε, τηλεφωνία που συνδέεται με τον ε, προσωπικό σου υπολογιστή, μπορείς να έχεις και φωνητική ε, τηλεφωνία. Η, η αγορά λοιπόν αλλάζει γρήγορα, αλλάζει μαζικά και ίσως σε μια περίοδο 5, 6, 7, 8, 10 ετών μπορεί το θέμα της περιαγωγής να μην απασχολεί κανέναν, να έχουμε περάσει σε άλλα πράγματα. Εμείς θέλουμε να μας εξηγήσουν, λοιπόν, γιατί θεωρείται καλό για τους Ευρωπαίους ε, καταναλωτές η ψήφιση της οδηγίας για την περιαγωγή. Ευχαριστώ. Πολύ γρήγορα θα περάσουμε στο επόμενο ε, θέμα. Ένα σύντομο σχόλιο, λοιπόν, από την Επιτροπή και θα ολοκληρώσουμε πάνω σε αυτό. Ε, Η Επιτροπή θα ήθελε καταρχήν να ευχαριστήσει τον κύριο Καμάλ για αυτή τη συζήτηση και ε, να ευχαριστήσουμε επίσης και τους σκιώδεις εισηγητές για την ε, συζήτηση στην Επιτροπή. Όπως ξέρετε, εμείς δεν συμφωνούμε με τις απόψεις σας για την αφαίρεση της διατίμησης, για τις ανώτατες τιμές δηλαδή, και αυτό γιατί πιστεύουμε ότι αυτό δεν είναι προς το συμφέρον του καταναλωτή και δεν εξυπηρετεί τους στόχους της εσωτερικής αγοράς. Θέλω να τονίσω ότι η πρόταση κανονισμού δεν έχει να κάνει με τη θέσπιση τιμών, ε, την επιβολή τιμών, ούτε για έχει να κάνει με την απάλληψη της κερδοφορίας. Ο στόχος είναι η απάλληψη της υπέρογκης κερδοφορίας. Πρέπει να θυμόμαστε ότι ο κανονισμός για την περιαγωγή ήταν απότοκο της αποτυχίας της αγοράς στο συγκεκριμένο τομέα και της ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι υπέρογγες τιμολογήσεις ε, στα τιμολόγια και υπήρχε έκκληση από όλους, ε, από τους καταναλωτές, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να κάνουμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να συμπεριλάβουμε σε αυτό και τα μηνύματα, τα SMS. Και επίσης ε, μας ζητήθηκε να πριν από το έτος του 2008 να ξαναδούμε το ζήτημα. Εμείς πιστεύουμε ότι η αξιολόγηση αντικτύπου είναι πολύ λεπτομερής, πολύ αναλυτική και βλέπουμε ότι τα νέα δεδομένα που παρουσίασε η ERG πριν από δύο εβδομάδες πραγματικά καταγράφουν τις ίδιες τάσεις όπως και οι προηγούμενοι. Το γεγονός ότι οι εταιρείες τηλεφωνίας δεν επέλεξαν να εκμεταλλευθούν τα πλεονεκτήματα της ευελιξίας του κανανισμού και να ανταγωνιστούν μεταξύ τους, δείχνει σαφώς πως η έλλειψη ανταγωνισμού υπάρχει. Και εξακολουθεί να ισχύει αυτή η έλλειψη ανταγωνισμού στον τομέα. Και αυτό δεν είναι μόνο η άποψη της Επιτροπής. Είναι η άποψη και των ομάδων καταναλωτών, των NRAs, των κυβερνήσεων και ακόμη και ορισμένων εταιριών κινητής τηλεφωνίας. Κατά την άποψή μας, η πρότασή μας είναι καλά ισορροπημένη, αναλογική, εξασφαλίζει ευελιξία και λαμβάνει πλήρως υπόψη τις εξελίξεις. Και γι' αυτό για την περιαγωγή των δεδομένων δεν έχουμε προτείνει ε, διατίμηση στις λιανικές τιμές. Παρακολουθούμε απλώς τις εξελίξεις στον τομέα της λιανικής στην αγορά αυτή. Ωστόσο πρέπει να πούμε επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί πως ο κανονισμός για την περιαγωγή είναι ένα εξαιρετικό μέτρο, ένα μέτρο που λαμβάνεται κατ' εξαίρεση. Ο στόχος δεν είναι να έχουμε έναν μόνιμο κανονισμό. Ο στόχος είναι οι παίκτες της αγοράς να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, προς όφελος των καταναλωτών. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει σήμερα και για το λόγο αυτό κάνουμε αυτή την πρόταση. Και, είμαστε... και θα είμαστε πολύ ευτυχείς να συζητήσουμε αναλυτικά τις προτάσεις μας μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Um, Uh, uh, Ευχαριστώ. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους κοιόδης ε, εισηγητές για τα σχόλιά τους. Ε, νομίζω ότι καλώς έκαναν και ήταν προκλητικοί, καλό είναι να είναι κανείς προκλητικός. Υπάρχει σίγουρα μία συνένεση ε, για την διαφάνεια. Νομίζω ότι αυτό μας παρέχει μια καλή βάση εργασίας. Ενδιαφέρον είναι ότι παρότι εγώ μίλησα με τις εταιρείες και τους παρουσίασα τα θέματα ε, με τη διαφάνεια και τα τιμολόγια, μου είπαν ότι ούτε και αυτούς τους συμφέρει να βγαίνουν στις εφημερίδες ιστορίες με καταναλωτές που παραπονιούνται για τα τιμολόγια τους και τους λογαριασμούς τους. Ε, νομίζω ότι είχαν αρκετά προβλήματα μέχρι στιγμής και οι εταιρείε με αυτά. Ο κύριος Μπουφόν είπε ότι θέλει να καταλάβει λίγο καλύτερα για τις διαφορετικές τιμές. Είναι πολλοί οι παράγοντες. Γιατί δεν απευθύνεται κατευθείαν σε μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας να τη ρωτήσει. Δεν, δεν είναι η θέση μας εδώ να συζητήσουμε τις διαφορετικές τιμές. Από πολλές παρεμβάσεις ε, φάνηκε να συνάγεται ότι όλες οι τιμές θα βασίζονται στο κόστος. Ε, υπάρχουν πολλοί τρόποι να αντιμετωπίσει κανείς το θέμα των τιμών. Όπως ο κύριος Χάρμπορ είπε, είναι πολύ πολύπλοκο το ζήτημα της ε, τιμολόγησης. Αν έχουμε ως βάση μας μόνο το κόστος, Ίσως τελικά σε ορισμένες ε, χώρες το κόστος να ανεβεί πάρα πολύ. Το κόστος των συσκευών δηλαδή μπορεί να αυξηθεί πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να δοθεί μια ευελιξία, να μπορέσει ο καθένας να βρει τη δική του εναλλακτική λύση, να γίνουν προσφορές περιαγωγής, δεδομένων, μηνυμάτων. Κάποιος ανέφερε και συμφωνώ κι εγώ ότι μερικές εταιρείες, ιδίως κατασκευαστές συσκευών, μπλοκάρουν κάποιες από τις φωνητικές λειτουργίες. Ε, εμείς, ε, ε, μάλλον αυτό το κάνουν για λόγους διαφάνειας και δεν δίδεται επιλογή στον αγοραστή, στον πελάτη επειδή ίσως η πλήρης ε, διαθεσιμότητα των φωνητικών λειτουργιών προς τους πελάτες είναι αντιανταγωνιστική. Πολύ φοβάμαι ότι η αγορά των SMS ε, πεθαίνει. Οι όγκοι αυξάνονται δραματικά, αλλά δεν νομίζω ότι θα επιβιώσουν. Εγώ ήδη έχω μια συσκευή στα χέρια μου που ε, μου δίνει άλλες επιλογές. Μπορώ να στείλω ένα ηλεκτρονικό μήνυμα και όχι ένα SMS. Μου έρχεται πιο οικονομικά. Όλα αυτά τα πράγματα θα καθίστανται πιο δυνατά όσο θα εξελίσσεται η τεχνολογία. Ε, εμείς δεν θα πρέπει να προκαταλαμβάνουμε εύκολα τη μελλοντική τεχνολογία γιατί δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτή. Οι ρυθμιστές δεν πρέπει να προσπαθούν να επιλύσουν προβλήματα που ακόμα δεν υπάρχουν. Ας μην λοιπόν αποφασίζουμε για τεχνολογίες που δεν υπάρχουν ε, ακόμη. Ας δούμε ποιες είναι οι τεχνολογίες σήμερα και ας επιλύσουμε τα υπάρχοντα προβλήματα. Ε, χαίρομαι πολύ που μερικοί εδώ μέσα εξακολουθούν να με αγαπούνε Ε, δεν, ε, δεν σας αποκάλεσα ε, κομμουνίστρια. Κάποιος από τους φιλελεύθερους συναδέλφους μου μου είπε κάποτε είσαι πολύ φιλελεύθερος για να είσαι φιλελεύθερος. Πας περιπτώσει. Ε, υπάρχουν οι προσεγγίσεις που βασίζονται στο κόστος και οι προσεγγίσεις που βασίζονται στις τιμές και πρέπει να τα διαχωρίζουμε αυτά. για την ε, τιμολόγηση των συσκευών. Θα ήθελα κάποια στιγμή να καθίσουμε να κουβεντιάσουμε, να μου πείτε ποια είναι η άποψή σας ε, για τις τιμές των συσκευών. Τώρα για την πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να δούμε τις τρεις-τέσσερις εναλλακτικές λύσεις που έχουν προταθεί να μου, και να μου πείτε τι σκέφτεστε για κάθε μία από αυτές. Τώρα προς την Επιτροπή. Όπως ο Μάλκομ είπε, έχει εργαστεί εκείνο στην διαμόρφωση των τιμών και εγώ έχω εργαστεί στην ε, διαμόρφωση των τιμών. Όπω και αν το, ονομάσουμε παρεμβατικά μέτρα, διατίμηση ή ξέρω εγώ, πάντω ερχόμαστε και παίζουμε το ρόλο του, του παίκτη τη αγοράς. Η εταιρεία κινητής τηλεφωνίας δεν πρόκειται να συμφωνήσει ποτέ να προσφέρει τέτοια προϊόντα εάν ξέρει ότι στο τέλος του χρόνου θα υπάρξει άλλη διατίμηση. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ήθελα να πω ότι σήμερα το πρωί αποφασίσαμε να αναβάλουμε την ψηφοφορία για τη Δευτέρα 2 Μαρτίου. Ο κύριος Μάντερς για την προστασία των καταναλωτών και των βιντεοπαιχνιδιών. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αφήνουμε τώρα πίσω μας ε, τα τηλεφωνικά παιχνίδια και φτάνουμε στα βίντεο παιχνίδια. Και εδώ μιλάμε για κίνητρα ώστε να λειτουργεί καλά η αγορά. Η έκθεσή μου ασχολείται με ε, τα ε, μειονεκτήματα των βιντεοπαιχνιδιών, ιδιαίτερα για τους ανηλίκους. Ε, στα, τον τελευταίο καιρό είχαμε τεχνικές τροποποιήσεις, ε, έχουμε όλο και περισσότερα επιγραμμικά παιχνίδια, όλο και περισσότερα βίντεο παιχνίδια υπάρχουν, ε, όλο περισσότερα αναπτύσσονται και για ενήλικες βέβαια μπορεί να τα παίξουν και τα παιδιά και ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, γύρω από αυτό επικεντρώνεται η πολιτική συζήτηση. Ουσιαστικά ήθελα να πω ότι τα βιντεοπαιχνίδια δεν είναι ε, από μόνο τους βλαβερά. Δεν θέλω να τα εξοραίσω. Ε, είχαμε σεμινάριο όπου ε, μίλησαν εμπειρογνώμονες από πολλές χώρες και Ήταν χρήσιμη αυτή η ανταλλαγή απόψεων διότι διαπιστώσαμε ότι έχουν πολύ περισσότερη προστιθέμενη αξία τα βιντεοπαιχνίδια ε, για την ανάπτυξη της ε, κοινωνίας μας. Ε, τα, ότι είναι νέο δεν είναι απαραίτητα τρομακτικό. Θα πρέπει να υποφεληθούμε από την πρόοδο και μην ξεχνάμε τα ωφέλη που μπορεί να έχει η νέα γενιά από αυτό το 0,30% ε, των ε, παιχνιδιών θα μπορούσαν να είναι ε, βλαβερά, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν είναι προβληματικά. Θα πρέπει να μεταφέρουμε τα πρότυπά μας στα σχολεία, στα παιδιά, στα σχολεία, στους καθηγητές. Υπάρχει το κουμπί για την προστασία των παιδιών, ώστε οι γονείς να, μπορούν, να φροντίζουν ότι τα ε, παιδιά παίζουν ε, παιχνίδια τα οποία δεν εξοραίζουν τη βία. Ε, Πέγγι λέγεται μια θελοντική ένωση που θέτει τα όρια ηλικίας για τα διάφορα παιχνίδια. Σωστό είναι λοιπόν να φροντίσουμε να τρέχουν ε, παράλληλα οι ε, πολιτικές ε, θέσεις στην Ευρώπη. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, έχουμε αρκετά αυστηρή νομοθεσία. Η παραγωγή παιχνιδιών μεταφέρονται στο εξωτερικό και κατόπιν παρέχουν τα ε, παιχνίδια αυτά επιγραμμικά και εντός της, ε, και εντός της Γερμανίας. Ε, θέλουμε λοιπόν ευρωπαϊκά μέτρα ώστε να μπορούμε να εφαρμόσουμε σωστά τα όρια ηλικίας. Θα πρέπει δηλαδή να συντονιστούμε μεταξύ μας και χρειαζόμαστε τη δυνατότητα να ελέγξουμε την πρόσβαση στα διάφορα παιχνίδια. Θα πρέπει δηλαδή να ε, γνωρίζουμε ότι δεν είναι υπερβολικά νέοι οι χρήστες. Η Γαλλική Προεδρία πρότεινε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ταυτότητα την οποία να χρησιμοποιεί κανείς σε όλη την Ευρώπη, όχι μόνο στη χώρα. Αυτό ήταν μια πρόταση σχετική. Βρίσκουμε σημαντικό να είναι ενιαία η σήμανση των παιχνιδιών αυτών στην Ευρώπη και πιστεύουμε ότι η αυτορύθμιση του τομέα μέσω του πέγι e έχει λειτουργήσει καλά. Έχουν γίνει δηλαδή πράγματα όλα αυτά ισχύουν για παιχνίδια που μπορεί να αγοράσει κανείς ε, σε κατάστημα, μπορεί να ε, ελεγχθεί η αγορά. Είναι πολύ απλό να δει κανείς εάν ο χρήστης ε, έχει την κατάλληλη ηλικία, μπορεί να ζητήσει την ταυτότητά του. Η Πέγγι λέει όμως ότι αυτή η ρύθμιση δεν αρκεί για τις πωλήσει μέσω διαδικτύου. Χρειάζεται περισσότερη δουλειά το θέμα αυτό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κληθούν ε, να ε, αναλάβουν ε, τις συστάσεις της ΠΕΚΙ σε μεγαλύτερο βαθμό στην νομοθεσία τους. Ο κοινός μας στόχος είναι η εναρμόνιση. Και φτάνω στα συμπεράσματά μου. Χθε επιβεβαιώθηκε από τους πυρογνώμονε στην ακρόαση ε, το συμπέρασμα μου δεν χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα πρέπει να δημιουργήσουμε κίνητρα. Ο Γάλλος εμπειρογνώμων ε, ήταν κάπω νεότερος από μένα, ήταν όμως πραγματικό επιρογνώμονας είπε λοιπόν ότι θα πρέπει να ε, μάθουμε να ε, ε, ζούμε καλά με τις καινοτομίες στην κοινωνία μας. Θα πρέπει να είμαστε περίεργοι, θα πρέπει να τις δεχόμαστε. Η τηλεόραση ήταν πριν από 30 χρόνια εργαλείο του διαβόλου. Οι γονείς μας μας μας προειδοποιούσαν για την τηλεόραση. Τώρα όμως είναι διαφορετικά τα πράγματα. Ναι, ανέφερε για παράδειγμα ε, στην πορνογραφία ε, χθε ο πυρογνώμων. Οι νέοι γνωρίζουν πολύ καλά τι ε, θα έπρεπε να βλέπουν και τι όχι αυτό. Μεταφέρεται μέσω της ανατροφής ή μέσω του σχολείου. Αυτό δεν μπορεί να μεταφερθεί μέσω της νομοθεσίας. Θα ήθελα να σας καλέσω το σύστημα πέγι, e το σύστημα ε, ορισμού ορίων ηλικίας, να εξελιχθεί περαιτέρω, να καλύψει και τα επιγραμμικά βιντεοπαιχνίδια. Θα ήθελα ε, να το τονίσω αυτό και θα ήθελα επίσης ε, στο εκπαιδευτικό σύστημα να υπάρχει να διδάσκεται ε, μια πιο ε, συνειδητή χρήση των βίντεο παιχνιδιών τα παιδιά, να μαθαίνουν ε, τις αξίες, τα πρότυπα, ώστε να μπορούν να κρίνουν μόνα τους εάν τους κάνει καλό ή όχι ένα βίντεο παιχνίδι. Ο καθηγητής Τζέφρι Γκόλστιν είπε ότι δεν υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι όταν παίζει κανείς βίντεο παιχνίδια επηρεάζεται αρνητικά και ότι θα ε, να κάνει την πραγματικότητα αυτά που κάνεις στο παιχνίδι. Αυτό δεν έχει αποδειχθεί επιστημονικά. Σημαντικό είναι κατά την ανατροφή να ε, μαθαίνουμε στα παιδιά να μην ε, κάθονται 30 ώρες την εβδομάδα μπροστά στον υπολογιστή, ε, τότε εντάξει, τότε δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα άλλο, ούτε να μάθει, ούτε να παρακολουθήσει μαθήματα, τίποτα. αυτό όμως δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο των παιχνιδιών. το ίδιο άλλο ισχύει με τις συνομιλίες μέσω κινητού, με τη χρήση του κινητού. δεν έχει να κάνει με το περιεχόμενο, έχει να κάνει με τις αξίες που μεταφέρουμε στα παιδιά. Δεν πρέπει κανείς να κάνει το ίδιο πράγμα την, όλη τη μέρα και αυτό ε, θα πρέπει να το μεταφέρουμε στα παιδιά με την ανατροφή τους. Ε, οι γονείς θα το κάνουν αυτό, τα σχολεία θα το κάνουν αυτό. Ελπίζω οι συνάδελφοι να συμφωνήσουν μαζί μου. Ε, αν όχι, σας παρακαλώ να μου το πείτε. Ε, η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 26 Ιανουαρίου στις 12. Και τελείωσα έτσι την παρουσίασή μου. Ευχαριστώ. Thank you. Um, Ευχαριστώ κύριε Αγγελάκας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο εισηγητής, ο κύριος Μάντερς, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά, πολύ καλή έκθεση. Ε, διαβάζοντας τον τίτλο της έκθεσης αλλά και την πρόταση της Επιτροπής ε, αναφέρεται στην προστασία των καταναλωτών και ιδίως των ανηλίκων από τη χρήση των βιντεοπαιχνιδιών ε, δεν σημαίνει και θα συμφωνήσω με τον εισηγητή ότι ένα βιντεοπαιχνίδι είναι κατά ανάγκη επικίνδυνο. Κάθε άλλο μάλιστα. Πολλά βιντεοπαιχνίδια οξύνουν το πνεύμα και ιδιαίτερα το πνεύμα των νέων, τους φέρνουν κοντά στην τεχνολογία, τους γνωρίζουν νέους κόσμους και γενικά θα συμφωνήσω ότι ασκούν θετική επίδραση στην διαπαιδαγώγησή τους. Αυτό μάλιστα φάνηκε και με τη χθεσινή ακρόαση και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να συμβάλλουν πάρα πολύ και σε εκπαιδευτικούς στόχους. Από την άλλη μεριά όμως επειδή εδώ εμείς έχουμε ε, μπροστά μας να συζητήσουμε την προστασία των καταναλωτών και των νέων πρέπει να δούμε ποιους πιθανούς κινδύνους ε, έχουμε από τη χρήση των βιντεοπαιχνιδιών. Να προσθέσω στα θετικά ότι οι βιντεοπαιχνίδια χρησιμοποιούνται στους ιατρικ, σε ιατρικούς στόχους. Να προσθέσω στα θετικά επίσης ότι ακούστηκε και χθες στην ακρόαση ότι δεν σημαίνει ότι ένα, βίντεο, ένα βίαιο βιντεοπαιχνίδι συνεπάγεται και βίαιη συμπεριφορά των νέων και αυτό είναι εντυπωσιακό και εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον κάτι τέτοιο δεν έδειξαν οι, οι μελέτες που μας παρουσιάστηκαν. Αυτά που εγώ συγκράτησα και θεωρώ σημαντικά είναι τα εξής προβλήματα. Πρώτα απ' όλα ότι δεν είναι αντιστοιχισμένο σωστά, αν θέλετε συσχετισμένη, η ηλικία των νέων που βλέπουν βιντεοπαιχνίδια με το περιεχόμενο αυτών των βιντεοπαιχνιδιών που μπορεί να περιέχουν βίαιο ή μη υλικό. Και μάλιστα κοιτώντα την έκδοση που μας μοιράστηκε χθε από το πρόγραμμα Πέτζι, τα περισσότερα παράπονα σχετίζονται με την αναντιστοιχία ηλικιών και περιεχομένου βιντεοπαιχνιδιών. Το πρόγραμμα αυτό, το Page, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Είναι ένα πρόγραμμα αυτορύθμισης δεν είναι ένα νομοθετικό πλαίσιο των κρατών μελών, αλλά ε, νομίζουμε ότι θα έπρεπε να προχωρήσει κάποια στιγμή ίσως σε κάποια άλλου είδους ε, νομοθετική ρύθμιση, διότι αυτή τη στιγμή άλλοι το ακολουθούν και άλλοι όχι. Ένα άλλο σχόλιο έχει να κάνει με την απαγόρευση συγκεκριμένων παιχνιδιών. Στην αιτιολογική έκθεση της ε, Επιτροπής αναφέρεται ότι μόνο σε τέσσερις χώρες έχουν απαγορευτεί βίντεο Και μου κάνει εντύπωση ένα βιντεοπαιχνίδι ή είναι βίαιο και βλαβερό ή δεν είναι. Δεν μπορεί άλλοι να το θεωρούν επικίνδυνο για την παιδική ηλικία και κάποιοι άλλοι όχι. Λοιπόν, πρέπει ίσως να, να μπει ένας προβληματισμός κατά πόσον πρέπει να υπάρχουν παρόμοιοι κανόνες στην απαγόρευση των βιντεοπαιχνιδιών σε όλα τα κράτη-μέλη. Ενώ μια τρίτη παρατήρηση έχει να κάνει με το ότι αυτά τα βιντεοπαιχνίδια διαφημίζονται σε ορισμένες τηλεοράσεις, σε ώρες που παιδιά μικρής ηλικίας βλέπουν ίσως ακατάλληλα και βία παιχνίδια. Ε, σκέψη θα ήταν αυτές οι διαφημίσεις να υπάρχουν στην ζώνη εκείνη των ενηλίκων και όχι των, ε, παιδιών. Και σίγουρα οι ενήλικες, οι προστάτες, οι γονείς είναι αυτοί που θα αποφασίσουν εάν το παιχνίδι είναι κατάλληλο ε, η έκθεση είναι πολύ ισορροπημένη ε, υπάρχει ένα σχόλιο που το έχω θέσει στον εισηγητή σχετικά με το πόσο αυτά τα βιντεοπαιχνίδια πώς μπορούν να ελεγχθούν στα ίντερνετ καφέ, ιδιαίτερα δημοφιλή στη δική μου χώρα. Ε, από τη χθεσινή ακρόαση φάνηκε ότι και αυτό είναι ευθύνη των γονέων, που συμφωνώ απολύτως, αλλά δεν ξέρω κατά πόσον κάποιος που έχει οικονομικό συμφέρον να έχει νέους μέσα στο ίντερνετ καφέ, οι οποίοι παραμένουν πολλές ώρες και κερδίζει χρήματα, εάν θα τους ε, θα οριοθετήσει τι είδους βιντεοπαιχνίδια βλέπουν τα νέα παιδιά. Σε κάθε περίπτωση είμαστε υπέρ των βιντεοπαιχνιδιών, διότι περισσότερα είναι τα θετικά, σαφώς περισσότερα. Ας δούμε δύο-τρία σημεία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Νέρης εκ εξ μέρους του κυρίου Αμού. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εκ μέρους του κυρίου Μπενουά Αμό κάποιες τοποθετήσεις και εκτιμήσεις που θα ήθελα να σας μεταβιβάσω γιατί εκείνος δεν μπορούσε να είναι σήμερα εδώ και κάποιες προσωπικές μου απόψεις βεβαίως. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη δουλειά του σε αυτό το θέμα. Οι σημαντικές εξελίξεις στον τομέα των βίντεο παιχνιδιών και ιδίω στο κοινό που στοχεύουμε, αξίζουν να μελετήσουμε την υπόθεση αυτή προσεκτικά. Ιδίω ό,τι αφορά του νεότερου καταναλωτέ. Δεν πιστεύω και εγώ ότι ένα βίο παιχνίδι οδηγεί στην πραγματικότητα σε βίαιη συμπεριφορά. Κάποια περιεχόμενα όμω μπορεί να είναι ελαφρώ επικίνδυνα ή τουλάχιστον τρομακτικά για το νέο, νεαρό κοινό. Μιλάμε για τα βία παιχνίδια ή και αυτά με σεξουαλικό περιεχόμενο ή αυτά που οθούν προς ε, το ρατσισμό ή άλλα τέτοια φαινόμενα. Όπως ε, συμβαίνει σε όλες τις περιπτώσεις των τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να υπάρχει καθαρή σήμανση που να βοηθά την προστασία των καταναλωτών και να υπάρχει διεξοδική πληροφόρηση για το περιεχόμενο του προϊόντος που πρόκειται να δουν. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν μια πολιτική έτη και μια λύση θα ήταν το σήμα να αναγράφεται, να επισυνάπτεται πάνω στο δίτο προϊόν και όχι υπό ορισμένε συνθήκε και προποθέσει μόνο, αλλά σε κάθε περίπτωση. Ο εισηγητή νομίζω δεν θα πρέπει να είναι τόσο ενθουσιώδη για την αυτορύθμιση τη αγορά αυτή των προϊόντων. Ίσως θα χρειάζονταν αυστηρότερα μέτρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να καταλήξουμε σε ενιαίες προδιαγραφές και πρότυπα στην επικράτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσο για τις αγορές στο διαδίκτυο, να θυμίσω ότι υπάρχουν πολλά παιχνίδια που πολλούνται στο διαδίκτυο που μπορούν να τα προμηθευτούν οι καταναλωτές και δωρεάν. Ε, αλλά οδηγούν και στην απόκτηση άλλων αναπιστώσεων και μπόνους. Ε, θα πρέπει λοιπόν να, να προβλέψουμε ειδικού κανόνες και για αυτές τις ιδιαίτερες περιπτώσεις. Αυτά εκ μέρους του κυρίου Μπενουά και τώρα κάποιες προσωπικές μου παρατηρήσεις. Ήθελα εδώ να επιστήσω την προσοχή και δεν μιλώ ως βουλευτής, αλλά ως ειδική εκπαιδεύτρια για την έρευνα και την κοινωνική συμπεριφορά. Μην ξεχνάτε ότι κάθε φορά που ανακοινώνουμε κάτι τέτοιο, απευθυνόμαστε σε παιδιά που ζουν κατά τρόπο κατά τα άλλα φυσιολογικό και δεν έχουν ειδικά προβλήματα. Να επισημάνω λοιπόν ότι τα παιχνίδια αυτά κάποιες φορές οι ειδικέ περιπτώσει προσελκύουν τα παιδιά που έχουν οριακή συμπεριφορά, τις λεγόμενε περιπτώσεις borderline. Όμως, εκεί μιλάμε για, εδώ γενικά μιλάμε για μοντέλα, τα οποία δεν έχουν σκοπό την διαστρέβλωση, αλλά την ε, συνήθως όταν έχουμε περίεργες συμπεριφορές από παιδιά, αυτό είναι όχι το αίτιο το βιντεοπαιχνίδι, αλλά η συνέπεια. Δηλαδή κάποια βιντεοπαιχνίδια που έχουν βίαιο περιεχόμενο ανήκουν σε μια ευρύτερη ομάδα που θα καταναλώσει αυτό το παιδί που έχει ήδη μια προδιάθεση για βίαιη συμπεριφορά. Υπάρχει ένα σχετικό εθισμό λοιπόν το να συμπεριλάβουμε λοιπόν τα βιντεοπαιχνίδια σε ένα νομοθετικό πλαίσιο εφόσον μπορεί να έχουν και εκπαιδευτικό περιεχόμενο και να είναι εκπαιδευτικά εργαλεία, νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Θα πρέπει να φροντίσουμε κάποιες δυνατότητες που προσφέρει το βίντεο παιχνίδι δεν θα πρέπει να αφαιρεθούν αναγκαστικά. Μην ξεχνάμε ότι παιχνίδια όπως η, Φλόμιγα εισήχθησαν με ένα τέτοιο τρόπο σε νερότερες ηλικίε. Κύριε Μάντερς, θέλετε να σχολιάσετε. Ευχαριστώ. Να απαντήσω σε ορισμένες από τις παρατηρήσεις. Αυτό που προέκυψε και από τη χθεσινή ακρόαση είναι ότι οι γονείς είναι οι πρώτοι υπεύθυνοι που θα πρέπει να ξέρουν ότι εάν λόγω χάρη αφήσουν τα παιδιά τους να τρέχουν τους δρόμους κάθε μέρα, δεν μπορούν να ζητάνε από τις δημόσιες αρχές να λάβουν μέτρα γι' αυτό, πρώτα πρέπει να ξέρουν οι ίδιοι τι κάνουν τα παιδιά τους και να τα παρακολουθούν. Έπειτα, για τα παιδιά που ήδη έχουν κάποια ψυχολογική προδιάθεση αρνητική και το πώς χρησιμοποιούν τέτοια βιντεοπαιχνίδια, θα έπρεπε τέτοια παιδιά ίσως να τίθενται υπό ψυχιατρική παρατήρηση, να τα παρακολουθεί ένας ψυχολόγος στα βιντεοπαιχνίδια. Θα έχουν ούτως ή άλλως πρόσβαση. Δεν είναι λοιπόν αυτό η απάντηση. Και επειδή όλα αυτά περνάνε από το διαδίκτυο, οι αρχέ δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση και να ελέγξουν το περιεχόμενο. Οι ειδικοί χθε μας έλεγαν ότι για τα βιντεοπαιχνίδια δεν υπάρχει θέμα εξάρτησης ή εθισμού, αλλά αιμονή. Αποκτά κανείς μια συμπεριφορά επίμονη, δηλαδή ένα αγοράκι που επί 24 ώρες 24 ώρο παίζει με ένα παιχνίδι δεν έχει πρόβλημα εξάρτησης. Αυτό ονομάζεται αιμονή δεν είναι σωματικά ασθενείς, αυτό τουλάχιστον λένε εμπειρογνώμονες. Και τέλος, πολύ συχνά ευνηδιάζομαι και καλό θα ήταν εδώ να χρησιμοποιούσαμε ένα άλλο βιντεοπαιχνίδι για να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Το βιντεοπαιχνίδι που ονομάζεται, ναι, αυτό είναι κάτι που φαντάζομαι ότι σε έναν εικονικό κόσμο όπως αυτός του διαδικτύου μπορεί να το φανταστεί κανείς. Γίνεται. Περιμένω λοιπόν τι τροπολογίε όλων των συναδέλφων έω τι 26 Ιανουαρίου. Ελπίζω να είναι όσο επικοδομητικέ και να οδηγηθούμε σε ένα αίσιο πέρα. Ευχαριστώ. Είπατε ότι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι στις 26 Ιανουαρίου, στις 10 Φεβρουαρίου έχουμε την ψηφορία και ώρα να περάσουμε στην ε, έκθεση του κυρίου Νιούτον Ντάν. Συμφωνείτε να βάλουμε τη συζήτηση Κύριε Χάρμπορ, για τις προμήθειες πριν από το εμπορικό στάδιο για αύριο το πρωί, μπορείτε να το δεχτείτε, διότι πραγματικά δεν έχουμε χρόνο για όλα τα θέματα. Υποθέτω ότι δέχεστε την πρότασή μου. Κύριε Νιούτον Ντάν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά είναι εκπληκτικό πόσο πολλά μέλη τη Επιτροπή βρίσκονται ακόμα εδώ. Η καλύτερη είναι εδώ. Δεν βλέπω να διαφωνεί κανεί, άρα έχω δίκιο. υπέβαλα σχέδιο της νομοδότησης γραπτό όσο όχι σε όλες τις γλώσσες. Να με συγχωρείτε, κάναμε όσο πιο γρήγορα μπορούσαμε όμως. Να, ευχαριστώ, να ευχαριστήσω τη γραμματεία της Επιτροπής μας για την, ε, για την σταθερή βοήθεια που μας ε, παρήσχε στην ετοιμασία της έκθεσης αυτής. Και το μόνο που θέλω να πω, Πρόεδρε, είναι ότι οι συνάδελφοι δέχονται τις προτάσεις μας για τον Γενικό Προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ρωτήσω και τους υπόλοιπους συναδέλφους που ενδεχομένως να μην συμφωνούν εάν έχουν προτάσεις να μας κάνουν. Yes. Ferreira Next, Ο κύριος Χάσε Φερέρα. Την άποψή μας ως ομάδας την ε, εξέφρασε η κυρία Κατού και εδώ και δύο χρόνια στην Επιτροπή του Δημοσιονομικού Ελέγχου και του προπολογισμού έχουμε κάποια σχετική εμπειρία. Θα συμφωνήσουμε λοιπόν με τι προτάσει του κ. Νιούτον όμως όμω θέλουμε να καταστήσουμε σαφέ ότι ο βαθμό ανάκτηση του 55% για δημοσιονομική γραμμή των τελωνιακών δεν επαρκεί. Θέλουμε να καταλάβουμε καλύτερα. Και ίσως μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί είναι τόσο χαμηλό το ποσοστό αυτό. Αυτό που μας κάνει να αμφιβάλλουμε είναι ότι μεταβλήθηκε η στάση της Επιτροπής σε κάποια ζητήματα και το Κοινοβουλίου. Όπως με την έκθεση Μανιατίσεν και υπήρξαν αλλαγές σε πολλές γραμμές του προπολογισμού. Αυτοί οι αριθμοί δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη μόνο σε εκδικητική. Έχουμε τα στοιχεία από το 2008, έχουμε και αυτά το 2007 Άρα αυτός, αυτό το ποσοστό ανάκτησης για τα προγράμματα προστασίας των καταναλωτών δεν θα πρέπει να, ξεχωριστούν, να εξεταστούν ξεχωριστά. Ποια είναι εδώ και η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Νίτον Τάιν ήταν πολύ προσεκτικός, συνετός εδώ, αλλά θα ήθελα να ακούσω και την τελική τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά. Διότι σε κάθε περίπτωση ζητούμε για περικοπές του προπολογισμού σε πολλές θέσεις. Και δεν χρησιμοποιούμε μετά όλα τα κονδύλια ή κάποιες φορές πηγαίνουμε και πολύ μακριά. Με 45% λιγότερη χρήση του, του εγκεκριμένου προπολογισμού και ένα άλλο 33%. Εδώ δεν είναι το θέμα, το, το πρόβλημα εδώ δεν είναι το 33%, είναι χαμηλότερο το ποσοστό αυτό από προηγούμενα χρόνια. Για το ποσοστό λοιπόν το 55% τι έχετε να μας πείτε, ή εσείς κύριε Σίγητα ή η Επιτροπή. Κατά την άποψη τουλάχιστον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το χρόνο σε αυτή τη συνάντηση να μα το διασαφηνίσει, τόσο καλύτερα. Νομίζω ότι τα πράγματα μπορεί να επιδεινωθούν με αυτά που βλέπω εδώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρούλα έχει μια σύντομη παρατήρηση. Μία πρόταση ήθελα να πω. Ήθελα να παρακαλέσω τον ε, κύριο Νιούτονταν να επιστήσει την προσοχή της κυρίας Φουρτού στο γεγονός ότι ε, δεν έχει εξαντληθεί η γραμμή 2.7 του προϋπολογισμού. Ε, είμαι λοιπόν της άποψης ότι όπως ο προλαλής σα, ότι θα πρέπει η Κομισιόν να μας το εξηγήσει αυτό. παρουσία όμως της κυρίας Φουρτού διότι ήταν υπεύθυνη για την έκθεση και είχαμε πάντα την επιτύπωση ότι το ποσό αυτό είναι υπερβολικά ε, χαμηλό και όχι υπερβολικά ψηλό. Ευχαριστώ. Θέλει η Κομισιόν να σχολιάσει ε, το θέμα αυτό των ε, τελωνίων. Εντάξει. Ευχαριστώ. Μπορώ μόνο να μιλήσω για τα τελωνία. Okay. Μπορώ να μιλήσω μόνο για τις προβλέψεις ε, για ε, το 1404. Ε, οι πιστώσεις υποχρεώσεων ήταν δύσκολο να προβλεφθούν ακριβώς για μια δεδομένη χρονιά. Η πλειοψηφία των συμβάσεων δεσμεύσεων πληρωμών ε, δηλαδή έχουν να κάνουν με πληροφορική και το μεγαλύτερο μέρος ε, έχει να κάνει με ε, υπηρεσίες που παρέχονται κατόπιν αίτησης και είναι πολύ δύσκολο να προβρεθούν οι δημοσιονομικές ανάγκες. Αυτό εξηγεί γιατί φέτος είχαμε χαμηλότερη εκτέλεση των πιστώσεων πληρωμών για τα τελωνία το ποσοστό εκτέλεσης είναι πολύ ψηλότερο το 2008. 97% είναι των ε, πιστώσεων πληρωμών λόγω πιο αυστηρής ε, αξιολόγησης των ε, αναγκών Αυτό ε, έχει συμβάλει στην ε, μείωση της διαφοράς ε, ανάμεσα στις πιστώσεις που προβλέπονται και στις πιστώσεις που τελικά χρησιμοποιούνται. Κύριε Νιούτον Ντάν, θέλετε να σχολιάσετε. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομη, πολύ καλή συζήτηση όμως. Θα ήθελα να πω στην κυρία Ρούλε ότι έχει δίκιο. Πράγματι δεν εξαντλήθηκε το ποσό. Μιλάμε όμως για το 2007. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για την εξάντληση των πόρων το 2007. Πάει αυτό. Απλά λέμε ότι δεν θέλουμε να γίνει αυτό στο μέλλον. Ε, χαιρόμαστε λοιπόν που η Κομισιόν λέει ότι το 2008 που επίσης πέρασε ε, δεν έχει ολοκληρωθεί όμως ε, ο έλεγχος για τη χρονιά αυτή. Ήταν πολύ καλύτερο έτος όσον αφορά το θέμα αυτό. Σημειώσαμε λοιπόν ότι η χρήση των πόρων ήταν πολύ χαμηλή το 2007 και ελπίζουμε κάτι τέτοιο να μην επαναληφθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 30 Ιανουαρίου. Εξέταση των τροπολογιών Λοιπόν, ε, στην ΙΜΚΟ θα γίνει στις 10 Φεβρουαρίου και ε, ε, στην Επιτροπή 16 Μαρτίου και κατά την 17η εβδομάδα του έτους ψηφοφορία. Συμφωνήσαμε ότι δεν θα κάνουμε σήμερα την έκθεση Χάρπουρ. Προχωρούμε λοιπόν στην παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές. Κυρία Μπερναντέτ Βερνιό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχά μια και δεν έχω δει ακόμη όλου τους συναδέλφους, καλή χρονιά σε όλε και όλου. Ελπίζω να συνεχίσουμε μαζί την επικοδομητική μα εργασία και μετά τι εκλογέ εφόσον έχουμε ήδη γνωρίσει τόσο καλά. Το ζήτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τα απόδειξη είναι ότι έλαβα πολλέ τροπολογίε. Πράγμα που δείχνει πόσο ενδιαφέρονται οι βουλευτές για την προστασία των καταναλωτών. Και με αφορμή ένα κείμενο της Επιτροπής που ούτως ή άλλως έχει πολλές θετικές πτυχές. Ιδίως ό,τι αφορά την πληροφόρηση των καταναλωτών. Ε, η πρόταση αυτή επικεντρώνεται σε δύο βασικούς άξονες. τι γενικές απαιτήσεις για την ετικετοθεσία των προφήμων ε, και από την άλλη την αντικατοθωσία σε άλλα γεωργικά προϊόντα. Ένα συνολικό κείμενο με τις απαιτήσει όλου του συστήματος. Και αυτό γιατί η παχυσαρκία γίνεται ένα φαινόμενο ανησυχητικό για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Ενώ οι Ευρωπαίοι ανησυχούν όλο και περισσότερο για την ποιότητα ορισμένων προϊόντων. Είναι λοιπόν καθοριστική σημασία οι καταναλωτέ να λάβουν όλε τι αναγκαίε πληροφορίε για την διατήρηση, τη διαφύλαξη τη υγεία του. Νομίζω ότι το γεγονό ότι οι τροπολογίε είναι πάνω από 200 δείχνει πόσο σημασία δείχνουν οι βουλευτέ στο θέμα αυτό. Γι' αυτό και ζήτησα και την αναβολή τη ψηφοφορία. Είχαμε τι διακοπέ, άλλαξε χρονιά, δεν είχαμε χρόνο να ειδωθούμε και να συζητήσουμε. Σημαντικό νομίζω λοιπόν είναι, θα είναι να τα ξαναπούμε όλα αυτά. Ακόμη και σε μια μήνυ συνεδρίαση μεταξύ συγητών και σκεδών για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Έλαβα, πήρα τι τροπολογίε μια μία-μία και είδα ότι με μερικούς από εσά ενδεχομένως να μπορούσα να συζητήσω και με τους κοιόδης εισηγητές, κύριε Ιτονάρης. Χάρης, ε, μπορούμε να οδηγηθούμε σε συμβαστικές λύσεις ενδιαφέρουσες και για πολλές τροπολογίες πιστεύω παρόλα αυτά ότι θα είναι πολύ πιο ενδιαφέρον να ψηφίσουμε εφόσον έχουμε καταλήξει σε ενδιαφέρουσες συμβαστικές προτάσεις ακόμη και αν υπάρχουν κάποιες αποκλήσεις μεταξύ των απόψεών μας. Πάντω, σε κάθε περίπτωση θέλω να διευκρινίσω ότι δεν θέλουμε να διαστρεβλώσουμε κάποιε από τι θετικέ πτυχέ του κειμένου τη Επιτροπή. Θα πρέπει να μπορούμε να ανταλλάξουμε και με την Επιτροπή Άγκρη, που και εκείνη ανέβαλε την ψηφοφορία τη έκθεση αυτή, γιατί και εκείνη έχει χρόνο να το συζητήσει, χρειάζεται χρόνο να το συζητήσει περιττέρω. Παρομοίω δε και η Επιτροπή ΕΝΒΗ, οπότε δεδομένων όλων αυτών των στοιχείων, σημαντικό είναι να έχουμε χρόνο στη διάθεσή μα. Παρ' όλα αυτά μου έκανε έκπληξη που εντό τη ίδια ομάδα, λυπάμαι που σα το λέω, γιατί με τον κύριο Ήτον Χάρι μπορεί να καταλήξω σε πολλέ συμβαστικέ λύσει, αλλά μου έκανε εντύπωση μέσα στην ίδια ομάδα υπήρξαν πολλέ τροπολογίε από άλλε πηγέ τη ίδια ομάδα που δεν ακολουθούσαν την ίδια κατεύθυνση. Ε, δεν μιλάω για το ίδιο άτομο βέβαια, ήταν άλλοι άνθρωποι. Και χωρί ε, αναγκαίως να ακολουθείται η ίδια προοπτική για την προστασία των καταναλωτών από την άποψη τη πληροφόρηση, τη υγεία και τη ασφάλεια. Ο κανονισμό αυτό θα έχει σοβαρέ συνέπειε και για του παραγωγού. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να αναζητήσουμε συμβιβαστικές λύσει για την απαιτούμενη ισορροπία προκειμένου να υλοποιηθεί ο κανονισμό αυτό στι διατάξει του και στι εξαιρέσει του σε ό,τι αφορά τι εξαιρέσει για τα αλκοολούχα ποτά. Ήταν πολλέ οι ομάδε που πρότειναν σχεδόν πανομοιότυπε τροπολογίε. Νομίζω εδώ ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβαστικέ λύσει, ιδίω αυτέ οι τροπολογίε του κυρίου Ιτων Χάρη, του κυρίου Μπούσκ, του κυρίου του Μπον, τη κυρία Φουρτού, να καταλήξουμε σε ένα συντελεστή δηλαδή περιεκτικότητα σε αλκοόλ και μια συγκεκριμένη προθεσμία. Εγώ θα έλεγα μια προθεσμία τριετία. Κάποιοι λένε πενταετία. Θα δούμε, θα τα συζητήσουμε. Ε, ε, να είναι πιο ελαστικά τα μέτρα για τα προϊόντα αυτά θέλουμε δηλαδή. Και κυρίω για όλα τα μην ποτά μηδενό ε, ξερουμένου για τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα ή τι χαρακτήρα θα έχει η ετικέτα που θα χρησιμοποιείται στο σύστημα ετικετοθεσία. Εγώ είμαι ανοιχτή να το συζητήσω. Υπάρχουν πολλέ προτάσει, αλλά πραγματικά είμαι πολύ ανοιχτό μυαλί. Εδώ δεν έχω καμία παροπίδα στο, στη σκέψη μου και είμαι στη διάθεσή σα για να βρούμε λύσει όσο δυνατόν πιο ισόρροπε και για να ε, προστατεύσουμε τους παραγωγούς, τους κατασκευαστές και τους καταναλωτές που πρέπει να είναι πλήρως ενημερωμένοι, αλλά να λαμβάνουμε υπόψη και τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις για την αντικοτοθεσία. Δεν είναι απλό. Σε ό,τι αφορά την αντικοτοθεσία με διατροφικά στοιχεία, προτείνω ένα σύστημα αναγραφή στην εξωτερική πλευρά του πακέτου. Μια καλή συμβαστική πρόταση. Αυτό το τρίχρωμο σήμα που. Την τρίχρωμη όπως όπω ονομάζεται, που θα δίνει ποσοστά για την ημερήσια πρόσληψη και ούτω Ε, είμαι έτοιμη να συζητήσω τον τρόπο που θα υλοποιηθεί αυτό ακριβώ. Ακόμα και τον αριθμό των χαρακτήρων που θα αναγράφονται στην προστινή πλευρά του πακέτου, πώς ακριβώς θα είναι η αναλογία, πώς θα είναι υπολογισμένες ποσότητες σε αναλογίες ή σε γραμμάρι λόγου χάρη, καθώς και την αναφορά της χώρας προέλευσης ή της χώρας καταγωγής. Αυτά μπορεί να διαφέρουν και μπορεί να είναι και περίπλοκη η παρακολούθηση μιας τέτοιας έννοιας. Ακόμα και η διατύπωση και η αναγραφή στην ετικέτα μπορεί να είναι περίπλοκη. Νομίζω το σχέδιο αυτού του κανονισμού, του ε, αποτελεί δήμα προόδου και μέχρι την ψηφοφορία μας μπορούμε να βελτιώσουμε πολύ την πρόταση. Ιδίω για να διαφυλάξουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών και έχοντας υπόψη και τις παρατηρήσεις των παραγωγών. Νομίζω ότι Πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά όλε τι τροπολογίε όπω τη κυρία Ρόιτοβα που ίσω να έχει φύγει, για τα αλλαργιογόνα, για τη γλουτόνη, γλουτίνη, τη κυρία Σαντεμόζε, η οποία ε, εγείρει το πρόβλημα των οξυδίων. Εδώ νομίζω ότι φτάνουμε σε ένα σημαντικό ζήτημα διότι πριν από μισή ώρα περίπου έλαβα αυτές τις τροπολογίε, που ήταν και στα αγγλικά οπότε δεν μπορούσα να τις μελετήσω και μάλιστα μια μελέτη τη Επιτροπή που είχε παραγγείλει η Επιτροπή για την ε, έκθεση αυτή τη μελέτη περί λιπαρών οξυδίων. Αποδεικνύεται ότι από τρική πλευράς είναι πολύ επικίνδυνη για την υγεία αυτά, κυρίω για καρδιογειακά επεισόδια. Νομίζω λοιπόν ότι καλό είναι να δούμε από κοινού ορισμένε από τι τροπολογίε αυτέ που είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσε και να καταλήξουμε και σε συμβαστικέ προτάσει. Αντιθέτω, το να περιορίσουμε την ε, πρόταση αυτή σε ελάχιστα, ε, στις ελάχιστες απαιτήσει, περιορίζοντα ένα μεγάλο μέρο του κειμένου και εξυπηρετώντα τα συμφέροντα των μεγάλων βιομηχανών τροφίμων που έχουν προβάλει τα συμφέροντά του μέσω κάποιων ενώσεων και έχουν ε, προκαλέσει την διάδοση πολλών ε, νόσων που σχετίζονται με τα θέματα αυτά. Όλο αυτό νομίζω θα είναι καταστροφικό για την υγεία των πολιτών μα. Πρέπει να το προσέξουμε λοιπόν. Γιατί είναι επιζήμιο και για την δική μα την αξιοπιστία. Σα ευχαριστώ όλου, όλου όσοι συμμετείχατε και υποβάλλατε και τι τροπολογίε σα, είτε ακολουθείτε τη δική μου τη γραμμή είτε όχι, για να βελτιώσουμε το κείμενο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Πρώτος είναι ο κύριος Κίτων Χάρης. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια που επέτρεψε την αναβολή της ψηφοφορίας γιατί νομίζω ότι απέχω, απέχουμε αρκετά από τις, ε, ε τους συμβιβασμούς ε, για τους οποίους ε, μιλάει. Δεν έχουμε βρεθεί, δεν έχουμε συναντηθεί ακόμα, μόνο με email έχουμε συνεννοηθεί. Θα ήταν λοιπόν χρήσιμο να αναβάλουμε την ψηφοφορία. Συμφωνώ μαζί σας, νομίζω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβασμό σε αρκετούς τομείς του θέματος αυτού. μου δίνετε την αίσθηση ότι σας ενδιαφέρουν κάποιες από τις ε, τροπολογίες ε, του κυρίου ε, Κάρους και κάποιες είναι αρκετά ενδιαφέρουσες και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπο να τις βάλουμε στο κείμενο. Πρέπει να παραδεχτώ ότι δεν καταλαβαίνω την χημεία πίσω από όλα όσα κάνουμε εδώ πέρα, ε, τις επιστημονικές εξηγήσεις. Ε, καταβάλω κάθε προσπάθεια να καταλάβω. Ε, χαίρομαι λοιπόν όταν άλλοι με συμβουλεύουν. Είναι χρήσιμο το να είναι κανείς σε ε, μεγάλη πολιτική ομάδα ε, για να έχουμε για παράδειγμα τον κύριο Κάρες που μας δίνει πληροφορίες αλλά απ' την άλλη ε, περιμένω εναγωνίες τις μέρες που θα είμαστε μικρότερη πολιτική ομάδα για να μην δημιουργούμε τόσα προβλήματα για όλους τους άλλους. Το θέμα είναι σε τι θα συμφωνήσουμε να συμφωνήσουμε. Καταρχήν έχουμε τα σημαντικά θέματα, έχουμε το GDA, το φανάρι όπως λέμε, τις συνιστόμενες ημερήσιες δόσεις ε, νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι αυτό είναι αυτό που καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε κατόπιν αν αυτό θα γίνει αναμερίδα ή ανά 100 γραμμάρια. Κάποιες ε, εταιρείε τροφίμων ε, αναγράφουν και τα δύο. Αυτά εξαρτώνται από το μέγεθος της συσκευασία. Θα είναι λοιπόν ενδιαφέρουσα η συζήτηση για το θέμα αυτό. Κατόπιν, τι θα μπαίνει στο μπροστινό μέρος του πακέτου ή στο βασικό πεδίο ε, ε, που βλέπει κανείς ε, και τι θα μπει σε άλλα μέρη της συσκευασίας. Διότι υπάρχει κίνδυνο να απαιτούμε να μπαίνουν τόσα πράγματα στο προστινό μέρο του πακέτου που να μην υπάρχει πίσω μέρο του πακέτου, να μην μένει χώρο για τίποτα άλλο. Ε, υπάρχει και το θέμα αν θα τα μετράμε σε θερμίδε, σε κιλοτζάουλ ε, κλπ. Είμαι ιδιαίτερα πεπισμένο ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε λογικό συμβιβασμό για το μέγεθο των γραμμάτων. Δεν πιστεύω ότι το συζητάμε αυτό τόσο καιρό και ότι ακόμα δεν έχουμε καταλήξει σε κάποια λύση. Είμαι όμως πεπισμένο ότι δεν είναι πολιτικό θέμα. Ε, το θέμα είναι να κάνουμε μια λογική πρόταση ώστε οι καταναλωτές να καταλαβαίνουν το μήνυμα, να είναι ευανάγνωστο, να, ε, μην μπορεί να σβηστεί εύκολα. Ε, θα πρέπει να είναι λογική η πρόταση τελικά και, ξέρω ότι όλοι συμφωνούμε ότι η πρόταση της Κομισιόν ε, δεν ήταν ε, απολύτως καλή, ολοκληρωμένη. Ε, υπάρχει σημαντικό λόμπι, η Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών. Έχω μιλήσει και με ενώσει ε, καταναλωτών ε, στα διάφορα κράτη-μέλη και αναρωτιέμαι... συγγνώμη για το κινητό, η μαμά μου με παίρνει. Ναι, με παίρνει να δει τι, τι τρώω. Και προφανώς πρέπει να κάνει πιο αυστηρούς ελέγχους. θα καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό που ε, θα μπορούν να δεχτούν ε, όλοι για το μέγεθος των γραμμάτων ε, και την αναγνωσιμότητα Ως προς τα, τις θρεπτικές ουσίες, ε, τα εθνικά σχέδια μπορούμε να εργαστούν πάνω σε αυτό. Όλοι νομίζω συμφωνούν ότι το κοινοβούλιο μας ε, θα πρέπει να έχει λέγει στις ε, τροποποίησεις που θα γίνουν στο θέμα αυτό με την Κομισιόν στο μέλλον. Είμαι πεπισμένος ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε, νομίζω όμως ότι έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Ε, ε, εγώ και η συγγήτρια μένουμε στο ίδιο ξενοδοχείο στο Στρασβούργο. Ίσως να μπορούμε λοιπόν να συναντηθούμε εκεί για ένα ποτάκι. Μια και μιλάμε για διατροφή, νομίζω ο Winston Churchill είχε πει ότι κάποιες φορές κατάπινε τα λόγια του. Οπότε αυτό ήταν τελικά μια ισόρροπη διατροφή. Ισορροπημένη μάλλον. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Θα είμαι σύντομος να συγχαρώ και εγώ την εισηγητρία γιατί νομίζω ότι πηγαίνουμε σε μια καλή κατεύθυνση. Για τα ετικέτε, ε, συμφωνώ με τα έξι θρεπτικά συστατικά που πρέπει να αναγράφονται στον προστινό τη συσκευασία, όπω έχει προτείνει και η Επιτροπή. Και για το ευανάγνωστο των πληροφοριών που θα παρέχονται, νομίζω ότι η Επιτροπή, αφού συζήτησε με όλε τι ομάδε ενδιαφέροντο, θα πρέπει να προβλέψει αυστηρού κανόνε, οι οποίοι θα πρέπει να ε, διατεθούν πριν από τη θέση ισχύ τη νομοθεσία. Γι' αυτό έχω προτείνει μια σχετική τροπολογία και ήδη θέλω να δούμε πώς μπορούμε να ε, επιλύσουμε αυτή την κρίση του δανάγνωστο που συμφωνομαστεί. Επίσης, για τη μεταβατική περίοδο ήδη συζητήσαμε γι' αυτό και νομίζω αν θέλουμε απλουστευμένη, συνεκτική και εύκολο να εφαρμοστεί νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρέπει να επιτρέψουμε εθνικές διατάξεις. Νομίζω για τα αλκοολούχα ποτά θα αποσύρω τη σχετική μου τροπολογία, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και σε αυτή την πρώτη φάση ήθελα να προτείνω πενταετία. Πενταετία για την έγκριση τη πρόταση από την Επιτροπή, αλλά μπορώ να στηρίξω και αυτό που ζητάει η συγγετρία την τριετία. Για την χώρα καταγωγή, ή για τον τόπο προέλευση, νομίζω ότι καλό αυτό είναι να διευκρινίζεται. Και όπου δεν διευκρινίζεται αυτό, μπορεί να παραπληνηθεί ο καταναλωτή. Για τι τροπολογίε του τη εισηγήτρια, νομίζω ότι τα χαρακτηριστικά συστατικά είναι μάλλον ακατάλληλο να αναγράφονται. Η χώρα προέλευση των πρώτων υλών δεν έχει θα πρέπει να αναγράφονται μόνο στην περίπτωση που εκπροσωπούν το 50% της συνολικής, της, του τελικού προϊόντος. Και όχι σε αντίθετη περίπτωση, αλλιώ θα είναι πολύ περίπλοκο το σύστημα. Ευχαριστώ. Mr. is the next one. Ο κύριος Σουάμπ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πολύ σύντομα. Ε, ο κύριος ε, ε, δυστυχώς δεν μπορούσε να είναι παρόν. Μου ζήτησε ε, Ε, ε, να απαντήσω όχι μόνο στον κύριο Χίτον Χάρης ε, αλλά και στην κυρία Βερνιό που έχει εκπονήσει την έκθεση αυτή ως ε, προς ε, την παρατήρηση του κυρίου Κάρασε για το μέγεθος ε, των γραμμάτων. Πρέπει να είναι ευανάγνωστο ο σοπίνακας αλλά δεν εξαρτάται αυτό αποκλειστικά από το μέγεθος των γραμμάτων. Ως προς τα προγράμματα, τα schemes, αφήνεται εδώ ανοιχτό το παράθυρο για εθνικά στοιχεία, Χρειάζεται ευρωπαϊκή λύση και εδώ υπάρχει συμφωνία ότι ε, άλλωστε ο συνάδελφος ε, Χίτον Χάρης ε, αναφέρθηκε στο θέμα αυτό. Επίσης, ο κύριος Κάρας βρίσκει προβληματική την υποχρέωση να αναφέρεται η προέλευση όλων των συστατικών, διότι δεν είναι βέβαιο ότι προέρχονται όλα αυτά τα ε, συστατικά από την ίδια χώρα, από την Αυστρία δηλαδή. Ε, πιστεύω όμως ότι έτσι με τα στοιχεία αυτά που θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε έναν καλό σύμβασμο. Ευχαριστώ κυρία Σάντεμόζε. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που βλέπω ότι συμφωνώ με τον συνάδελφο Κρισχή τον Χάρης. Αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά. Ε, πράγματι πάντως ε, ε, ανακαλώ, λέει ο κύριος Χίτον Χάρης. Ε, ε, θα, θα μας πάρει λίγο χρόνο να συμφωνήσουμε για, πάνω στις τροπολογίες. Θα πρέπει να κάνουμε δουλειά. Μία παρατήρηση έχω Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό ε, όταν αποφασίσουμε αν θα επιλέξουμε τη μία ή την άλλη λύση, αν θα πρέπει να βρίσκονται στο πρωθυνό μέρο τη συσκευαστία ή στο πίσω μέρο τη συσκευαστία ε, οι πληροφορίε. Ε, τα περισσότερα από αυτά είναι θέμα γούστου στο κάτω-κάτω. Τι πιστεύουμε ότι είναι καλύτερο για του καταναλωτέ. Κάποιε πληροφορίε όμω είναι σημαντικέ για την υγεία των ανθρώπων, γι' αυτό είναι σημαντικό να προσέξουμε το θέμα. Θα πρέπει όμω να φροντίσουμε οι καταναλωτέ να μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίε σχετικά με τι πρωτενε ε, στα τρόφιμα, διότι υπάρχουν άνθρωποι ε, που ε, πάσχουν από ασθένεια που καθιστά σημαντικό να λαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με το ποσοστό πρωτεϊνών στα τρόφιμα. Τα υπόλοιπα είναι βέβαια θέμα γούστου, θέμα γνώμη. Τι πιστεύει κανεί ότι είναι πιο αποτελεσματικό για του καταναλωτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τελευταία παρέμβαση είναι της Κομισιόν. Μια παρατήρηση θέλω να κάνω όμως. Ε, όταν ε, άρχισα να ασχολούμαι με το θέμα των θρεπτικών πληροφοριών, ε, δεν μπορούσα να τις, όταν έφτασα στην ηλικία να ενδιαφέρομαι ε, για τις πληροφορίες για τις θρεπτικές ουσίες, δεν μπορούσα πια να τις διαβάσω. Ήταν πολύ μικρή η γραμματοσυρά. η Κομισιόν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή το διάλογο που είχατε στην Επιτροπή, μελετήσαμε και τις διάφορες τροπολογίες και είχαμε και την ευκαιρία να τοποθετηθούμε κατά την παρουσίαση της έκθεσης της κυρίας Βερνό και επαναλάβαμε την ικανοποίησή μας με το σχέδιο αυτό γνωμοδότησης, το οποίο βρήκαμε ιδιαίτερα επικοδομητικό. Δεν διαφωνούμε με την άποψη της κυρίας Βερνιό για ορισμένε από τις τροπολογίες που πιστεύουμε ότι αντίκεινται στα συμφέροντα των καταναλωτών και σε γενικές γραμμές η Επιτροπή είναι και αυτή αρκετά ανοιχτή, μπορεί να εξετάσει τροπολογίες που στοχεύουν να καλύψουν ακόμη περισσότερο και με πιο αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα της βιομηχανίας, έχοντας πάντα κατά νου ότι η πρόθεση της πρότασης αυτής είναι κατά πρώτον να βελτιώσει την πληροφόρηση των καταναλωτών. Αντιθέτως, οι τροπολογίες που αποδυναμώνουν ή ισοπεδώνουν τελείως το σκοπό αυτό που επιδιώκει η Επιτροπή και οδηγούν στη διατήρηση του status quo, ε, δηλαδή σε καμία περίπτωση να μην προβλέπεται καμία αλλαγή, εκεί βεβαίως έχουμε σοβαρούς ενδιασμούς και επιφυλάξει. Δεν θα μπορούσαμε να το δεχτούμε. Σας συγχαίρουμε για την αποφασή σας να αναβάλλετε την ψηφοφορία, εάν αυτό μπορεί να μας οδηγήσει σε ακόμη καλύτερες συμβαστικές λύσεις και να διευκολυνθεί η πρόοδος του συγκεκριμένου θέματος και παραμένουμε στη διάθεσή σας. Ιδίως γερισμένα θέματα. Απλώς να σταθώ στο θέμα των αρκολούχων ποτών βλέπουμε ότι εδώ υπάρχει τάση όλα τα αλκοολούχα ποτά να συμπεριληφθούν στην ίδια ομάδα. Εξαίρεση δηλαδή για όλα αυτά τα προϊόντα, συλλήβδιν, ακόμα και για τα αλκοπόψ που εμείς η Επιτροπή θεωρούμε πολύ σημαντικό να διακρίνονται από άλλα προϊόντα όπως η ίνη, η άλλα είναι ο πνευματόδη με ιδιαίτερες ιδιότητες. Εδώ μιλάμε για αναψυκτικά που αναμειγνύονται με ποτά κλασικά, συνηθισμένα, χωρίς καθόλου καμία περιεκτικότητα σε αλκοόλ και που καταναλώνει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, του νεαρού πληθυσμού ιδίω. Σε ό,τι αφορά τα μη προσυσκευασμένα προϊόντα, για μας είναι πολύ σημαντικό οι πληροφορίες και οι υποχρεώσεις πληροφόρησης για τα λεγόμενα να διατηρηθούν, να διατηρηθούν στο τελικό κείμενο. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες εναλλακτικέ οδοί για να αποφύγουμε το περιττό άχθος για τους ε, εμπορευόμενους. Αυτές τις εναλλακτικέ λοιπόν ευχαριστώ να τις κρατάσουμε μαζί σας. Και επιπλέον για τη χώρα καταγωγής να πω ότι είδαμε τροπολογίες που θα οδηγούσαν στην πλήρη κατάργηση από την πρόταση της Επιτροπής αυτής της έννοιας. Εκεί προφανώς δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Έχουμε επιφυλάξεις και όπως προείπαμε να κρατάσουμε ευχαρίστως τρόπους να κάνουμε πιο ελαστική την υποχρέωση αυτή για τη βιομηχανία, αλλά η πλήρης κατάργηση μάλλον θα έπλητε το σκέλος της πληροφόρησης των καταναλωτών. Αυτά ήταν τα σχολεία μας. Ευχαριστώ. Now we finally can... Και τώρα νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Κυρία Βερνιό. Κοιτάξτε. Νομίζω ότι ήταν απαραίτητη αυτή η χρονική καθυστέρηση. Να ευχαριστήσω τον κύριο Σφάμπ. Κοιτάξτε, δεν τα έχω πετάξει κιόλα. Το κύριο Κάρα έχω διατηρήσει ένα μεγάλο μέρο των τροπολογιών. Άρα θα πρέπει να τα συζητήσουμε. Όσα είπε ο κύριο Τον Χάρη και Αυτά είναι πράγματα που θα τα ξανασυζητήσουμε. Για τα αλκοόλουχα τα πράγματα. αυτό που ανέφερε η Επιτροπή είναι κάτι που και αυτό μπορούμε να το διαπραγματευτούμε. Νομίζω η ουσία είναι ότι διαφέρει η πρόταση των ΜΕΝ και των ΔΕ, δηλαδή τι θα μπει ω προτεραιότητα, τι θα μπει στο προστινόμενο τη συσκευασία, τι στο πίσω, τι θα γίνει με τα αλλεργιογόνα, με τα συσκευασμένα μη προσυσκευασμένα προϊόντα, ναι, συμφωνώ, εδώ πρέπει να παραμείνουν οι πληροφορίες και να διατίθενται στον καταναλωτή, ίσως όχι αναγκαστικά να επικολώνται πάντοτε οι πληροφορίες, αλλά εκεί που είναι αναγκαίο, ναι. Ε, και σημαντικό είναι να βρούμε απλές λύσεις, διότι πλήρης εναρμόνιση όπως ζητήθηκε για τα δικαιολογητικά 27 χωρών. Δεν έχω τέτοιες φιλοδοξίες, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο μαγικά. Αλλά πρέπει να ακολουθούμε μια κοινή τάση, να, να στείλουμε λογότυπα, καθαρά σήματα, χρώματα, πράγματα τα οποία μπορεί κανείς εύκολα και να τα, να τα μάθει και να τα χρησιμοποιήσει όπως θα γινόταν με έναν απλό κωδικό, μια γραμμή κωδικού αλλά φανταστείτε αν δεν υπάρχει τίποτα άλλο πάνω στο προϊόν. Εάν κάποιο να περάσει στο μηχάνημα του σούπερ μάρκετ, να περάσει το code bar για να διαβάσει σε μία οθόνη τι πληροφορίε για το προϊόν. Μια κυρία 65 χρονών που δεν μπορεί καλά-καλά να περπατήσει, πώ θα φτάσει μέσα στο του σούπερ μάρκετ να διαβάσει το κωδικό αυτό και να λάβει τι απαραίτητε πληροφορίε. Αυτά είναι απαράδεκτα εννοείται. Τώρα όμω, όσε τροπολογίε ε, μιλούν για τον τομέα των τροφίμων που των που θέλουν να είναι και ενδιαφερόμενο μέρο και κριτή στο τι πληροφορίε θα διατίθενται στον καταναλωτή, ε, νομίζω ότι αυτό είναι ανέφικτο επίση. Διότι στόχο είναι προστασία του καταναλωτή. Δεν μπορεί ο ίδιο που διαθέτει τα προϊόντα να αποφασίζει τι θα διαθέσει στον καταναλωτή ω πληροφορία. Ο Ευρωπαίο πολίτη πρέπει επίση να αναλάβει τι ευθύνε του. Είναι και αυτό πολύ σημαντικό εδώ πέρα. Ευχαριστούμε κυρία Βερνιό. Θα συνεχίσουμε αύριο το πρωί με πρώτη ομιλήτρια την κυρία Βασιλείου. Παρακαλώ να είστε εδώ.